Καλημέρα σα, συνάδελφοι λέει ο Πρόεδρο Κυρίσω την έναρξη της συνεδριάσεως. Στην πρώτη εβδόμου η Συμβουλευτική Επιτροπή για την Διοντολογία πρότεινε επιβολή κυρώσεων στον Γιάννη Ζαχράντιλ για έλλειψη σεβασμού προς τα όσα επιβάλλει και επιτάσσει το άρθρο 3 άρθρο 4 παράγραφος 2 του κώδικα διοντολογίας. Επρόκειτο για σύγκρουση συμφερόντων. Επίπληξη είναι η κύρωση. 7 Ιουλίου κοινοποιήθηκε στον ενδιαφερόμενο. Σύμφωνα με το άρθρο 176 έχει δύο εβδομάδες από την κοινοποίηση της κύρωσης να προσφύγει στο Πρόεδριο. Πριν να αρχίσουμε τις συζητήσεις, θα πρέπει να σας ανακοινώσω τα αποτελέσματα της δεύτερης ψηφοφορίας και της πρώτης ψηφοφορίας για σήμερα. Ψηφοφορίας Τετάρτης. Όσον αφορά τις ε, διατάξεις για την ε, απόσπαση των οδηγών. Έχουμε το, την τροπολογία 5 που απορρίπτεται. 6 ε, ε, και 7 απορρίπτονται. 8, 10 και 11 απορρίπτονται. 9 και 30 απορρίπτονται. Η τροπολογία 31 απορρίπτεται. Τροπολογίες 12 και 32. 13 και 3 και 33 απορρίπτονται. 14 και 34 απορρίπτονται. 35 απορρίπτεται. 15 επίσης. 36 απορρίπτεται 16 απορρίπτεται 37 απορρίπτεται 17 απορρίπτεται 18 και 38 απορρίπτονται 19 και 39 απορρίπτονται 20 επίσης 21 επίσης 22 επίσης 40 απορρίπτονται και το 24 τα 2 και 25 το 26, το 3, το 4 και το 27. Όσον αφορά τώρα τα, ε, το χρόνο οδήγησης το ανώτατα όρια και τα όρια διαλυμάτων και εβδομεδίας ανάπαυσης. Έχουμε το 10, το 11, το 4, το 12 απορρίπτονται, τα 13, επίσης το 5, το 6, το 7 απορρίπτονται, 8, 14, 15, τροπολογία 16 και αυτό. Ε, επίσης ε, η τροπολογία 17, η 18 απορρίπτονται, η 19, 9, 9 δεύτερο τμήμα απορρίπτεται και η τροπολογία 20. Όσον αφορά τις ε, ρυθμίσεις για τις οδικές μεταφορές, έχουμε 7, 17, 8, 18, 9, 19 τροπολογίες απορρίπτονται. 10 και 20. Οι 11, 21, 22 απορρίπτονται. Η τροπολογία 12, η 12 δεύτερο τμήμα απορρίπτεται. Η 23, οι τροπολογίες 3 και 14 επίσης οι τροπολογίες 4 και 5 απορρίπτονται. Οι 15η, 6 και 16η επίσης απορρίπτονται. Όσον αφορά την προστασία οικονομικών συμφερόντων και καταπολέμηση της απάτης. Το 18, 14, 18, δεύτερο τμήμα επίσης εγκρίνεται 23 ε, εγκρίνεται ε, όπως και οι προηγούμενες 23, 52, 53, 57, 58 εγκρίνονται Τροπολογίε 61, 62 εγκρίνονται 63 εγκρίνεται 63 δεύτερο τμήμα εγκρίνεται 64 εγκρίνεται 65 εγκρίνεται 66 εγκρίνεται 69 εγκρίνεται 111 και αυτή η τροπολογία εγκρίνεται Όσον αφορά τώρα τη θέση του Συμβουλίου για τους κανόνες που αφορούν την απόσπαση οδηγών για οδικές μεταφορές και τη σχετική εφαρμογή της σχετικής οδηγίας όσον αφορά διαλύματα, ε, περιόδους ανάπαυσης και επίσης τους ταχογράφους όσον αφορά την ε, εφαρμογή ε, δεν εγκρίθηκε καμία τροπολογία. Σύμφωνα με το άρθρο 67 έχουμε τρία αιτήματα σε σχέση με τη θέση του Συμβουλίου, οπότε θεωρούνται εγκριθήσεις οι θέσεις αυτές. Και τώρα προχωρούμε στον πρώτο γύρο ψηφοφορίας. Πρώτα-πρώτα. Η ψηφοφορία υπαριθμών 1 θα γίνει από τις 9 και 4 μέχρι τις 10 και 30 με την ίδια διαδικασία όπως χθες. Θα γίνουν οι ψηφοφορίες ως ονομαστικές και μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα στο website της Ολομέλειας. Οι δηλώσεις, οι σχετικές θα υποβληθούν εγγράφως. Το σχετικό κείμενο μπορεί να φτάσει τις 400 λέξεις. Είπαμε 13 λίγη ψηφοφορία και στις 2 ε, και 4 θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα. Συνάδελφοι, μισό λεπτό θέλω την προσοχή σας θα προβώ σε μια ανακοίνωση διότι όπως γνωρίζετε στο Χονγκ την προηγούμενη εβδομάδα άρχισε η ισχύ του νόμου για την εθνική ασφάλεια η κατάσταση γίνεται όλο ένα και δραματικότερη κάθε μέρα έρχονται ειδήσει για φυλακίσεις, συλλήψεις και άσκηση βίας. Δεν υπάρχει η ελευθερία του συναθρίζεστε, του λόγου. Βιβλιοθήκες και σχολεία έχουν αποστερηθεί τα βιβλία τους τα οποία κατασχέθηκαν. Προβληματιζόμαστε και όλοι θαυμάζουμε την αποφασιστικότητα, το θάρρος των πολιτών του Χονγκ Κόνγκ, διότι παίζεται η προσωπική τους ελευθερία στην αγώνα που δίνουν για μια δημοκρατική και ελεύθερη και ανοιχτή κοινωνία. Αυτό που κάποτε ήταν ε, η πραγματικότητα, δηλαδή η δημοκρατία, θεμελιώδεις ελευθερίες, κράτος δικαίου, η αυτονομία, κάτι το οποίο ήταν δεδομένο στην καθημερινή ζωή, τώρα αυτό, αυτό κινδυνεύει να εκλείψει και εμείς ως βουλευτές θα πρέπει να επιδείξουμε αλληλεγγύη, να τοποθετηθούμε κατά αυτών των χτυπημάτων που δέχεται η ελευθεροτυπία από αυτόν τον αυξανόμενο αυταρχισμό. Φαντάζομαι ότι αυτά τα οποία λέω τα συμμερίζεστε και θα πρέπει επομένως να καλέσουμε τις αρμόδιες αρχές να σεβαστούν τις ε, διεθνείς δεσμεύσεις της χώρας και τις θεμελιώδεις ελευθερίες και σας ευχαριστώ. Ci fermiamo un attimo, no? Un attimo di sospensione e poi riprendiamo con... Κάνουμε ένα και εγώ θα συνεχίσουμε με την ημερησία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 Είναι το Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. είναι Good morning everybody. Καλή σας ημέρα. Ξεκινούμε με τη συζήτηση. Σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη, έχουμε συζητήσει επί των δηλώσεων του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είπα το εκπροσώπη της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας τον οποίο θέλω και θερμά να καλωσορίσω για τρία θέματα ετήσια έκθεση του 2019 για τα ανθρώπινα δικαιώματα, σταθερότητα και ασφάλεια στη Μεσόγειο και ο αρνητικό ρόλο τη Τουρκία και η κατάσταση στη Λευκορωσία. Θα ήθελα να ενημερώσω τους ευρωβουλευτές ότι στην κοινή αυτή συζήτηση δεν ε, υπάρχει δυνατότητα ε, προσέλκυσης προσοχής του Προέδρου ούτε η διαδικασία της ε, μπλε κάρτας. Παρακαλώ κύριε Μπορέλ, κύριε Αντιπρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είπατε εκπρόσωπε. Έχετε το λόγο. Αξιότιμα μέλη, μια και δεν έχουμε πολύ χρόνο να περάσουμε απευθεία στα ζητήματα που μα απασχολούν σήμερα, η έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα για το 2019, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία. Ένα σημαντικό ζήτημα είναι η συσχέτιση μεταξύ ανθρωπίνων δικαιωμάτων και περιβάλλοντος. Το Δεκέμβριο συμμετείχα στην 21η, στο 21ο Φόρουμ των Ηνωμένων Εθνών ε, με τις οργανώσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με πολλές μαρτυρίες. Ε, το 2018, 77% των ανθρώπων που δολοφονήθηκαν και που εργάζονται υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, ασχολούνταν ασχολούταν με ζητήματα περιβαλλοντικών δικαιωμάτων, προστασία των δικαιωμάτων των ηθαγενών μεταξύ άλλων, κατά της αρπαγής της γης. Θα πρέπει να ενισχύσουμε τις προσπάθειές μας λοιπόν ε, για να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα αυτό. Η έκθεση ε, υπογραμμίζει την, την σχέση μεταξύ της ψηφιακής ε, μετάλλαξης της κοινωνίας μας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας. Οι νέες τεχνολογίες δίνουν, δικαι... δίνουν δυνατότητες προώθησης της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δημιουργούν όμως και, και ασάφεια, δημιουργούν και προκλήσεις. Χρειάζεται λοιπόν μια συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να αντιμετωπίσουμε τις ηθικές πτυχές της ψηφιακής νοημοσύνης της τεχνητής νοημοσύνης. Υπάρχει η δήλωση του Πεκίνου για την ισότητα μεταξύ των δύο φύλων. Δυστυχώ, ε, δυστυχώς, με βάση τα στατιστικά των ΟΕΕ, Εθνών, ένα τρίτο των γυναικών ανά τον κόσμο εξακολουθούν να πλήττονται από βία, κάποια μορφή βία στη ζωή τους. Παρά το γεγονός ότι βασιζόμαστε στις γυναίκες ε, για να μπορέσουμε να έχουμε όλο αυτό το εργατικό δυναμικό, το τόσο σημαντικό, νοσοκόμες κτλ. Ε, είναι αυτές που υποφέρουν περισσότερο από την πανδημία. Υπάρχουν όμως και καλά νέα. Υπάρχει πρόοδος σε επίπεδο ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δημοκρατίας Ε, να πούμε παραδείγματο χάρη ότι υπάρχει η απόφαση ε, τη κατάργηση τη θανατική ποινή στο Τσάντ. Η απόφαση τη Χέρα, της Χέρα Λεόνε να πάυσει την ε, απαγόρευση για τα κορίτσια να πηγαίνουν στο σχολείο. Στην Σρι έχουμε μια πολύ σημαντική μείωση της εργασίας των παιδιών. Λιγότερο από... Ε, περισσότερο μάλλον από 600.000 παιδιά δεν εργάζονται πια σε σχέση με πριν από κάποια χρόνια, σε Σρι Λάνκα, στην Γκάμπια. Ε, στις χώρες αυτές είχαμε, δημοκρατικές, είχαμε δημοκρατική πρόοδο και βεβαίως ε, η αντίσταση κατά της δικτατορίας ε, επίσης ε, αυξάνεται ανά τον κόσμο. Θα μπορούσα να πω περισσότερα για αυτή την έκθεση. Θα περάσω όμως τώρα στο δεύτερο ζήτημα που έχετε θέσει σταθερότητα και ασφάλεια στη Μεσόγειο και αρνητικός ρόλος της Τουρκίας. Αυτό είναι ο τίτλος σας. Στο δεύτερο θέμα της ημέρας διάταξης. Μόλις επέστρεψα μετά από εντατικές συζητήσεις με την Τουρκία και τη Μάλτα επισκέφθηκα την Ελλάδα και την Κύπρο την περασμένη εβδομάδα ε, για να επιδείξω την ελεγγύη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι σαφές ότι η σταθερότητα και η ασφάλεια στη Μεσόγειο απαιτούν μια συλλογική δέσμευση. Πολλά πολιετή σειράξει στην Συρία, στη Λιβύη έχουν πολύ μεγάλο αντίκτυπο στην περιοχή και επηρεάζει αυτό άμεσα ε, πλήττει τα συμφέροντά μας, την ασφάλειά μας σε ό,τι αφορά τον έλεγχο της μετανάστευσης, της τρομοκρατίας, ε, ε, την πολιτική σταθερότητα, από το Σαέλ μέχρι τη Μέση Ανατολική Τουρκία επηρεάζεται από αυτήν την ε, κατάσταση. Είναι ενεργή μάλιστα και στις Ιράξεις και στη Συρία και στη Λιβύη. Είναι από τους βασικούς παράγοντες και στις δύο αυτές εμπόλεμες καταστάσεις. Έχουμε πολύ σημαντικές αποκλίσεις ό,τι αφορά ε, την δράση της Τουρκίας στην Συρία. Τον περσμένο Οκτώβριο το Συμβούλιο καταδίκασε την ε, στρατιωτική επέμβαση της ε, Τουρκίας στη Βανατολική Συρία πρέπει όμως ε, να αναγνωρίσουμε ότι υπάρχουν και σημεία όπου τα συμφέροντά μας συμπίπτουν. Η Τουρκία έχει επιδείξει αλληλεγγύη, έχει επιδείξει γενοδορία σε πάνω από 3,5 εκατομμύρια Σύριους πρόσφυγες και έχει δώσει διασυνοριακή συνδρομή και βοήθεια προς τους ανθρώπους αυτούς. Ε, βεβαίως ε, λυπάμαι για την απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας να μην συνεχίσει να αφήνει ανοιχτά τα σύνορα ε, με την Τουρκία για να μπορέσει να περάσει ανθρωπιστική βοήθεια. Χρειάζεται βεβαίως μια πιο καλή συνεργασία σε, σε ό,τι αφορά τη Λιβύη. Ε, θυμίζω ότι χθες στην παρέμβασή μου στο Συμβούλιο Ασφαλείας ε, το επισήμενα αυτό, υπογράμμισα τη σημασία της διαδικασίας του Βερολίνου και ότι εμεί δεσμευόμαστε να εφαρμόσουμε το εμπάργκο στα όπλα των ΗΠΑ με τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας, αυτά που έχουμε. Με την επιχείρηση Ειρήνη θα συνεχίζουμε να παρακολουθούμε την, το ύποπτο εμπόριο όπλων. Ε, βεβαίως ε, είναι ανησυχητικό αυτό που κάνει η Τουρκία με τα ελληνικά νησιά ε, και υπάρχει και το μνημόνιο με τη Λιβύη εμείς προφανώς δεν αναγνωρίζουμε την ισχύ αυτού του μνημονίου σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης το μνημόνιο Λιβύης Τουρκίας έχουμε στείλει σαφή μηνύματα προς την Τουρκία για τα ζητήματα αυτά είμαστε αποφασισμένοι να προστατεύσουμε τις αρχές μας ε, τα σύνορα, τα κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών μελών ε, και βεβαίως ε, θα προσπαθούμε πάντα να, να βρούμε μια πολιτική λύση και στο ζήτημα της Συρίας και στο ζήτημα της Λιβύης. Η Τουρκία είναι σημαντικός εταίρος, είναι μια υποψήφια χώρα, είναι ένα σύμμαχο στα πλαίσια του ΝΑΤΟ και αυτή η αρνητική τάση που υπάρχει στις σχέσεις μας τα τελευταία χρόνια, το είπα και στην Άγκυρα πριν από μερικές μέρες στους Τούρκους ε, συναδέλφους μου ε, η αρνητική τάση που υπάρχει λοιπόν στην ε, σχέση μας πρέπει να αλλάξει, πρέπει να ανατραπεί. Αυτά τα αντίπεινα δεν δημιουργούν ασφάλεια για τη Μεσόγειο. Η ασφάλεια θα έρθει μέσω διαλόγου, μέσω συζητήσεων. Βεβαίως και υπάρχουν διαφωνίες και αποκλήσεις. Αυτό συζητούσα με τους Τούρκους ομολόγους μου στην τελευταία μου επίσκεψη. Έχουμε πολλά κοινά συμφέροντα, του είπα, πάνω στα οποία μπορούμε να οικοδομήσουμε μια σχέση. Ε, και θα εξετάσουμε ε, το πώς θα προχωρήσουμε στο Συμβούλιο Εξωτερικών ε, τη Δευτέρα. Τρίτο ζήτημα, Λευκορωσία. Θα ήθελα καταρχήν να σας αναφέρω τις τελευταίες εξελίξεις. Σας ε, διαβεβαιώ ότι παρακολουθούμε πολύ στενά την κατάσταση εκεί μετά τις την προεδρική εκλογή της 9 η Αυγούστου ανησυχούμε για τους περιορισμούς ελευθεριών, ε, ελευθερίας συνάθρησης, ελευθερίας έκφρασης, διώξεις ε, δημοσιογράφων. Πρέπει να σταματήσει επίσης η παρενόχληση και η δίωξη των ε, ηγετών της αντιπολίτευσης. Πρέπει να μπορούν όλοι να ασκήσουν τα αστικά τους, τα πολιτικά τους δικαιώματα. Ελπίζουμε να μας καλέσει η Λευκορωσία το μέτρο δυνατόν ε, για να παρακολουθήσουμε τις μελλοντικές προεδρικές εκλογές ε, έχουμε ζητήσει την άμεση και χωρίς όρους απελευθέρωση όλων των αντιφρονούντων και θα παρακολουθούμε βεβαίω στενά, θα παρακολουθούμε στενά τις εκλογές αυτές στη Λευκορωσία έτσι ώστε να υπάρχει κυριαρχία, ε, ανεξαρτησία, ελευθερία στη Λευκορωσία. Είναι ο μόνος δρόμος για να οικοδομηθεί ένα μέλλον ευημερία για τους πολίτες της χώρας αυτής. Η Λευκορωσία έχει αποδείξει ε, με την ενεργή τη συμμετοχή ότι θέλει αυτή την εταιρική σχέση. Ε, έχουμε πετύχει ε, σημαντικά ωφέλη για τους πολίτες της Λευκορωσίας, όπως παραδείγματος χάρη διευκόλυνση ε, χορήγηση θεωρήσεων από τον Ιούλιο, από τις αρχές Ιουλίου. Η οικονομική συνεργασία με τη χώρα αυτή είναι αμοιβαία επικερδής ε, Έχουμε ένα συνεχή διάλογο για να βελτιωθούν τα πρότυπα και προδιαγραφέ και για την κλιματική αλλαγή, τα περιβαλλοντικά πρότυπα. Αυτό είναι σημαντικό για όλου του Ευρωπαίου. Ελήψη ενό νομικού δεσμευτικού πλαισίου συμφωνία, οι προτεραιότητε ε, τη εταιρική σχέση Ευρωπαϊκή Ένωση και Λευκορωσία ε, και το σχετικό συμφωνητικό ε, εξακολουθεί να αποτελεί προτεραιότητα. Βεβαίω πρέπει να λάβουμε υπόψη μα και την ανθρωπινά δικαιώματα και την πυρηνική ασφάλεια Αυτά είναι στοιχεία που θα μας δώσουν μεγαλύτερη διαφάνεια, μεγαλύτερη λογοδοσία στις σχέσεις με τη χώρα αυτή. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, θα πρέπει εμείς να παραμείνουμε ανοιχτοί στις περαιτέρω εξελίξεις ε, των σχέσεών μας με τη Λευκορωσία και να ασχίσουμε να υποστηρίζουμε την ε, ανεξαρτησία της χώρας αυτής και την κυριαρχία της όμως αυτές οι εξελίξεις μπορούν να βαστούν μόνο σε θετικά βήματα στον τομέα των δικαιωμάτων, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, των θεμελιωδών ελευθεριών. Και επανέρχομαι βεβαίω στα αρχικά μου λόγια. Στις 9 Αυγούστου, στις προεδρικές εκλογές, ε, θα δούμε πώς θα προχωρήσουμε από εκεί και πέρα με βάση τις εκλογές αυτές. Αυτό είναι που θα καθορίσει την πραγματικότητα της σχέσης μας. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σα. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Αντιπρόεδρε. Και τώρα ξεκινά η συζήτηση με το γύρο των εκπροσώπων πολιτικών ομάδων. Ο κύριο Βέμπερ, εκ μέρου του ΕΛ, καταρχά. Έχετε τώρα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε εκπρόσωπε ε, Μπορέλ. Στην σημερινή μου παρέμβαση από τη συνάδελφη θα μιλήσω με την Τουρκία. Έχουμε πολλούς ε, κοινούς δεσμούς με την ε, Τουρκία, οικονομικούς, ιστορικούς, ε, μέλος του ΝΑΤΟ είναι και σίγουρα πολλοί Ευρωπαίοι ζουν στην Τουρκία και πολλοί Τούρκοι στην Ευρώπη και φυσικά υπάρχει η δέσμευση των Τούρκων σε ό,τι αφορά το θέμα των προσφύγων. Όμως υπάρχουν κάποια ζητήματα. Εξού και είχαμε ζητήσει ο να γίνει αυτή η σημερινή συζήτηση ότι έχουμε ανησυχίε. Παραδείγματο χάρη σε ό,τι αφορά τι ε, συνεχεί επιθέσει ε, ε, στα σύνορα ε, με την Ελλάδα, οι γεωτρητικές εξορρυκτικές δραστηριότητες ε, και στα θέματα που άπτονται της ελευθεροτυπίας ε, υπάρχουν μεγάλες πιέσεις και οι προωθήσεις των μεταναστών στα σύνορα. Ήθελα λοιπόν να ε, πω πρώτα απ' όλα ε, για τον κύριο Αναστασιάρ και τον κύριο Μητσοτάκη ε, ένα μεγάλο ευχαριστώ για τις προσπάθειες που κατέβαναν το Φεβρουάριο που είδαμε να έχουμε αυτές τις επιθέσεις της πρόθεσης ουσιαστικά παράνομων μεταναστών και το μήνυμα ουσιαστικά πίσω από ε, την ε, αντίσταση ε, ήταν της Ελλάδας και της Κύπρου είναι ότι δεν θα αφήσουμε τον Ερντογάν να μας εκβιάζει διότι δεν πρόκειται μόνο για την Ελλάδα και την Κύπρο πρόκειται για την Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν θα αφήσουμε αυτά τα δύο κράτη της Ένωσης μόνα τους. Αυτό λοιπόν το μήνυμα που έχουμε απέναντι στον κύριο Ερντογάν είναι ότι ναι είμαστε έτοιμοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση να έχουμε μια εταιρική σχέση με την Τουρκία να επανέλθουμε στις διαπραγματεύσεις θέλουμε όμως έναν εταίρο που θα ε, συμμετέχει σε αυτή την προσπάθεια. Δεν είμαστε αφελείς ε, και η Τελωνιακή Ένωση που ξέρουμε ότι είναι υπαρξιακή οικονομική σημασία για την Τουρκία, είναι ένα από τα εργαλεία που θα έχουμε για να ασκήσουμε πιέσει προ την Τουρκία. Θέλω να υπάρχουν ειλικρινεί διμερεί σχέσει. Έχουμε ε, ξεκινήσει κάποιε συνομιλίε ε, και ενταξιακέ κάποια στιγμή, οι οποίε ήταν ένα λάθο και δημιούργησαν ε, πάρα πολλέ προσδοκίε. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει αυτό το κεφάλαιο να κλείσει και να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο σε σχέση με την εταιρική μα σχέση. Σίγουρα πρέπει να συζητήσουμε Τουρκία, αλλά ο στόχο μα πλέον θα πρέπει να είναι μια νέα εταιρική ε, σχέση. Ευχαριστώ πολύ κύριε Βέμπερ, ε, λέει πρόεδρος εκ μέρους ε, των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Τώρα το λόγο έχει η κυρία Σάντο. Παρακαλώ έχετε το λόγο κυρία Σάντο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κύριε, είπατε εκπρόσωπε. Σήμερα εξετάζουμε ακόμη μια έκθεση για την δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα παντού στον κόσμο. Δυστυχώ όμω δεν διαπιστώνουμε κάποια θετική αλλαγή. Και σύμφωνα με αυτήν την έκθεση μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι οι αλλαγές αργούν να έρθουν και θα μπορούσαμε να πούμε ότι ε, έχουμε ακόμα μία έκθεση γιατί κάθε χρόνο λέμε για τα θύματα του ρατσισμού, λέμε για ηθαγενείς πληθυσμούς που τους πετάνε έξω από τη γη τους, λέμε για το πόσο φημώνονται, καταδιώκονται και φωνεύονται ακτιβιστές για τα ανθρώπινα δικαιώματα και αυτούς όλους που υποφέρουν απάνθρωπη συμπεριφορά, βάσει ιστήρια φεύγει ο κόσμος να ξεφύγει, να αναδραπετεύσει από τον πόλεμο, από την πείνα. Πολλές φορές αυτός ο κόσμος ε, πεθαίνει προσπαθώντας να περάσει στην Ευρώπη, εδώ στα σύνορά μας, εκεί που προσπαθούν να βρουν την ευκαιρία για μια καλύτερη ζωή, ασφάλεια, αξιοπρέπεια. Ε, ε, οπότε σε αυτή την έκθεση διαπιστώνουμε ότι είναι εκατομμύρια εκείνοι οι οποίοι απαιτούν σεβασμό των δικαιωμάτων, απαιτούν δικαιοσύνη, όλα αυτά τα οποία πασχίζουμε κι εμείς να ισχύουν για όλους, ε, διαβάζουμε στην έκθεση ε, για το ότι ε, πρέπει να βλέπουμε τι γίνεται σήμερα και να μην κουβεντιάζουμε το αύριο. Θα πρέπει να μην συμβαζόμαστε όσον αφορά τις πολυμερεί δημόσιε σχέσει. θα πρέπει να μην υπάρχει ατιμορρησία, θα πρέπει να λάβει δράση η Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει να προστατεύσουμε το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο έναντι αυτών των ντροπιαστικών επιθέσεων που δέχεται, να υπάρξουν κυρώσει κατά αυτών που καταπατούν τα ανθρώπινα δικαιώματα θα πρέπει να υπάρξει ένας μηχανισμός της δέουσας επιμέλειας να είναι υποχρεωτικός για τα ανθρώπινα δικαιώματα ε, δεν θα πρέπει να έχουμε προϊόντα ε, που παράγονται με καταπάτηση δικαιωμάτων ε, θα πρέπει να έχουμε τέτοια μεσταναστική συμπεριφορά που να μας τιμά. Ευχαριστώ πολύ. Ροντρίγκε Ράμο, ε, τώρα εκ μέρου τη Renew Europe. Θα έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Εκπατεκπρόσωπε. Η ε, παρουσίαση αυτής της έκθεσης ε, είναι πάρα πολύ σημαντική γιατί ουσιαστικά μιλάμε και για έναν οδικό χάρτη της στρατηγικής για τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Υπάρχουν θετικά επιτεύγματα, τα είπατε κι εσείς. Ωστόσο υπάρχουν ε, και πάρα πολλά αρνητικά στοιχεία τα οποία αναφέρονται σε αυτή την έκθεση. Ένα θετικό που θέλω να πω είναι ότι αναγνωρίζεται η κλιματική αλλαγή και η απώλεια βιοπικιλότητας. Αναγνωρίζεται ως μια σημαντική απειλή σε βάρος των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Ανοίγει ένας σωστός δρόμος πιστεύω. Όμως το 2019 ουσιαστικά ε, θα μείνει ως ένα πολύ κακό έτος γιατί ήταν πολύ καλό έτος για το λαϊκισμό που κάνει πιο εύθραυστες τις δημοκρατίες και επιδεινώνει τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις ελευθερίες. Κάθε φορά περισσότερο βλέπουμε ότι η αποδυνάμωση των δημοκρατιών μας γίνεται εκ των έσω, δηλαδή με τη χρήση δημοκρατικών θεσμών για τη δημιουργία ε, απολυταρχικών, αυταρχικών ε, καθεστώτων. Το βλέπουμε το βλέπουμε πώς γίνεται. Επίθεση σε βάρος ε, της δικαστικής εξουσίας, σε βάρος του τύπου. Η ελευθεροτυπία, θεμελιώδες δικαίωμα. Γι' αυτό λοιπόν ε, οι δημοκράτες, ε, κύριε Πατεκπρόσωπο, δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να επιτρέψουμε να, να θεωρηθεί κάτι λογικό η παρενόχληση της ελευθεροτυπίας ε, και ε, να μιλάμε μόνο. Πρέπει να κάνουμε έργα. Θέλουμε λοιπόν ε, μια στρατηγική συνεπή υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πάνω απ' όλα αυτή τη χρονική περίοδο πρέπει να εργαστούμε υπέρ του πολυμερούς συστήματος, της πολυμερούς προσέγγισης. Να υπερασπιστούμε δηλαδή τη νομιμότητα, γιατί έτσι υπερασπιζόμαστε όλων τα δικαιώματα. Επίσης, είπατε εκπρόσωπε, θα πρέπει να επιτρέψουμε και να επιταχύνουμε το θεματολόγιο 2030, ιδίως ό,τι αφορά το κεφάλαιο και το στόχο 16. Τέλος, θα πρέπει πολύ σημαντικό και αυτό και αυτονόητο για μια μεγαλύτερη δημοκρατική ανθεκτικότητα, προώθηση της ε, μετανάστευσης ε, υπό το πρίσμα όμως ε, των δικαιωμάτων κατά των αποθεσιών και κατά των επιπτώσεων της παράτυπης μετανάστευσης. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Ροντρίγε. Συνεχίζουμε με την ταυτότητα και δημοκρατία και τον κύριο Μπέργκ. Παρακαλώ έχετε το λόγο. Κυρία Πρόεδρε, κύριε Πατεκπρόσωπε, η έκθεση ε, απευθύνεται στην κατάσταση και στα επιτεύγματα σε όλες τις χώρες. Αλλά ε, πολλές φορές ε, θα πρέπει να βλέπουμε κατά πρόσωπο την πραγματικότητα. Ε, στην Ιεμένη πρέπει να στρέψουμε τα βλέμματά μας. Στόχος των παραστατικών ομάδων εκεί είναι γυναίκες και παιδιά. Πάρα πολύ κακές συνθήκες οι υγιεινής που οδηγούν σε πάρα πολύ μεγάλες μερίδες αυτού πληθυσμού να πλήττονται από ασθένειες οικογένειες, χάος και παρόλα αυτά πολύ λίγα πράγματα λέει η έκθεση γι' αυτό. Έχουμε ε, θέσει αυτό το ε, θέμα ουσιαστικά στα χέρια του ΕΚΕ της Σαουδικής Αραβίας ε, και των χωρών της περιοχής. Έχουμε επίσης ένα κεφάλαιο για την θρησκευτική ελευθερία, αλλά δεν μιλάμε συγκεκριμένα για την Δυτική Αφρική και τις διώξεις των χριστιανών που διώκονται για τις πεπιθήσεις τους, για τα πιστεύω τους. Λέμε για τις γυναίκες τις Αφγανές και σίγουρα ένας πολύ αξιέπαινος στόχος και η χειραφέτησή τους και όλα αυτά. Όμως, ε, ναι μην είναι σημαντικό να υποστηρίξουμε τις Αφγανές, αλλά τι θα κάνουμε σε σχέση ε, με την ε, πολιτική κατάσταση εκεί. Λέμε τίποτε για τις εκλογικές νοθευμένες διαδικασίες εκτελέσεις και τις δράσεις της κυβέρνησης. Ας τα βλέπουμε λοιπόν τα πράγματα πιο αντικειμενικά και όχι με κομματικά γυαλιά να υποστηρίξουμε τους αδύνατους και να μην ε, χαιρόμαστε με κάποιες ε, ε, περιστασιακές τέτοιες εξέλιξεις. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Νόημαν εκ μέρους των Πρασίνων έχει τώρα το λόγο. Κύριε Μπορέλα, ξέρετε συνάδελφοι, στο ψήσιμο του Κοινοβουλίου μιλήσαμε για την έκθεση του 2019 για τα ανθρώπινα δικαιώματα και ζητήσαμε συντονισμένη διαδικασία για τη χορήγηση θεωρήσεων σε όσου υπερασπίζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και για άλλη μια φορά βρίσκομαι εδώ σήμερα και δεν έχει γίνει τίποτα έκτοτε. Ακόμα χειρότερο, όταν ζήτησα από την Κομισιόν γι' αυτό το Μάρτιο, η Κομισιόν μου απάντησε το εξή. Η Κομισιόν δεν γνωρίζει να υπάρχουν συστηματικά προβλήματα όσων υπερασπίζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα, έτσι ώστε να μπορούν να έχουν πρόσβαση στη, στην, στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς θεώρηση. Το λέτε σοβαρά αυτό. Στις 15 Οκτωβρίου πέρυσι ένας 25χρονος ε, ακτιβιστής του LGBTI ε, ζήτησε ε, μια θεώρηση για να έρθει εδώ να μιλήσει. Δεν έλαβε ποτέ θεώρηση. Αύριο ο κ. Γκογκύρ θα δικαστεί στην Τουρκία για οργάνωση μίας ε, διαδήλωσης χωρίς καμία βία ε, για, για τα δικαιώματα των, ε, της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ. Ε, διότι λέμε ότι για να το δοχωρήσουμε θεώρηση δεν πρέπει κάποιος να έχει πάει φυλακή ή να είναι σε, σε αντιπαράθεση με τις το, κυβερνητικές αρχές. Είναι δυνατόν οι άνθρωποι αυτοί κινδυνεύουν ακριβώς γιατί τους κυνηγούν οι αρχές και κάνουν κάτι του οποίου του ενθαρρύνουμε να το κάνουν και μετά λέμε ότι δεν έχουμε συστηματικά και συστημικά προβλήματα. Κύριε Μπορέλ, το γνωρίζετε πολύ καλά, όπω και εγώ. Οι υπερασπιστέ ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι εταίροι μα. Χωρί αυτού δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα όταν μιλάμε για την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και ο χώρο του συρρυκνώνεται. Και οι δικέ μα πολιτικέ θεωρήσεων έρχονται να συρρυκνώσουν ακόμα περισσότερο τον χώρο αυτών. Σα ζητώ λοιπόν να αποκοινούμε την Επίτροπο Γιώχανσον να κάνει μια προσπάθεια για να σταματήσει αυτή η αδικία έτσι ώστε να μπορούν οι άνθρωποι αυτοί να ταξιδεύουν, να δημιουργούν δίκτυα, να πηγαίνουν σε διασκέψεις. Ο ρόλος μας είναι να προωθήσουμε, να προστατεύσουμε όσου υπερασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και δημοκρατία και όχι να δυσκολεύουμε ακόμα περισσότερο τη ζωή του. Σα ευχαριστούμε πολύ εκ μέρους ε, των Ευρωπαίων Συντηρητικών Μεταρρυθμιστών ε, Ρόισεν. Έχετε το λόγο. Κυρία Πρόεδρε, κύριε Μπορέλ, συνέχεια δέχομαι μηνύματα στο κινητό μου για βία, για επιθέσεις που καταλήγουν πολλές φορές σε θάνατο όλα αυτά γιατί είμαστε χριστιανοί και μόλις χθες μου είπαν για κάποια γυναίκα που δολοφονήθηκε ενώ σε ένα δάσος μάζευε ξύλα. Άφησε τέσσερα ορφανά. Αυτά στην ιδέα και θα πρέπει να δείτε τι θα γίνει με την παράταση της ε, εντολής για την ελευθερία πίστης. Θα πρέπει να αναθεωρήσετε αυτή την απόφαση. Κάτι πρέπει να κάνετε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρξει εκεί προσωπικό περισσότερο από ότι στο παρελθόν η μονάδα για την ελευθερία της πίστης δεν πρέπει να είναι τόσο α, άσχημα επανδρομένη. Η ελευθερία της πίστης δεν έχει την προτεραιότητα που πρέπει στην ευρωπαϊκή ατζέντα. Θα πρέπει να πιέσετε κάθε φορά που κλείνετε τις εμπορικές ε, συμφωνίες να πιέζετε εκεί που η ελευθερία πίστης δεν υπάρχει. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Είμαστε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και δεν πρέπει να διστάζουμε. Ο κύριος Ουρμπάν Κρέσπο για την ΚΟΕ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Μπορέλη, το 2019 η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, λέει ότι ηγήθηκε της προστασίας τη προώθησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Για μένα ήταν η χρονιά που φτάσαμε στη συμφωνία του Μερκοσούρ ενώ ο Μπολσονάρο ε, έκαιγε τον Αμαζόνιο ή προωθούσε την ε, δίωξη των Ιθαγενών. Το 2019 επίσης ε, η Καρόλα Ρακέτε ποινικοποιήθηκε και άλλες μη κυβερνικές οργανώσεις επειδή έσωζαν ανθρώπινες ζωές από σίγουρο θάνατο στη Μεσόγειο. Ενώ το κοινοβούλιο, αυτό το Ευρωκοινοβούλιο, δεν δεχόταν, απέρριψε το ψήφισμα για να συνεχιστούν οι επιχειρήσεις ε, αναζήτησης και διάσωσης στη Μεσόγειο. Αγνοήσαμε το διεθνές δίκαιο, επικυρώσαμε μια εμπορική συμφωνία με το Μαρόκο που περιλαμβάνει και τα κατεχόμενα εδάφη της Σαχάρας. Ξέπλυμα λοιπόν ανθρωπίνων, ε, ε, εγκλημάτων ανθρωπίνων δικαιωμάτων όπως ε, του, της κυβέρνησης του Ερντογάν και του Αλ Να το κρίνετε εσείς, για μένα είναι σαφές, πρέπει να σταματήσουμε να δίνουμε μαθήματα και να αρχίσουμε να δίνουμε παράδειγμα. Εμείς να ε, τηρούμε τα ανθρώπινα δικαιώματα στις εμπορικές συμφωνίες, να τηρούμε τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Μεσόγειο, να τηρούμε τα ανθρώπινα δικαιώματα και στο ευρωπαϊκό έδαφος. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος ε, Καστάλτο δεν είναι παρόν. Προχωρούμε λοιπόν με τον κύριο Λόπεθ Χίλ, εκ μέρους του ΕΛΚ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η έκθεση την οποία συζητούμε σήμερα ε, σηματοδοτεί το τέλος ε, ε, της περίοδου 2015-2019. Ένας από τους στόχους του σχεδίου 2015-2019 είναι η αντιμετώπιση των βασανιστήριων. Είναι ένα σημαντικό εργαλείο που υπάρχει γι' αυτό. Ο διάλογος για τα ανθρώπινα δικαιώματα με τρίτες χώρες, όπως με την Κούβα τον Οκτώβριο του 2019 όπου δυστυχώς ξεκολουθούν να υπάρχουν ε, πολιτικοί κρατούμενα, κρατούμενοι ε, κρατήσεις αυθαίρετες και συλλήψεις. Ε, ένας άλλος στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να προωθεί τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στην υπόλοιπο κόσμο. Το 2019 είχαμε 8 αποστολές παρατήρησης και 7 αποστολές εμπειρογνωμών για να υποστηριχθούν οι εκλογικές διαδικασίες. Αυτά μπορούν να βοηθήσουν για μια πολιτική μετάβαση στη Βενεζουέλα με δίκες, ελεύθερες εκλογές ε, έτσι ώστε να σταματήσει το καθεστώς ε, να προσπαθεί να καταλύσει τη δημοκρατία ε, και να καθορίζει την πολιτική ζωή της χώρας. Χρησιμοποιήστε όλα τα εργαλεία που έχετε στη διάθεσή σα, κύριε Πατεκπρόσωπε, στη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα να επανέλθουν στι χώρε όπου δεν υπάρχουν. Σας ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Αρενά, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Κύριε είπατε πριν από το COVID τα ανθρώπινα δικαιώματα σε πολλές περιοχές του κόσμου ε, υποχωρούσαν. Όμως η πανδημία μόνο χειροτέρευσε τα πράγματα. Μια τεταμένη κατάσταση ήδη ε, και βεβαίως η πιο ευάλωτη είναι αυτοί οι οποίοι πληρώνουν το μάρμαρο. Είδαμε κινήματα νέων και λιγότερων νέων και πριν το COVID που έτυχαν καταστολής κατά τη διάρκεια του εγκλισμού στην Αλγερία, στο Χονγκ Κόνγκ, στη Χιλή. Αυτό αυτά τα κινήματα δημιουργούνται επειδή υπάρχουν ε, βαθιά προβλήματα. Το είδαμε και στι δικέ μα δημοκρατίε, στι ΗΠΑ με το Black Lives Matter και στην Ευρώπη. Είναι αλήθεια ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε καταφέρει να αναπτύξουμε μια πολιτική ανθρωπίνων δικαιωμάτων φιλόδοξη και στεναρή. Και σα ε, ε, συγχαίρω που υπάρχει ένα νέο μηχανισμό κυρώσεων για να αντιμετωπιστούν αυτέ οι πραγματικότητε όπου παραβιάζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Πρέπει όμω να είμαστε να είμαστε πιο συνεπεί στι πολιτικέ μα. Οι ευρωπαϊκέ πολιτικέ πρέπει να σέβονται τι συνθήκε ιδιαίτερα το άρθρο 21 τη συνθήκη. Είτε μιλάμε για την εμπορική πολιτική, είτε μιλάμε για τη μεταναστευτική πολιτική, είτε μιλάμε για την ανθρωπιστική πολιτική, την πολιτική ανάπτυξη, την πολιτική για το κλίμα, για το περιβάλλον. Όλε αυτέ οι πολιτικέ πρέπει να σέβονται την αρχή ότι δεν πρέπει να οπλίζουμε, δεν πρέπει να ενθαρρύνουμε την αποδυνάμωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον κόσμο. Πρέπει να είμαστε πιο φιλόδοξοι λοιπόν στην πολιτική μα. Χρειαζόμαστε πιο αποτελεσματικέ ρυθμίσει, πιο συμπεριληπτικέ ρυθμίσει που να συμπεριλαμβάνουν δηλαδή την κοινωνία των πολιτών. Θα πρέπει επίση να αντιμετωπίσουμε την ατιμορρησία ε, υποστηρίζοντα το Διεθνέ Ποινικό Δικαστήριο. Ευχαριστώ πολύ. Σα ευχαριστώ. Επόμενο ο κύριο Άντριου. Παρακαλώ, έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, κύριε Πατεκπρόσωπε, δράτω με της ευκαιρίας ε, για να σας παρακαλέσω να ορίσετε έναν ειδικό ε, εκπρόσωπο για το Συριακό. Ξέρω ότι υπάρχει απεσταλμένος ενβόη. Δεν είμαστε ΟΗΕ ε, και δεν είναι ακόμη ξεκάθαρα τα πράγματα, αλλά μόνο έτσι ε, θα μπορέσουμε να οδηγήσουμε σε Δεν μπορούμε να αφήσουμε την μοίρα αυτών των ανθρώπων στη Ρωσία. Και ξέρετε ότι η ανθρωπιστική βοήθεια που θα έπαιρναν δύο εκατομμύρια Σύριοι σταματά από αύριο λόγω του στο βέτο που άσχεσε η Κίνα και η Ρωσία σε αυτό το ψήφισμα ε, για την παράταση, ε, να, να παραταθεί δηλαδή. Πραγματικά νιώθω ντροπή. Νιώθω ε, ντροπή απέναντι στην αδυναμία της διεθνούς κοινότητας να προστατεύσει αυτά τα άτομα. Είχαμε εξαφανίσεις, χημικές επιθέσεις, επιθέσεις σε δομές αμάχων. Και τώρα δεν μπορούμε ούτε καν να εξασφαλίσουμε την παροχή ανθρωπιστική βοήθειας. Σας παρακαλώ λοιπόν σήμερα να ορίσετε έναν ειδικό εκπρόσωπο που θα ξεκινήσει τη διαδικασία ανάπτυξη σχέσεων για μια βιώσιμη ειρήνευση ε, ε, στη Συρία. Ευχαριστώ πολύ. Συνεχίζουμε. Το Βαλιέρι είναι ο επόμενος ομιλητής. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η Ευρώπη υποπτεύει την ε, τη συνδρομή δικαιωμάτων και αυτό είναι κάτι το αξιόλογο, αλλά θα πρέπει βέβαια να γίνει έρευνα, θα πρέπει να γίνουν καταγγελίε και αυτό θα πρέπει να γίνει με αποφασιστικότητα όσον αφορά την παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Αλλά πρώτα πρώτα να δούμε τι γίνεται εδώ στο περιβόλι μα, γιατί έχουμε όλο ένα και περισσότερε παραβιάσει λόγω τη μαζική μετανάστευση από τι Ισλαμικέ χώρε. Και αυτοί οι άνθρωποι μαζί του παίρνουν κάποια αρχαϊκά έθιμα. Ε, έχουμε τους ακροτηριασμούς των ε, γυναικών, μόνο 70.000 στη Γερμανία. Έχουμε ε, κάποιους γάμους ανηλίκων υποχρεωτικούς, έχουμε το ε, την μπουρκα και ε, αυτό γίνεται υπό την σιωπή της διεθνούς κοινότητας. Θα πρέπει πρώτα-πρώτα αυτά να καταγγελματά τι γίνονται στο σπίτι μας. Βέβαια αυτό είναι πιο άβολο από όταν λέμε για τα στατιστικά στοιχεία σε όλο κόσμο. Αλλά δεν θα πρέπει πια να κολλησιεργούμε. Θα πρέπει να έχουν οι κυβερνήσεις της κάθε ευρωπαϊκής χώρας το θάρρος που τους λείπει μέχρι τώρα. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει αντιπρόεδρος κυρία Χάουταλα. Κύριε, κυρία Πρόεδρε. αξιότιμη είπατε εκπρόσωποι. Στην ετήσια έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα, το φάσμα των δραστηριοτήτων και πρωτοβουλειών στον τομέα επιχειρήσεων και ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι κάτι αξιέπαινο. Ωστόσο, δικαιώματα που δεν μπορούν ε, νομίμως να ε, εφαρμοστούν στην πράξη, ουσιαστικά μένουν στο χαρτί. Επί σειρά ετών και ε, μετά από προσ... τις προσπάθειές μας ε, επί σειρά ετών λοιπόν να βλέπουμε να αρχίζει να γίνεται αποδεκτή ανάγκη αποδεκτή, ε, υποχρεωτικής ε, νομοθεσίας, δεσμευτικής νομοθεσίας για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις επιχειρήσεις. Ε, είχαμε ένα ορόσημο στα τέλη Απριλίου. Ο Επίτροπος Δικαιοσύνης Ράιντερς είπε ότι θα πρέπει να υπάρχουν ε, υποχρεώσεις δεούσα επιμέλεια στον τομέα αυτό για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε ευρωπαϊκό έδαφος. Και τώρα η Γερμανική Προεδρία δεσμεύθηκε σε ένα σχέδιο δράσης ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Κάτι που το περιμέναμε εδώ και καιρό. Διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δείχνει μεγάλη επιμέλεια ε, ως προς τα κράτη-μέλη για να εγκρίνουν αυτά σχέδια ε, δράσης. Αλλά πολλές φορές, ξέρετε όπω λέμε, ε, τα παιδιά των ε, ε παπουτσίδων ε, είναι ξυπόλυτα. δηλαδή είναι καιρός να γίνει και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης το ίδιο. Τώρα νομίζω ότι είναι πολύ κατάλληλη η χρονική στιγμή για να αρχίσουμε με νόημα να ε, ασκούμε την επιρροή μας και στο πλαίσιο του ΟΗΕ και στις γενικότερε διαπραγματεύσεις σε σχέση με τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Παρακαλώ λοιπόν ζητήστε εντολή από τα κράτη-μέλη για να ξεκινήσει αυτή ε, η πρωτοβουλία. Ευχαριστώ πολύ πρόεδρο. Ε, ο κύριο Πουτσιτεμών έχει τώρα το λόγο. E committed to the defense of human rights around the world η Ευρωπαϊκή Ένωση πασχίζει την ανθρώπινη δικαιώματα σε όλο τον αλλά για να είμαστε αποτελεσματικοί ω Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να έχουμε και το ηθικό κύρο. Δεν το έχουμε. Και δεν το έχουμε διότι η Ευρώπη ανέχεται, ανέχεται την κράτηση, την φυλάκηση ηγετών πολιτικών σε χώρε τη όπω η Ισπανία. Οπότε δεν έχει έτσι αξιοπιστεί εναντίον των τριών χρόνων. Είδατε, λέμε για την Τουρκία πριν από ένα χρόνο αποφάσισε η τουρκική κυβέρνηση να καταργήσει κάποιους δημάρχους του Κουρδιστάν. Αυτοί οι δημάρχοι είχαν ε, ε, εκλεγεί δημοκρατικά και ε, από την άλλη μεριά είδατε τι έγινε και στην Ισπανία με κάποιους πολιτικούς υπέρ της ανεξαρτησίας στη χώρα των Βάσκων και στην Καταλωνία χωρίς δίκη, χωρίς δίκη τους καταργήσανε οπότε δεν βλέπω να γράφετε τίποτα σε αυτή την έκθεση τίποτα για τους Κούρδους. Σε άλλες ε, εκθέσεις όμως γράφονται αυτά όπως ε, το Human Rights Watch, το παρατηρητήριο των ανθρώπινων δικαιώματα, κύριε Μπορέλ. Ε, το κάνετε, όλος ο κόσμος θα σας ευχαριστήσει. Ευχαριστώ. Προχωρούμε τον κύριο Μιλιάν Μον. Πρόεδρε, ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, είναι βασικό γνώρισμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εξωτερική πολιτική ε, δεν μπορεί ε, να παραγνωρίζει αυτή τη διάσταση. Πρέπει να συνεχίσει λοιπόν τι προσπάθειέ μα ε, με τι εκθέσει για την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ανά τον κόσμο. Σε γενικέ γραμμέ, οι χώρε που σέβονται ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτο δικαίου είναι και αυτέ που υποστηρίζουν ένα διεθνέ δίκαιο που βασίζεται στην ειρήνη. Αυτό είναι που επιθυμούμε εμεί οι Ευρωπαίοι. Το Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών του περασμένου Δεκέμβριου αποφάσισε να ξεκινήσει ένα γενικό καθεστώς κυρώσεων ε, για τις παραβιάσεις των δικαιωμάτων και υπάρχει ένα σχετικό ε, κείμενο της, των προτεραιοτήτων της Γερμανικής Προεδρίας ε, για το ζήτημα αυτό. Θα ήθελα να γνωρίζω λίγο πιο λεπτομερώς ποιοι είναι οι στόχοι ε, αυτών των εργασιών. Βεβαίω και πρέπει να βελτιωθούν οι μηχανισμοί για να μπορέσουν να επιβληθούν οι κυρώσεις. Δεν μπορούμε να επαναλάβουμε αυτά που συνέβησαν στη Μαδρίτη τον περασμένο Ιανουάριο. Ευχαριστώ πολύ. Βόλατ είναι επόμενο μητέρα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πατεκπρόσωπε. Έχω ένα λεπτό και θα ήθελα να εστιάσω στην ε, Τουρκία διότι συστηματικά καταπατά το διεθνέ δίκαιο και αποσταθεροποιεί την ευρύτερη περιοχή ε, και πρέπει να βλέπουμε τι γίνεται στην Βόρεια Συρία από την Τουρκία. Οι Κούρδοι εκεί και ιδίω οι θρησκευτικέ μειονότητε, οι γεσιντοί ε, τρομοκρατούνται, εκφοβίζονται και εμεί εδώ συζητάμε. Προχωράει και επεμβαίνει και στον εμφύλιο στη Λιβύη όσο εμείς εδώ συζητάμε ε, και την Κύπρο, την Ελλάδα. Βλέπετε μέλη της κράτης, ε, της, κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, πώς τα εκβιάζει με πολύ επιθετική, όλο και περισσότερο επιθετική εξωτερική πολιτική προσπαθεί να επιτύχει τους στόχους, καταπατώντας τα ανθρώπινα δικαιώματα, αποσταθεροποιώντας την ευρύτερη περιοχή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μιλάμε για ανθρώπινα δικαιώματα και απαιτούμε από άλλους και εμείς θα πρέπει να τα τηρούμε, δηλαδή στα εξωτερικά μας σύνορα. Και μετά να μιλήσουμε και ε, να είμαστε και αξιόπιστοι για τα δικαιώματα σε εξωτερικό επίπεδο. Ευχαριστώ πολύ. Τούμα είναι τώρα η επόμενη ομιλήτρια. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Πέρα, αγαπητή συνάλφη, είναι καλοδεχούμενη αυτή η συζήτηση. Τουλάχιστον δείχνει ότι η Ένωση μα εδράζεται επί αξιών. Συμφωνώ με τα όσα είπαν οι περισσότεροι συνάλυφοι που προηγήθηκαν. Ε, Να πω κάτι ακόμα. Στο 2019 έχουμε μιλήσει πολλές φορές για τα ανθρώπινα δικαιώματα ε, και στο πλαίσιο της ε, Γενικής Συνέλευσης στο ΙΕ. Μιλήσαμε για τα θέματα των μειονοτήτων και στο επίπεδο του φόρουμ για ε, τις μειονότητες υπήρξε και ένα περιφερειακό φόρουμ που οργανώθηκε εδώ. Ε, και σε όλες αυτές τις ε, συνεδριάσεις, όπως λέγεται και στην ετήσια έκθεση, επισημαίνονται οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μιλάμε για τα γλωσσικά δικαιώματα, τα δικαιώματα των μειονοτήτων. Δίνουμε όμως εμείς και το καλό παράδειγμα. Αυτό είναι το θέμα. Λέει είναι προτεραιότητα το θέμα ε, των μειονοτήτων. Έχουμε εκατοντάδες χιλιάδες ε, απάτριδες, ε, ανιθαγενείς. Τι γίνεται με αυτούς, με αυτούς που δεν μπορούν να μάθουν τη γλώσσα τους, γιατί κλείνονται τα μειονοτικά σχολεία. Έχετε τεθεί αυτό το θέμα. Εγώ θέλω η συμμετοχή μας σε αυτές τις πλατφόρμες ε, για ε, τα δικαιώματα των μειονοτήτων να δώσουμε πολύ πιο πιστικά μηνύματα. Και αυτό θα το επιτυχαίναμε αν ήμασταν και πιο σωστοί εμείς εδώ σε αυτά που κάνουμε. Ευχαριστώ πολύ. Κολακούτσιτς είναι ο επόμενος ομιλητής. Κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, για να έχουμε το δικαίωμα να κουνάμε το δάχτυλο σε άλλους για τα ανθρώπινα δικαιώματα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρώτα-πρώτα να δούμε τι γίνεται εδώ, στο σπίτι μας, στο περιβόλι μας, εάν τηρούνται τα δικαιώματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ισπανία, στην Καταλωνία, υπάρχουν διώξεις, διώξεις κατά πολιτικών. Ούτε καν το θίξαμε το θέμα. Ε, είναι πάρα πολύ σημαντικό και επίσης έχουμε καταπάτηση θεμελιωδών δικαιωμάτων όσον αφορά τις καραντίνες σε διάφορες χώρες. Οι ίδιες οι το κάνουν και σε κάποιες χώρες όπως η Κροατία. Η αντίστοιχη εξουσία μεταβιβάστηκε σε κάποιους χωρίς νομική βάση. Και ο κόσμος δεν μπορεί ούτε να δουλέψει, ούτε να πάει στο γιατρό, ούτε τίποτα. Σας ευχαριστώ. Συζητούμε με την ε, συνεχίζουμε τη συζήτηση με την Συνάδελφο κυρία Πύρμπακας. Κυρία Πρόεδρε, αξιότιμοι συνάδελφοι, θα ήθελα σήμερα ε, να μιλήσω για τη μνήμη των Ευρωπαϊκών Λαών. Πρότεινα στον πρώτο Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίου ένα ψήφισμα για την συμφιλίωση του ευρωπαϊκού λαού γύρω από μια κοινή ιστορία, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα υπερπόλη διαμερίσματα. Η ε, κληρονομιά των ανθρώπων αφρικανικής προέλευσης της κλαβιάς είναι κάτι που δεν μπορούμε να ξεχνάμε. Αυτούς εκπροσωπώ εγώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το να καταπολεμήσουμε τη σκλαβιά σημαίνει να καταπολεμούμε και, το μοντέρνα, και τη μοντέρνα σκλαβιά και να κατα, καταδικάζουμε ένα υπερφιλελεύθερο μοντέλο το οποίο οδηγεί σε πολύ καταστροφικά αποτελέσματα. Μια δικία που λαμβάνει χώρα σε μια χώρα, λαμβάνει χώρα παντού, όπως είπε πει ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ. Χρειαζόμαστε λοιπόν ένα μέλλον χωρί διακρίσει, έτσι ώστε οι ευρωπαϊκοί λαοί είναι ελεύθεροι, να είναι ίσοι το λέω στους ανθρώπους του Γουαδελούπη από τη Μαρτινίκα, την Γουιάννα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Κοκαλάρη είναι επόμενη ομιλήτρια. Κυρία Πρόεδρε, κύριε είπατε εκπρόσωπε Μπορέλα, αγαπητοί συνάδελφοι, η δημοκρατία υφίσταται επίθεση και υποχωρεί το κράτος δικαίου. Τα δε ατομικά δικαιώματα υπονομεύονται. Βλέπουμε ένα σωρό αυταρχές κυβερνήσεις να υπάρχουν όπως στη Ρωσία και στην Κίνα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να προστατεύει τα άτομα δικαιώματα. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να έχει τα κατάλληλα μέσα προς τούτο. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να θεσπίσουμε νομοθεσία που να επιβάλλει κυρώσεις για την παραβίαση δικαιωμάτων γιατί αυτοί που κάνουν κάτι τέτοιο θα πρέπει να τιμωρούνται. Θα πρέπει να προστατεύσουμε τους ακτιβιστές των ε, ε, ανθρώπινων δικαιωμάτων να ρισκαρούν τη ζωή τους. Θα πρέπει να σταματήσει στο Συμβούλιο να υπάρχει ο κανόνας της ομοφωνίας για τέτοια θέματα και έτσι η φωνή της Ένωσης να ακούγεται περισσότερο. Άρα θα πρέπει να προστατεύσουμε, θα πρέπει να λάβουμε δράση. Αν δεν το κάνουμε εμείς, ποιος θα το κάνει. Σας ευχαριστώ πολύ. Άγγελ. Συγχαρητήρια κύριε, είπατε εκπρόσωποι για τα όσα κάνετε όσον αφορά την ισότητα ανδρών γυναικών και προστασία δικαιωμάτων. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή να κάνει περισσότερα για αυτές τις ε, αξίες με ανάληψη δράσης πολιτική αλλά και με πρικοδότηση οικονομική. Πολύ σημαντικό. Θα πρέπει να σταματήσουμε ε, αυτά τα οποία ε, γίνονται ε, κατά της ισότητες των φίλων αλλά θα πρέπει κάτι να γίνει σε όλα τα διεθνή φόρα για τα δικαιώματα των ΛΟΑΔΚΙ. Θα πρέπει βέβαια να δίνουμε εμεί το καλό παράδειγμα, αλλιώ δεν έχουμε αξιοπιστία. Κομισιόν, Συμβούλιο, Κοινοβούλιο, να μην περιορίζονται σε λόγια, αλλά θα πρέπει να αναλυφθεί ταχαίω δράση, γιατί ε, η κατάσταση έχει χειροτερέψει για τα δικαιώματα των ΛΟΑΔ και σε πολλά κράτη-μέλη. Στην Πολωνία, επίση, υπάρχει νομοθεσία, διακρίση στην Ουγγαρία και επομένως θα πρέπει η Επιτροπή και το Συμβούλιο να λάβουν τη δράση, να έχουμε συνέπεια, έτσι θα έχουμε την αξιοπιστία ε, όταν θέλουμε να υπερασπιστούμε τα ανθρώπινα δικαιώματα σε όλο τον κόσμο. Ο κύριος Αντιπρόεδρος Καστάλντο, παρακαλώ. Κύριος Καστάλντο, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Ακριβώ ε, αυτό, όπω το είπατε, κύριε Πάτε, για αυτή την έκθεση, ότι η πανδημία άλλαξε άπαξ και διαπαντό στον κόσμο, την κοινωνία μας ε, ήταν μια εμπειρία. Ε, τώρα μας οδήγησε σε περισσότερη συνέστηση, σε ανθρωπιά, όμως πολλές φορές σε πολλά μέρη του κόσμου ε, η πανδημία χρησιμοποιήθηκε για καταστολή, για καταπίεση, για λογοκρισία. Θα πρέπει να είμαστε περήφανοι γιατί δεν διστάζουμε να διατρανώσουμε αυτές μας τις αξίες ε, και αυτό και προς τους εταίρους μας πολιτικούς, εμπορικούς θα πρέπει να συνεχίσουμε ε, έτσι να είμαστε ο φάρος μέσα στο σκοτάδι υπέρ των δικαιωμάτων επίσης θα πρέπει να ε, είμαστε υπέρ της πολυμερούς πολιτικής και θα πρέπει να κάνουμε κάτι για την επίθεση των δικαιώματα που γίνεται ακόμα και από τις είπα. Άρα θα πρέπει να υιοθετηθεί σύντομα ένα σύστημα κυρώσεων για παραβιάσματα των δικαιωμάτων σε όλο τον κόσμο. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Κέλλην, επόμενος ομιλητής. Καλημέρα. Καλωσορίζω αυτήν την έκθεση. Νομίζω ότι έχει επιτυχθεί έτσι ε, μια ηγετική ε, πυγμή. Θέλω να ευχαριστώ τον κύριο Γκίλμορ που συνεργάζεται με τα ε, Ηνωμένα Έθνη από πέρυσι. Βλέπουμε στις συζητήσεις ε, και στην Ιρλανδία και στο Κοινοβούλιο εδώ ότι θα πρέπει να υπερασπιστούμε αυτούς που κινδυνεύουν τους δημοσιογράφους ε, αλλά και τους απλούς ανθρώπους ε, αυτά που, που πρέπει να υποστούν οι γυναίκες σε κάποιες χώρες ε, η καταστολή στην Κίνα για όλους τους ανθρώπους πρέπει να είμαστε εκεί διότι συχνά είμαστε η μόνη ισχυρή φωνή που έχουν αυτοί οι άνθρωποι. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Ζωρίνιο είναι ο επόμενος. Η έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία που εξετάζουμε σήμερα ε, εστιάζει ε, στις περιπτώσεις, ε, στις στρατηγικές, στη δράση, στο πολυμερές σύστημα που πρέπει να υποστηριχθεί και νομίζω ότι είναι η καλύτερη δυνατή ανταπόκριση στην οικονομική, υγειονομική, πολιτική κρίση της πανδημίας και πραγματικά θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε την αύξηση του αυταρχισμού, το κλείσιμο συνόρων, μεγαλύτερη ε, μυσαλλοδοξία. Εμείς πρέπει να δείξουμε το μονοπάτι ε, προς την πολυμερή προσέγγιση και την πράσπιση των ε, θεμελιωδών δικαιωμάτων. Κύριε, είπατε εκπρόσωπε, θα ήθελα εγώ να εστιάσω στην κατάσταση στο Κάπο Ντελγάδο της Μοζαμβίκης. Ε, ε, είναι μια περίπτωση πολύ ε, εμφανής, εμφανούς καταπάτησης ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ε, σε πάρα πολύ εύθραυστες συνθήκες ε, ε, ζουν εκεί άνθρωποι, υπάρχουν θρησκευτικά οικονομικά προβλήματα, υπάρχει οι νέες γεωτρετικές δραστηριότητες και Πρέπει εμείς να τα έχουμε όλα αυτά υπόψη, πρέπει να ε, έχουμε ευρωπαϊκή ηγεσία, πρωταγωνιστικό ρόλο. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Λόπεθ έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, κύριε είπατε εκπρόσωπο, θέλω να σας ευχαριστήσω και για την έκθεση και για το έργο σας. Για μας ε, η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον κόσμο δεν είναι μόνο ανησυχητική, είναι και ένα σημάδι ε, υποβάθμισης, επιδίνωσης όπως βλέπουμε από τις γενικές τάσεις ε, και σε ό,τι αφορά το πολυμερή σύστημα και τους μηχανισμούς προστασίας ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αμφισβητείται το διεθνές δίκαιο, το ανθρωπιστικό δίκαιο και κάθε φορά βλέπουμε ε, να εφαρμόζονται κάποιοι κυβερνώντες που στο όνομα υποτίθεται της δημοκρατίας παραβιάζουν τα δικαιώματα αυτών που τους εξέλεξαν. Γίνεται λόγος ε, για κάποιες ομάδες ε, ε, συστηματική παραβίαση των δικαιωμάτων των παιδιών, των γυναικών, των ευάλωτων, ευπαθών ε, πληθυσμών και των μεταναστών, ακόμη και στα σύνορά μα. Εγώ όμω θέλω να αναφερθώ στη Λατινική Αμερική. Όλο και περισσότερο, όλο και πιο ανισχυτικό είναι το φαινόμενο ε, δολοφονιών ηγετών των αυτοχθόνων, περιβαλλοντικών υπερασπιστών και διαφόρων άλλων που αγωνίζονται στο πλαίσιο τη κοινωνία των πολιτών και εξαφανίσει. Όλα αυτά είναι πολύ ενσχετικά και πρέπει να γνωριστούμε. Ευχαριστώ πολύ ο κύριο ε, Βίλαντ. Ευχαριστώ πολύ. Προχωρούμε λοιπόν ε, στην κατάσταση στη Λευκορωσία, λέει ο πρόεδρο <laughs> κατά λάθο. ο κύριο Χριστοφόρης, τώρα για ένα λεπτό. Από αυτό το βήμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καταγγέλλω την Τουρκία για τι συνεχιζόμενε και κλιμακούμενε απειλέ, εκβιασμού και επιθέσει σε βάρο τη Κύπρου και τη Ελλάδο, δύο χωρών μέλων τη Ευρωπαϊκή Ένωση και ταυτόχρονα προειδοποιώ την ευρωπαϊκή ένωση ότι αν δεν λάβει σήμερα άμεσα και αποφασιστικά μέτρα για να αναχαιτήσει την τουρκική επιθετικότητα αύριο θα είναι πολύ αργά και θα είναι ανεξέλεκτες οι συνέπειες. εάν όλοι μας μέσα στην ευρωπαϊκή ένωση πιστεύουμε ότι η θεμελιωδική αξία της είναι η αλληλεγγύη ένα έχουμε να πράξουμε να καλέσουμε τις χώρες μέλη της ευρωπαϊκής ένωσης να διαθέσουν τις ναυτικές τους δυνάμεις στην ευρωπαϊκή ένωση για να μπορέσει να προασπιστεί και να διαφυλάξει τα εξωτερικά της σύνορα που είναι τα σύνορα της κύπρου και της ελλάδας είμαι περήφανος και ευτυχής γιατί ανήκω στο ευρωπαϊκό λαϊκό κόμμα που υιοθετεί αυτή τη θέση και στηρίζει ανεπιφύλακτα τις θέσεις υπέρ της κύπρου και της ελλάδας ταυτόχρονα υιοθετώ τη θέση του ηγέτη του ευρωπαϊκού λαϊκού κόμματο Μάφρε Βέμπερ ότι αν η Τουρκία συνεχίσει σε αυτή τη γραμμή πρέπει να ανασταλεί την τελωνιακή τη Ένωση. Όμω και εμεί ω Ευρωκοινοβούλιο οφείλουμε να περικόψουμε τα ενταξιακά κονδύλια τη Τουρκία και να αφαιρέσουμε την Τουρκία από το πολιετέ δημοσιονομικό πλαίσιο γιατί μόνο έτσι η Τουρκία μπορεί να κατανοήσει το πρόβλημα που δημιουργεί στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Ισχυρή Ευρωπαϊκή Ένωση, δυνατή με αλληλεγγύη, σημαίνει Ευρωπαϊκή σας ευχαριστώ πολύ κύριε Χριστοφόρου. Με συγχωρείτε, λέει ο κύριος ε, Βίλαντ, έκανα λάθος στην αρχή. Είπα ότι θα συστήσουμε την κατάσταση στη Λευκορωσία, ενώ βεβαίως συζητούμε ε, την κατάσταση της στην Ανατολική και τον ε, αρνητικό ρόλο της Τουρκίας. Θα... Ελπίζω να μην ενοχλήθηκε ο κύριος Χριστοφόρο από το λάθος που έκανα. Ο κύριος Σάντσεφ Αμόρ έχει τώρα το λόγο. Κύριε Μπορέλ, είναι περίπλοκη η σχέση με την Τουρκία αλλά είναι μία σχέση έτσι ε, γίνεται μια προσπάθεια ε, ε, να συνδέουμε πράγματα τα οποία δεν έχουν σχέση μεταξύ τους στην Τουρκία έχουμε προσφέρει ό,τι μπορούμε να προσφέρουμε ε, μέχρι και υποψηφιότητα είναι μια χώρα υποψήφια εντάξει αλλά θα πρέπει σιγά σιγά να ευθυγραμμίζεται με τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η κατάσταση εκεί δεν είναι καλή, διότι υπάρχει έλλειψη εμπιστοσύνη. και αυτό επηρεάζει το σύνολο της σχέσης. Έχει βεβαίως επιδεινωθεί η κατάσταση από τα ανθρώπινα δικαιώματα και για την απελευθέρωση των θεωρήσεων. Η Τουρκία δεν έχει ε, σεβαστεί τις δεσμεύσεις της. Ε, σε ό,τι αφορά τη μετανάστευση, ε, τα πράγματα επίσης είναι πολύ κακά. Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα και την Κύπρο, εμείς δεν μπορούμε να λέμε ότι είμαστε αλληλέγγυοι με την Ελλάδα και την Κύπρο. Είμαστε η Ελλάδα και η Κύπρος. Δεν είμαστε κάποιοι ενδιάμεσοι δημοσιολογητέ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αξιότιμη είπατε εκπρόσωπε, έχω ένα ερώτημα για σας αναρωτιέμαι κατά πόσο ο πρόεδρος Ερντογάν θέλει να προσχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δείτε τις τελευταίες δράσεις της Τουρκίας, τις ενέργειές της. Πάνε κατά όλων των αξιών και συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι δραστηριότητε στα διεθνή ύδατα, οι παράνομες, παραβίαση του εμπάργου όπλων των Ηνωμένων Εθνών, ο εκφοβισμός ε, χωρών μελών της Ένωσης και του ΝΑΤΟΥ, ε, το σύστημα, τα, τα συστήματα τα πυραυλικά τα ρώσικα τα οποία αγόρασαν ε, η καταπίεση του λαού των δημοσιογράφων των συνδικαλιστών και βεβαίως ε, η συνεχής, ο συνεχής εκβιασμός που θα ανοίξουν τις πόρτες προς την Ευρώπη και η λίστα δεν τελειώνει ποτέ Κύριε είπατε εκπρόσωπε, είναι ένα αστείο η διαδικασία προσχώρησης της Τουρκίας. Βεβαίως και η Τουρκία είναι στρατηγικός εταίρος και για την Ευρώπη και για το ΝΑΤΟ και είναι και γείτονα, βεβαίω. Και βεβαίω πρέπει να έχουμε μια ισχυρή σχέση με την Τουρκία. Όμω εξακολουθεί να απομακρύνεται η Τουρκία όλο και περισσότερο. Αυτό το κοινοβούλιο είναι σαφές. Αυτή η αυταρχική Τουρκία δεν μπορεί να προσχωρήσει στην Ένωση. Δεν μπορεί να ενταχθεί. Σας ευχαριστώ για τις προσπάθειες που κάνετε να συνεχίσετε το διάλογο με την Τουρκία. Σας ρωτάω όμως, σας ζητάω μάλλον, να είστε σαφείς, να είστε ειλικρινείς απέναντι στην Τουρκία. Δεν μπορεί να υπάρξει αναβάθμιση της σχέσης με τη χώρα αυτή όσο οι ενέργειές της, οι δράσεις της δεν αλλάζουν και όσο η Τουρκία δεν δείχνει πραγματική ετοιμότητα για σοβαρές μεταρρυθμίσεις. Σας ευχαριστώ και καλή τύχη. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Φωτμάνς. Μαριάννη, ένα λεπτό. Monsieur le Président, merci. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε, είπατε εκπρόσωπε, μέχρι πότε πρόκειται να, αναχθείτε αυτή την ε, κατάσταση. Είναι στην πόρτα μας, μπροστά μας, είναι ένας εχθρός. Ο Χαλίφης Ορντογάν, ε, έχουμε τώρα και τις ε, επιθέσεις του. Επομένως, είναι διπλό στοίχημα. Έχουμε όλους τους μουσουλμάνους εδώ που ε, είναι κάτω από αυτή την σημεία και έχουμε και αυτά που γίνονται στην Μεσόγεια. Αυστριακοί, Ούγγροι, Ελλάδες, Έλληνες, νόμοι Κύπροι, Ρώσοι και άλλοι Ευρωπαίοι ε, θα πρέπει να αντιμετωπίσουν αυτή την διπλή απειλή από τότε που έπεσε η Κωνσταντινούπολη και ε, βλέπουμε ότι πρόκειται για μια ιστορική αποστολή αλλά όταν η Αλβανία και το Κόσοβο γίνονται προτεκτοράτα τουρκικά κλείνουμε τα μάτια και από την άλλη τι γίνεται επιταχύνουμε τη διαδικασία της ένταξης στην Λιβύη αναπαράγουμε τα ίδια ασφάλματα ξανά τα ίδια ό,τι κάναμε στη Συρία και βλέπουμε αυτές τις στρατοχωροφυλακές που ε, πληρώνται από τους Τούρκους το, το βλέπουμε σαν να μην σημαίνει τίποτα. Έγινε επίση πράξη πολέμου ει βάρο της Γαλλίας από την Τουρκία στην ε, θάλασσα. Τι γίνεται, καμία αντίδραση, καμία ελεγγύη. Κύριε Πατή εκπρόσωπο, μέχρι πότε θα τα ανεχόμαστε όλα αυτά, μέχρι πότε θα συνεχίσουμε αυτή την ε, ε, πορεία τη Τουρκία Τουρκίας για την ένταξή τη που δεν συμμερίζεται καμία από τι αξίε μα. Θα πρέπει να είναι αποφασιστική η Ευρώπη και αν θέλουμε την ε, ειρήνη, θέλουμε να προσθέτουμε τα σύνορά μας, να σταματήσουμε να μας ελέγχει η Τουρκία και άρα να είμαστε αποφασιστικοί. Και οπότε προσέξτε ε, να μην μείνετε στην ιστορία ως ε, κάποιος πάρα πολύ αδύναμος. Η κυρία Στρίκη για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ. Να ευχαριστήσω και τον κύριο ε, Μπορέλ. Δίνεται η εντύπωση με τον τίτλο ότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε ε, ένα κακό ε, μόνο παράγοντα. Είναι απλό το αφήγημα, αλλά δεν μας οδηγεί πουθενά. Η κατάσταση στα σύνορά μας είναι άκρος πολύπλοκη και το πιο ανησυχητικό είναι η έλλειψη επιρροής εκ μέρου μας και στη Συρία και στη Λιβύη. Και αυτό νομίζω ότι πρέπει να αναστραφεί, στραφή. Αλλά θα αποκτήσουμε περισσότερη επιρροή αν υιοθετήσουμε περιφερειακή συνολική προσέγγιση ε, με του ε, Λίβιου. Βλέπουμε ότι υπάρχουν πολλά κράτη που προσπαθούν να επέμβουν ε, γιατί ουσιαστικά αγωνίζονται η μία χώρα για τα δικά τη συμφέροντα. Θέλουν λοιπόν τη δική μα υποστήριξη για τη δημιουργία ενό κράτου όπου η δημοκρατία, το κράτο δικαίου, η λογοδοσία θα υπερτερούν, θα κυριαρχούν. Οι απειλέ ασφαλεία θα παραμείνουν όσο η Λιβύη είναι, είναι ένα αποτυχημένο κράτο. Η Τουρκία είναι ναι, ένα από τα κράτη τα οποία παρεμβαίνουν για τα δικά τη συμφέροντα. Το ίδιο κάνει όμω και η Ρωσία, η Γαλλία, η Ιταλία και άλλε χώρε. Η συμμόρφωση με τη διαδικασία του Βερολίνου είναι άκρο ε, σημαντική και είναι απογοητευτικό το γεγονό ότι ακόμη και κράτη-μέλη τη Ένωση δεν σέβονται πάντοτε την συμφωνία αυτή. Γι' αυτό λοιπόν ε, Ζητώ από τον είπα το εκπρόσωπο να μας πει ποιες δυνατότητες βλέπει για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και διεύνηση του πεδίου της επιχείρησης Ειρήνη παρά ε, το μπλοκάρισμα από τη Ρουσία στο Συμβουλίο Ασφαλείας. Πέραν αυτού, νομίζω ότι θα πρέπει να επενδύσουμε περισσότερο στην περιφερειακή σταθερότητα και αυτό ξεκινά με την πιο κοντινή σε εμά περιοχή που είναι η Κύπρος. Πρέπει να βρούμε μια λύση ε, στο Κυπριακό. Είναι κάτι το οποίο έχουμε παραμελήσει εδώ και καιρό, αλλά και στη Βορειοαφρική, ε, οι γειτονικέ χώρε Λιβύης πρέπει να συμμετέχουν. Αυτό θα οδηγήσει στην εξέβρεση πιο βιώσιμης λύσης. Συμφωνώ με τον κύριο Μπορέλ πως παρά ε, το πολύ κακό ιστορικό ε, επιδόσεων της Τουρκίας έχουμε ε, κοινό συμφέρον, κοινό ενδιαφέρον και απέναντι στην ευρύτερη περιοχή και δεν θα πρέπει να παραμείνουμε στο δινεκές, σε αυτό το αδιέξοδο και να μην έχουμε καμία συνεργασία ή να μείνουμε σε αυτή την κοινή δήλωση του ΚΕΑΣΟΠΗΚΙΣ Εγώ θεωρώ ότι ναι, πρέπει να έχουμε στρατηγική, όχι όμως μόνο για τους λόγους ασφαλείας Σομαλίας αλλά και για την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Στρίκ. Για 1,5 λεπτό κυρία Κάνκο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Επιθετικότητα στην Ανατολική Μεσόγειο. Επιθετικότητα απέναντι στην Κύπρο. Αγοράζει τα S400 από την Ρωσία. Αντιμάχεται το γαλλικό πολεμικό ναυτικό. Εκβιάζει την Ευρώπη με του μετανάστε. Εάν δεν υποστηρίξουμε τη δράση του στη Συρία. Αγαπητοί συνάδελφοι, πρέπει να ρωτήσω, με τέτοιου φίλου, τι να του κάνει στου εχθρού. Οι τελευταίοι μήνε δείχνουν ότι η Τουρκία υπό την Ερντογάν δεν μπορεί να είναι ένας σύμμαχος αξιόπιστος στην Ευρώπη. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να έχουμε αυταπάτες την Τρίτη και, και την Τετάρτη συνεχίζουμε εμείς να λέμε ότι η Ήπειρός μας βασίζεται στις δημοκρατικές αξίες. Η συμφωνία με την Τουρκία όμως δεν βασίζεται στην πραγματικότητα. Πρέπει να αλλάξει η σχέση με την Τουρκία. Να έχουμε μια εμπορική ενδεχομένω συμφωνία, αλλά δεν μπορεί να μας ταγαθεί. Οι αξίες μας, τα συμφέροντά μας δεν είναι κοινά, αποκλίνουν οι φίλοι δεν συμπεριφέρονται όπως συμπεριφέρεται η Τουρκία. Εάν δεν μπορούμε να είμαστε φίλοι τουλάχιστον, ας έχουμε τότε μια σχέση αμυγός εμπορική. Θα πρέπει να βελτιώσει οπωσδήποτε την συμπεριφορά της Τουρκία ως γείτονος χώρα. Ευχαριστώ. Ε- Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Κάνκο. Ένα λεπτό ο κύριος Γεωργίου. Ο κύριος Γεωργίου. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Μπορέλ, στις μέρες μας η Ανατολική Μεσόγειος φλέγεται χώρες διαλύονται και άνθρωποι σκοτώνονται για να γίνει το ξαναμοίρασμα εδαφών και πλούτου. Πρωταγωνιστή σε αυτήν την προσπάθεια με έναν πειρατικό τρόπο η Τουρκία για να γίνει ηγεμόνα τη περιοχή. Κατέχει ήδη παράνομα τη μισή Κύπρο, τώρα επεμβαίνει στη Συρία, στη Λιβύη, στο Ιράκ, στη Σομαλία. Η ε, ε, απειλή επιπλέον την Ελλάδα και τρυπά με παράνομο τρόπο στην Κυπριακή ΑΟΣ. Η Ευρώπη τη προτείνει διάλογο. Να γίνει, κύριε Μπορέλ, ο διάλογο, αλλά να καθοριστούν με αξιοπρέπεια τα όρια το πλαίσιο και το διακύβευμα αυτού του διαλόγου. πώ απαντά η τουρκία; απαντά με απειλέ εργαλειοποιεί το μεταναστευτικό και ξανααπειλεί ότι θα εξαπολύσει νέα κύματα προσφύγων. η ευρώπη οφείλει να συνειδητοποιήσει επιτέλου ότι τώρα δεν απειλείται μόνο η κύπρος και η ελλάδα απειλείται και η αξιοπιστία της ίδιας της ευρωπαϊκής ένωσης. χωρίς χωρίς επαναλαμβάνω κυρώσεις αυστηρές και νόμιμες συνολικές λύσεις στα προβλήματα της περιοχής οι τουρκικές απειλές απειλούν να πνίξουν στο τέλος την ίδια την Ευρώπη. Η ανοχή της Ευρώπης απέναντι στο θηρίο εν τέλει μπορεί να την καταφάει. Αυτό θέλουμε. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Γεωργίου. Επόμενος είναι ο συνάδελφος κύριος Μακάλιστερ. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι η πρόσφατη κλιμάκωση από την Τουρκία στην Ανατολική Μεσόγειο και η παραβίαση της ε, χωρικής ε, ακεραιότητας τη ακεραιότητας ε, της, της Ελλάδας και της Κύπρου πραγματικά είναι μεγάλες προκλήσεις για την εταιρική μας σχέση. Θα πρέπει να καταστήσουμε σαφές ότι οι τουρκικές δραστηριότητες όπως οι παράνομες γεωτρήσεις στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κύπρου, οι υπερπτήσεις πάνω από ελληνικά νησιά είναι απαράδεκτε τις ενέργειες. Θα πρέπει να πάρει σημαντικά ε, μέτρα η Τουρκία για να αποκλιμακώσει αυτή τη συμπεριφορά. Θέλω να ευχαριστήσω τον είπα το εκπρόσωπο τον Ζωζέπ Μπορέλ που πήρε την πρωτοβουλία να ξαναξεκινήσει διάλογο με την Τουρκία. Πράγματι, και είπατε εκπρόσωπε, πρέπει κατεπηγόντως μάλιστα να μιλήσουμε, να συνομιλήσουμε αλλά επί τη βάση ε, στεναρών αρχών και, ε, πλήρη, και πλήρως ενωμένη ως Ευρώπη των 27. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ ο Πρόεδρος. Ε, επόμενος για ένα λεπτό είναι ο κύριος Πίτσουλα. Thank you, Mr. President. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε είπατε εκπρόσωπε. Επανειλημμένα έχουμε επικρίνει την Τουρκία για τις γεωτρήσεις στην Κύπρο, στην ΑΟΣ της Κύπρου. Προκαλεί εντάσεις στο Αιγαίο, έχει εμπλακεί στην Λιβύη. Τελικά αποφάσισε το Συμβούλιο ότι τα περιοριστικά μέτρα θα πρέπει να ισχύσουν για την ε, Τουρκία. Οι σοσιαλδημοκράτες συμφωνούμε. Υπάρχουν πάρα πολλά γκρεμή ζητήματα. Έχουμε τις διεκδικήσεις της Τουρκίας κατά θάλασσα και όσον αφορά τον ενέργειο χώρο. Έχουμε επιδείνωση στη σχέση Ελλάδας-Τουρκίας. Επίσης, η Τουρκία συνεχώς έχει εμπλακεί στα εσωτερικά της Λιβύης, παραβιάζει το εμπάργο, ε, δυναμητίζει τις προσπάθειες ε, ξεύρεσης λύσης του ΟΗΕ. Ε, θα πρέπει να σεβαστούν τα κερδικά δικαιώματα της Κύπρου, να μην συνεχίσουν αυτές τις παρανομίες. Αν συνεχιστούν οι παρανομίες θα πρέπει να δώσουμε μια απάντηση, να είμαστε αλληλέγγυοι με την Κύπρο και την Ελλάδα που είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πίτσουλα. 1,5 λεπτό κυρία Λουαζό. Κύριε είπατε εκπρόσωπε, είπατε πριν από μερικές μέρες ότι μεταξύ της Τουρκία και της Ευρωπαϊκής Ένωσης η κατάσταση ε, δεν είναι ιδανική. Γνωρίζω βεβαίως την χάρη της διπλωματικής γλώσσας, αλλά πρέπει να λέμε πράγματα με το όνομά τους κάποιες φορές. Ε, εδώ και πολύ καιρό το, το καθεστώ τη Τουρκία έχει γυρίσει την πλάτη στι αξίε μα, ιδιαίτερα σε επίπεδο ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πολύ συχνά η Τουρκία πλέον ε, μάχεται και τα συμφέροντά μα. Η παρουσία τη στη Συρία αποδυναμώνει την προσπάθεια που κάνει η συμμαχία κατά του Νταέ. στη Μεσόγειο κάνει γεωτρήσει παράνομες παραβιάζει το διεθνέ δίκαιο και βεβαίως ε, επιβουλεύεται την κυριαρχία της Κύπρου και της Ελλάδας. Στη Λιβύη στέλνει μισθοφόρους Σύριους, ορισμένου από αυτούς που είναι δεν σέβεται τις δεσμεύσεις ε, της διάσκεψης του Βερολίνου και αυξάνει τον κίνδυνο διχοτόμησης της χώρας. Ένα πολεμικό πλοίο της Τουρκίας επιτέθηκε ε, σε ένα γαλλικό πολεμικό πλοίο πριν από λίγες μέρες, δύο μέλη του ΝΑΤΟ ε, ενώ προσπαθούσε να παραβιάσει τους κανόνες του εμπάργου όπλων. Είναι εξαιρετικά σοβαρό αυτό. Δεν μπορεί να μείνει χωρίς συνέπειες. Ε, εδώ δεν χρειαζόμαστε πλέον ε, διπλωματικά λόγια απέναντι στην Άγκυρα, κύριε είπατε εκπρόσωπε. Αυτό που περιμένουμε από εσά είναι μία γλώσσα στεναρή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε είπατε εκπρόσωπε, από το 2002 δώσαμε στην Τουρκία πάνω από 16 δις για να μας βοηθήσουν στη διαχείριση του μεταναστευτικού και του επιτρέψαμε του Ερντογάν να μας εκβιάζει όσον αφορά τους μετανάστες στη Βαλκάνια και τώρα το ίδιο γίνεται και με την ε, Μεσόγειο. Προκαλούν οι Τούρκοι το χάος και προσιλητίζουν οι μήκυό τους στο Οθωμανική ιδεολογία ε, τον κόσμο. Ζορίζεται η Ένωση να δώσει αυτά που πρέπει στην Ιταλία αλλά τα δίνει στην Τουρκία. Αυτό είναι αυτοκτονικό να αναθέτουμε διαχείριση των συνόρων μας αυτό που θέλει να μας ε, δυναμητήσει. Το θέμα είναι ότι δεν θα πρέπει να συνεχίσουμε να προσκυνούμε τους Τούρκους. Θα πρέπει πολιτικά και οικονομικά να βοηθήσει η Ένωση Ιταλία, Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία και κυρίως την Ιταλία γιατί μόνο αυτές οι χώρες είναι οι φύλακες, οι φρουροί στη Μεσόγειο, οι φρουροί της ε, Ευρώπης. Διακόπτεται ο μιλητής. Ευχαριστώ κύριε Σόφο. Ο επόμενος είναι για ένα λεπτό ο κύριος ε, Μπέζελάγκερ. Ε, για 1,5 λεπτό ο κύριος Μπέζελάγκερ. Πρόεδρε, κύριε Μπορέλ, το είπε χθε η Καγκελάριο. Δεν θα μπορούμε να αποστρέφουμε το βλέμμα μα από όλα αυτά. Θα πρέπει κάτι να γίνει για άσυλο και μετανάστευση. Θα πρέπει επίση να αποκατασταθεί η ασφάλεια. Αλλά τι πάει να πει η ασφάλεια. Άπαξ και κλείνουν τα λιμάνια τους προς πρόσφυγες και μετανάστες οι ευρωπαϊκές χώρες. Δεν υπάρχει ασφάλεια στη Μεσόγειο. Όσο η πανδημία είναι η πρόφαση για να υπάρχουν τέτοια κέντρα κράτη στα ελληνικά νησιά, δεν υπάρχει ασφάλεια στη Μεσόγειο. Άπαξ και ε, δίνουμε χρήματα στην ε, ε, Λιβική εκτοφυλακή για να εμποδίζει τους μετανάστες δεν είναι ασφάλεια αυτό. Ασφάλεια είναι μόνο όταν ισχύσει το δίκαιο της μετανάστευσης, το θαλάσσιο δίκαιο, να επιτρέπουμε στον κόσμο να έρθει, να αποβιβαστεί. Θα πρέπει να μεταγκαστήσουμε τον κόσμο τον, να τον βγάλουμε από τα κέντρα κράτη στα ελληνικά νησιά. Κάθε μέρα κινδυνεύουν οι ζωές των αδελφών μας όπως θα έλεγαν οι δημοκράτες ε, συνάδελφοι αλλά θα πρέπει να αλλάξουμε ρότα να διδαχτούμε από τα λάθη μας και πρώτα πρώτα να φτιάξουμε ένα σύστημα ε, ασύλου ε, το οποίο να κάνει πιο εύκολη τη διαδικασία και θα πρέπει να αλλάξουμε τα στιγμή στρατηγική, να βρούμε νέους διάβλους, ναι, ναι, νέους δρόμους, ούτως ώστε ο κόσμος να μπορεί να έρθει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ κύριε Μπεζελάγκερ. 1,5 λεπτό το λόγο έχει ο κύριος Φράγκος. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Βρισκόμαστε σήμερα εδώ για να μιλήσουμε για την ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο. Μια ασφάλεια που όλοι όσοι μας ακούν γνωρίζουν πως απειλείται αποκλειστικά και μόνο από την, από την Τουρκία. Και είναι λογικό να απειλούμαστε τη στιγμή που η Τουρκία σφετερίζεται με παράνομες συμφωνίες στον ορυκτό πλούτο της Ελλάδας, διακινεί λαθρομετανάστες, παραβιάζει καθημερινά τα ελληνικά σύνορα και διακατέχεται από ένα νεοοθωμανικό επεκτατισμό και τη στιγμή που συμβαίνουν όλα αυτά όλο έκπληξη είδαμε τον κύριο μπορέλ να συζητά με τον τσαβούσογλου και λίγο πολύ να μας λέει πως η ευρωπαϊκή ένωση είναι έτοιμη να διαπραγματευτεί με την τουρκία για τον ορυκτό πλούτο της ελλάδας. μέχρι πότε η ευρωπαϊκή ένωση θα γυρίζει την πλάτη της στα μέλη της και όχι απλώς γυρίζει την πλάτη της αλλά άμεσα και έμεσα στηρίζει μια χώρα που σύμφωνα με χιλιάδες καταγγελίες τον 21ο αιώνα στρατολογεί ανήλικα παιδιά 6 και 7 χρονών και στο όνομα μιας θρησκείας τα καλεί να γίνουν μάρτυρες και να θυσιαστούν για την τουρκία. όλοι εσείς που μιλάτε για ανθρώπινα δικαιώματα τι έχετε να πείτε για αυτή την κατάσταση. κλείνοντας και για τους λόγους που σας ανέφερα η ελληνική λύση απαιτούμε να διακοπεί κάθε χρηματοδότηση από την ευρωπαϊκή ένωση προς την τουρκία και να διακοπεί κάθε διάλογος μαζί της. σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Φράγκο. Για ένα λεπτό το λόγο η κυρία Ντεμιρέλ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μπορέλ. Ναι, πράγματι η κλιμάκωση στην Μεσόγειο είναι ανησυχητικό. Η ρητορική μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων οξύνεται η κατάσταση. υπάρχει οικονομική και, και, οικονομική και ε, πολιτική ε, κρίση ε, και κοινωνική κρίση στην Τουρκία. Ε, και προσπαθούν να στρέψουν αλλού το βλέμμα οι Τούρκοι. Έχουμε τι ε, επεμβάσει στη Λιβύη. Είναι πράγματι ο Ερντογάν ε, παραβιάζει το διεθνέ δίκαιο και είμαστε ανήσυχοι κτλ. Γιατί όμω μιλάτε μαζί του, γιατί συζητάτε με Λίβιου πολεμάρχου. Μιλάμε εδώ πέρα για την επιχείρηση ειρήνη. Όμω εκεί που μιλάμε για το εμπάργκο υπάρχουν τα κρατημέλη που πουλάνε όπλα. Πρέπει να πάψουν εξαγωγέ όπλων στην Τουρκία για παράδειγμα. Αυτό θα ήταν είναι πιο αποτελεσματικό στο σύνολο τη όλη επιχειρηματολογία και συζήτηση. Το θέμα είναι μόνο το φυσικό αέριο και το πετρελαίο και το ΑΚΑΠΕ, αλλά και η Γαλλία ε, και η Ιταλία ε, συμμετέχουν και ουσιαστικά για τα δικά του ε, τα πετρελαϊκά συμφέροντα αγωνίζονται. Όλοι έξω. Ευχαριστώ πολύ κυρία Ντεμιρέλ για ένα λεπτό. Κύριο Φούρλα. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Μπορέλ, όταν επιτρέπει σε κάποιον να σου επιτίθεται να σε εκβιάζει να σε προσβάλλει και να μην αντιδρά ουσιαστικά το μόνο που πετυχαίνει είναι να δημιουργεί μια κατάσταση η οποία συνεχώ βγαίνει εκτό ελέγχου και μια χώρα η οποία συνεχώ αποθρασύνεται. αυτό πάθατε αυτό πάθαμε ω ευρώπη με την τουρκία. μια χώρα η οποία είναι από ένταξη αν είναι δυνατόν μια χώρα η οποία σα ζητά να διαπραγματευτείτε μαζί τη αυτά που έχει κλέψει. και το πιο εξωφρενικό είναι ότι βρίσκει έδαφο δύο χώρε μέλη τη ευρωπαϊκή ένωση βρίσκονται υπό συνεχή απειλή από μια χώρα η οποία κατέχει ευρωπαϊκό έδαφο μπήκε παράνομα σε ευρωπαϊκά ύδατα για γεωτρήσει μια χώρα η οποία επιτέθηκε σε γειτονικέ χώρε τάχα για να φέρει την ειρήνη και δεν έχει φύγει ποτέ. δεν θέλουμε να μα πείτε ότι έχουμε δίκιο ξέρουμε ότι έχουμε δίκιο. θέλουμε να μα πείτε το τι θα πράξετε για να μα υποστηρίξετε έμπρακτα ουσιαστικά και όχι με λόγια πώς θα διασώσετε έστω και την στάτη την αξιοπρέπεια της ευρωπαϊκής ένωσης η οποία φέρθηκε να εκβιάζεται από τον κύριο ερντογάν. είναι η ώρα να υπερισχύσουν επιτέλους οι αρχές και οι αξίες της ευρωπαϊκής ένωσης και όχι τα συμφέροντα. ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ κύριε Ε, ο κύριος Ανδρουλάκης έχει το λόγο για ένα λεπτό. Ένα μεγάλο τμήμα του πολιτικού προσωπικού της Τουρκίας επενδύει στον εθνικισμό και την ένταση ο κύριος ερντογάν με τη στρατηγική του ανοίγει ζητήματα που είχαν κλείσει 100 χρόνια πριν με τη συνθήκη της λοζάνης. ο επικίνδυνος αναθεωρητισμός του ακουμπάει την ελλάδα την ανατολική μεσόγειο την λιβύη και τη συρία και βέβαια πρόσφατα με τη μεγάλη του πρόκληση δήλωσε ότι θέλει να μετατρέψει την αγία σοφία σε τζαμί προκαλώντας τους χριστιανούς όλου του κόσμου. σε αυτή την κλιμάκωση η απάντηση δεν μπορεί να είναι μόνο λόγια αλλά ένα ολοκληρωμένο σχέδιο. Και βέβαια το σχέδιο αυτό θα περιέχει εμπάργκο όπλων και όχι να μην έχουμε την επιχείρηση Ειρήνη, αλλά αυτοί που μεταφέρουν τα όπλα στην Λιβύη να είναι οι ίδιοι οι Τούρκοι. Και βέβαια κυρώσει όσου εμπλέκονται στι παράνομε ενέργειε τη Κυπριακή ΑΟΣ και βέβαια εάν συνεχίσει αυτά, αυτές τις προκλήσεις της Τουρκίας τον ξαφνικό θάνατο της Τελωνιακής Ένωσης. Διότι η οικονομική εξάρτηση της Τουρκίας είναι μεγαλύτερη από ότι η Ευρώπη έχει ανάγκη την Τουρκία. Τέλο, εμεί θέλουμε ειρήνη και ευημερία στην ευρύτερη περιοχή. Αλλά το Συμβούλιο επιλέξει την ανοχή, το κόστος για του Ευρωπαϊκού λαούς θα είναι. Σας ευχαριστώ. Κυρία Ζαχαροπούλου, τα έχει μπερδέψει ο Πρόεδρο Ριβιέρ επόμενο. Κύριε, είπατε εκπρόσωπε στη Συρία. Στη Συρία, στη Λιβύη και εδώ και πολύ καιρό τα κάνει αυτά η Τουρκία στην Κύπρο και στην Ελλάδα και πολλές φορές λέμε ότι αυτή η συμπεριφορά της Τουρκίας είναι κάτι το μακρινό, είναι ένα πρόβλημα της Μεσογείου. Αντίθετα, όλους μας θίγει αυτές οι τουρκικές παρεμβάσεις. Είναι ένας κίνδυνος, είναι γεωπολιτικό πρόβλημα και καταπατά το διεθνές δίκαιο, το δίκαιο της θάλασσας. Η Ευρώπη παρατηρεί, δεν αναλαμβάνει δράση. Εδώ μπροστά στο, στο σπίτι μας βλέπουμε μια συριοποίηση, ε, ανθρωπιστική τραγωδία, ε, νέα κύματα μεταναστευτικά και ε, έξαρση της τρομοκρατίας. Είμαστε διηρημένοι. Για άλλη μια φορά εκμεταλλεύεται την αδυναμία μας, την αδρανιά μας ο πρόεδρος Ερντογάν. Δεν θα πρέπει να αφήνουμε τα ενία της Μέσης Ανατολής και της Μεσογείου. Ευχαριστώ κυρία Ζάχαροπούλου και τώρα είναι ο κύριος Ριβιέρ. Για τρίτη φορά ε, επίθεση σε, γαλλικό πλοίο από τους Τούρκους. Σταματήσαμε τη συμμετοχή στην μια επιχείρηση του ΝΑΤΟ ε, ε ως Γαλλία, αλλά τίποτε άλλο, τίποτα περισσότερο. Παράνομες γεωτρήσεις, Εκβιασμό με του μετανάστες που χρησιμοποιείται ω μέσο πίεσης, ε, ουσιαστική σύμπλευση με τον τζιχαντισμό στην Τουρκία, στη Συρία, ε, σφαγή των Κούρδων που είναι σύμμαχοί μα στη μάχη αυτή. Η πλειοψηφία σα ε, εξακολουθεί να ε, διαπραγματεύεται κατάξει της Τουρκίας, να δίνει δισεκατομμύρια στους Τούρκους. Κύριε Πίτροπε, το είπατε κι εσεί. Μόνο η Κύπρο, η Ελλάδα και η Γαλλία είναι αυτέ που να περάσουν τον εαυτό του. Εγώ ήμουν στα σύνορα Ελλάδα-Τουρκία. Είδα τον ελληνικό στρατό να φυλάσει τα σύνορα τη Ευρώπη μόνη. Ήρθε η στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση, στο Κοινοβούλιο, να βάλει τέρμα στην ενταξιακή διαπραγμάτευση τη ε, ε Τουρκία για ένταξη στην Ευρώπη. Ευχαριστώ πολύ κύριε Ριβιέρ. Τζαμπάσκι για μισή λεπτό. Ευχαριστώ, λέει ο κύριο Τζαμπάσκι. Αγαπητέ κύριε, είπατε εκπρόσωποι, τι άλλο, τι άλλο θα πρέπει να συμβεί ούτω ώστε να κατανοήσουμε τις πολιτικές του Ερντογάν. Είδατε, πολεμάει τους Κούρδους μέσα στην Τουρκία, στη Λιβύη, στην ε, Συρία, προσπαθεί να καταλάβει την Μεσόγειο. Σήμερα ε, λένε οι τουρκικές εφημερίδες ότι ελήφθη ήδη η απόφαση να γίνει τζαμί η Αγία Σοφία. Σας υπενθυμίζω ότι πρόκειται για την μητέρα όλων των ναών. Μα τι άλλο θα πρέπει να κάνει ούτως ώστε για να μπορέσετε να διακρίνετε την αλήθεια πίσω από τα προσχήματα, πίσω από την βιτρίνα. Να καταλάβετε ότι η Τουρκία δεν είναι ευρωπαϊκή χώρα και ούτε ποτέ θα γίνει ευρωπαϊκή χώρα από καμία άποψη πολιτιστική, πολιτική από καμία άποψη μα γιατί συνεχίζουμε αυτό το καραγκιοσιλίκι της μελλοντικής της ένταξης. Γιατί δίνουμε χαρτζηλίκη στην Τουρκία για να χρηματοδοτούνται οι πολιτικές αυτές. Κύριε, είπατε εκπρόσωπε, είναι ξεκάθαρο, θα πρέπει οι διαπραγματεύσεις των νωρίτερο να σταματήσουν. Ευχαριστώ κύριε Τσαμπάσκι. Για ένα λεπτό έχει το λόγο ο κύριος Μογέλ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Για πολύ καιρό ακόμη θα μείνουμε αδρανείς πάνω στις ε, επαναλαμβανόμενες προκλήσεις της και στη Μεσόγειο, επιθετική στάση μιας ε, τουρκικής ε, φρεγάτας ε, σε βάρος ενός σκάφους του γαλλικού ναυτικού που δρούσε όμως από την αιγίδα του ΝΑΤΟ. Είναι ένα ανησυχητικό επεισόδιο αλλά δεν είδαμε και τόσο πολλές αντιδράσεις ενώ δείχνει την ασυνέπεια του ευρωπαϊκού πυλών αν θέλετε της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας και αυτοί που μιλάνε τελικά για εγκεφαλικό θάνατο του ΝΑΤΟ θα βγουν δικαιωμένοι. Λέμε και ξαναλέμε ότι θέλουμε μια Ευρώπη ανεξάρτητη ε, αλλά τελικά εμείς είμαστε ε, αυτοί που αδρανώντας επιτρέψαμε στην Τουρκία να, ε, να αναζητήσει επιρροή σε άλλες περιοχές. Δείτε τι κάναμε με τη Συρία. Δεν μπορέσαμε να βοηθήσουμε τους Κούρδους συμμάχους. Δείτε σήμερα τι γίνεται στη Λιβύη. Ναι, ο κύριος Ερτογάν πράγματι εποφελείται και εκμεταλλεύεται τις αδυναμίες μας, τους δισταγμούς μας και γι' αυτό θα πρέπει η Ευρώπη να κερδίσει το σεβασμό που της αναλογεί και αυτό το χρωστό ευχαριστούμε και στους ίδιους μας τους πολίτες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μογέλ. Για ένα λεπτό κύριο Σαλίνη. Ο κύριος Σαλίνη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητέ είπατε εκπρόσωπε. Εσείς μας χαρακτηρίσατε, μας περιγράψατε τη σχέση μας με την Τουρκία μέσα από αυτή την έκθεση και μας ε, αναφέρατε αρνητικές τάσεις. Παρακαλώ, θα πρέπει η διατύπωσή σας να είναι λιγότερο αφελής, εάν είναι δυνατόν, γιατί αυτά τα οποία γίνονται μεταξύ μόνο και της Τουρκίας δεν είναι αρνητική τάση, είναι έλλειψη σεβασμού για τους συνήθεις κανόνες θεσμικής συνεργασίας. Αυτά τα οποία γίνανε δεν έγιναν κατόπιν της ε, αίτησης, της ε, ένταξης. Απλώς αυτό το οποίο κάνανε αντικατέστησαν ε, μια νεοοθωμανική στρατηγική που είδαμε ότι εφαρμόζεται σε Αίγυπτο, την Ισία, Κύπρο, Ελλάδα, Αλγερία και Λιβύη. Δηλαδή έχει ε, έχουν υποκαταστήσει την Ευρώπη στον χώρο της Μεσογείου. Ο, ο Άλντο Μόρο, ο ηγέτης, ο χριστιανοδημοκράτης, έλεγε ότι η Ευρώπη είναι μία ήπειρος στην Μεσόγειο. Η Ευρώπη είναι η Μεσόγειος, έλεγε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Σαλίνη. Ένα λεπτό, η κυρία Ινσύρ. Μικρόφωνο. Λειτουργεί τώρα. Κύριε Πρόεδρε, η κυβέρνηση του Ερντογάν είναι μια απειλή. Απειλή για τον τουρκικό λαό, απειλή για τη Μέση Ανατολή, απειλή για την Ευρώπη. Οι δράσει τη Τουρκία, οι ενέργειε τη Τουρκία είναι ανησυχητικέ εδώ και καιρό. Οδηγούν σε κλιμάκωση στην Βόρεια Αφρική, στη Μέση Ανατολή. Και βεβαίω ε, μπορεί να έχουμε και νέε σειράξει στη Μεσόγειο. Ο Ερντογάν χτυπάει την αντιπολίτευση αλίπητα. Ε, ε, στο Κουρδιστάν οι βόμβες του Ερντογάν πέφτουν πάνω σε άμαχους. Οι παραβιάσεις ε, των χωρικών υδάτων της Ελλάδας, οι, οι γεωτρήσεις, η ε, κατοχή στην Κύπρο Όλα αυτά παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο και βλέπουμε βεβαίως ότι οι απειλές ε, της ε, Τουρκίας πάνε από τη μια χώρα της Ευρώπης στην άλλη. Ε, υπάρχει πραγματικό κυνήγι μαγισσών απέναντι σε τρεις ε, σοσιαλδημοκράτησες από τη Σουηδία παραδείγματος χάρη. Ε, κύριε Μπορέλ, είναι πολύ σημαντικό ο διάλογο, βεβαίω. Και ήταν σημαντικό ότι επισκεφτήκατε την Τουρκία την περσμένη εβδομάδα. Πόσο καιρό όμω ακόμα θα είμαστε καλοί με την Τουρκία. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριο Τσίμνιοκ έχει το λόγο για ένα λεπτό. Κύριε... Ο κύριο Τσίμνιοκ. Η ε, κρίση με την Τουρκία υπάρχει από το 2015 ε, και κανείς δεν θέλησε να πάρει τα απαραίτητα μέτρα, ιδιαίτερα στη Γερμανία και η κυρία Μέρκελ έτσι ώστε να λυθούν τα προβλήματα. Άδεια λόγια, ε, συνθήματα, δεν βοηθούν αυτά. Αυτή τη στιγμή μας ε, εκβιάζει ο Ερντογάν. Υπάρχει πόλεμο στη Συρία κατά τον Κούρτον από, από την Τουρκία. Ε, βλέπουμε τι γίνεται στα χωρικά ύδατα. Βεβαίως υπάρχει η μαφία της μετανάστευσης στην Ελλάδα όπου δεν ελέγχει μόνο τη Βαλκανική οδό Ερντογάν, αλλά η στρατιωτική του παρουσία πλέον στη Λιβύη σημαίνει ότι ελέγχει και την οδό από την κεντρική Μεσόγειο. Ο Ερντογάν λοιπόν δεν είναι λύση εδώ, είναι πρόβλημα και θα πρέπει πραγματικά να αντιδράσουμε και να του μιλήσουμε τη γλώσσα που καταλαβαίνει. Δεν μπορεί να υπάρχει καμία υποστήριξη. Πρέπει να κλείσουμε ε, τη βρύση της ενίσχυσης της οικονομικής έτσι ώστε να σταματήσουν οι εγκληματικές πράξεις του Ερντογάν. Κύριος Φιντάντσα, 1,5 λεπτό. Μέσα σε μισό αιώνα έχει αναδειθεί ως ε, δύναμη και θα γίνει πιο μεγάλη στον κόσμο. Τα ε, είπε τον Φεβρουάριο φέτος στο τουρκικό κοινοβούλιο ο, ο Σουλτάνος ε, Ερντογάν. Όλο ένα και πιο φανερό είναι αυτό. Ισλαμισμός, ε, διώξεις των Κούρδων, ε, εξορίξεις στην Κύπρο κόντρα στα συμφέροντα Γαλλίας, Γαλλίας, Κύπρο, Κύπρο, όλων και βλέπουμε ότι πιέζουν με το μεταναστευτικό πρώτα στη ελληνικά σύνορα, μετά στην Λιβύη και η Ευρώπη αδρανή συνεχίζει να πληρώνει. Τι γίνεται με τους Τούρκους ε, που διαμένουν στην ε, Ευρώπη. Πρόκειται περί επικισμού ε, αυτών και των παιδιών τους. Θα πρέπει να δούμε τι γίνεται από το Ισλάμ μέχρι, μέχρι το Σουδάν. είδαμε ότι πώς απελευθερώθηκε η Ιταλίδα Όμηρος των Ισλαμιστών με διαμεσολάβηση τουρκική η όμοιρος της Σαμπάμπ επομένως ε, η, Τουρκία δεν έχει καμία σχέση με την Ευρώπη όπως την αντιλαμβανόμαστε πώς είναι υποψήφια για ένταξη θα πρέπει να κόψουν τους δεσμούς μας με την Τουρκία Ευχαριστώ πολύ κύριε ένα λεπτό κύριος Γουόλας Η Τουρκία έχει εισβάλει στο Ιράκ. Όποτε θέλει βγαίνει στην Συρία. Παραβιάζει το εμπάργκο του ΟΗΕ στην Λιβύη. Τι γίνεται, έχει το πράσινο φως από τη ΣΥΠΑ και εμείς έχουμε υποταχθεί σε αυτό. Τι γίνεται με τις αξίες μας. Είμαστε κομπάρσι. Θα, αυτό το οποίο γίνεται είναι να πλήσονται χωρίς έλεος οι Σύριοι. Εμείς δεν κάνουμε τίποτα. Και συνεννόηση με τον Νετανιάχου, αλλά κύριε Μπορέλ, μας λέτε για αυτά τα 3,5 εκατομμύρια πρόσφυγες, μα τι μέλλον έχουν, δεν τους θέλει η Ευρώπη, θα μείνουν για πάντα στην Τουρκία. Συνεργαστείτε με την ε, Συρία αγνοήστε τις απειλές των Αμερικανών. Θα πρέπει να σταθεί στα πόδια της Συρία για να επιστρέψουν οι πρόσφυγες. Ντροπή. Ευχαριστώ κύριε Για ένα λεπτό κύριος Μάντελ έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Μας δίδαξε η πανδημία ότι θα πρέπει να είμαστε συσπηρωμένοι ε, και οι συμπολίτες μας από την Τουρκία είναι και αυτοί οι άνθρωποι όπως όλοι οι άλλοι. Η ηγεσία της Τουρκία όμως που ε, δεν συμφωνεί μαζί της οι περισσότεροι, ε, από τους Τούρκους κάνει τα, όλα, τα πάντα λάθος και αυτό που κάνει είναι να αποσταθεροποιεί την ευρύτερη περιοχή κλιμακώνει αντί να αποκλιμακώνει και αυτό ε, χρειάστηκε να έρθει η πανδημία για να το μάθουμε μάλλον όλοι. Βλέπουμε τι γίνεται με τη Λιβύη ε, πώς φέρεται σε βάρος εταίρων του ΝΑΤΟ ε, στη Μεσόγειο. Και υπάρχουν και στην ίδια την Ευρώπη αψιμαχίες που υποκινούνται από την Τουρκία. Στους ίδιους δρόμους χωρών πρωτευουσών ή πόλεων της Ένωσης. Ευρώπη δεν είναι όριμη και πρέπει να πάρουμε τα σωστά μέτρα κάποια στιγμή. Ευχαριστώ πολύ. Κύριος Μαυρίδης έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι σημαντικό σήμερα ότι συζητάμε τις παρανομίες τη Ένωση. η ευρωπη δεν ειναι οριμη και πρεπει να παρουμε τα σωστα μετρα καποια στιγμη ευχαριστω πολυ Κύριο Μαυρίδη εχει τωρα το λογο ευχαριστω κυριε προεδρε ειναι σημαντικο σημερα οτι συζηταμε τις παρανομιες της τουρκιας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ανατολική Μεσόγειο ευρύτερα. Αλλά αυτό δεν αρκεί. Κορυφαία λάθη στην ιστορία, αγαπητέ μου κύριε Μπορέλ, επαναλαμβάνονται επειδή οι έχοντες εξουσία δεν διδάσκονται από τα λάθη του παρελθόντος. να αναφέρω ένα η πολιτική του κατευνασμού απέναντι στο ναζιστικό καθεστώς τελικά το πλήρωσε αυτό το μέγιστο λάθος η ανθρωπότητα με ποταμούς αίματος γιατί δεν διδαχθήκαμε από την ιστορία και οι υποστηριχτές εκείνης της πολιτικής καταδικάστηκαν από την ιστορία. επομένως η αξιοπιστία της ευρωπαϊκής ένωσης κρίνεται στην ανατολική μεσόγειο. θα προασπιστούμε το διεθνές δίκαιο και το ευρωπαϊκό δίκαιο και τις αξίες μας ή θα συνεχίσουμε να πουλούμε όπλα στην τουρκία; καθώς μιλάμε η γερμανία πουλάει υπερσύγχρονο οπλισμό στην τουρκία τον οποίο θα χρησιμοποιήσει εναντίον των συμφερόντων της ευρωπαϊκής ένωσης. αυτή δεν είναι αξιοπιστία ούτε αξίες αγαπητέ μου κύριε borrell. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Μαυρίδη. Για ένα λεπτό το λόγο έχει η κυρία Ντονάτο. Ευχαριστώ αγαπητέ υπατή εκπρόσωπε. Τι γίνεται με αυτόν τον διάλογο με την ε, Τουρκία. Ε, ε, είσαστε ευγενικοί, είσαστε επίοικείς με ένα τέτοιο κράτος που συνέχεια παραβιάζει το διεθνές δίκαιο που ε, έχουμε 11 εκατομμύρια πρόσφυγες, 400.000 θύματα από αυτόν τον πόλεμο στον οποίο έχει εμπλακεί η Ρωσία. Έχει μισθοφόρους στη Λιβύη, παραβιάζει το εμπάρκο των όπλων. Εδώ και χρόνια δισεκατομμύρια δίνουμε στην Τουρκία από το Ταμείο της Προένταξης για να διαχειριστούν το προσφυγικό του σύρους πρόσφυγες και τώρα πάμε για περισσότερη ε, χρηματοδότηση παρά όλα αυτά τα οποία κάνουν ε, είδατε στην Ανατολική Μεσόγειο ότι γίνεται, επιθετικότητα κατά Κύπρου και Ελλάδας παραβιάζουν ανθρώπινα δικαιώματα, είναι αυταρχικό το καθεστώς, έχει λογοκρισία, καταπιέζει και τις χριστιανικές μειονότητες και την κουρδική μειονότητα ε, αδράνεια εμείς επιδεικνύουμε θα πρέπει άπαξ πρέπει να βάλουμε φρένο σε αυτές τις παραβιάσει με κυρώσεις και με πάυση πάση συνεργασία με τους νεοθωμανούς. Ευχαριστούμε. Για ένα λεπτό. Ο κύριος Μπουσαντέ Μπιγιάλμπα. Ευχαριστώ πρόεδρε. Κύριε Μπορέη, στην κρίση του περσμένου Μαρτίου, όταν χιλιάδε μετανάστε έστειλε ο Ερντογάν σύνορα με την Ευρώπη, πλέον έχουμε τις προκλήσεις απέναντι στην Κύπρο, την Ελλάδα, τη Γαλλία, αλλά και τις απειλές που ακούστηκαν όταν πήγατε εσείς στην Άγκυρα. Βλέπουμε ότι δεν υπάρχει επαρκή αποφασιστικότητα με την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν υπερασπιζόμαστε επαρκώ τι αξίε μα τι χριστιανικέ. Ε, υπήρξε μια επιστολή από όλου του βουλευτέ του Vox εσά. σα ζητήσαμε, να σταματήσετε να πληρώνετε εκατομμύρια στην Τουρκία και μα είπατε ότι τα χρήματα δεν πάνε όλα στην κυβέρνηση και ότι εσεί είστε υπέρ του να συνεχιστούν αυτέ οι πληρωμέ. Εντάξει, να συνεχίσουμε να πληρώνουμε λοιπόν 1,7 ε, τρισεκατομμύρια ευρώ ε, προς μια χώρα που δεν είναι εταίρο. Το ίδιο συμβαίνει και με το Μαγκρέμπ. Πολλέ χώρε δεν ε, συνεργάζονται μαζί μα ό,τι αφορά την, την έλεγχο τη παράνομη μετανάστευση. Συζητάμε λοιπόν να σταματήσετε αμέσω όλε τι πληρωμέ προ τρίτε χώρε που δεν συνεργάζονται σαφώ μαζί μα ό,τι αφορά τι πολιτικέ μετανάστευση. Και να μπει ένα τέλο στην διαδικασία την ενταξιακή τη Τουρκία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πουσαντεβιλιάλμπα. Ένα λεπτό κυρία Ζόφκο. Εγώ προέρχομαι από μεσογειακή χώρα και πρέπει να σας πω ότι πραγματικά το λίκνο του ευρωπαϊκού πολιτισμού παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο για την ασφάλεια και την ευημερία όλων των Ευρωπαίων πολιτών. Όταν η ασφάλεια λοιπόν στη Μεσόγειο διακυβεύεται πρέπει να τη δρούμε όλοι μαζί. Οι συμπατριώτες μας ε, οι Έλληνες, οι Κύπροι υποφέρουν από τις απειλές της Τουρκίας. Παραβιάζεται το διεθνέ δίκαιο, δημιουργούν ένταση, δημιουργούν σειράξεις. Ε, τους τελευταίους μήνες έχουμε δει συμπεριφ... Ε, παρεμφερή συμπεριφορά και σε ό,τι αφορά τη μεταναστευτική πολιτική στα ευρωπαϊκά σύνορα. Έχουμε στείλει ένα ισχυρό μήνυμα, το στείλαμε τότε, ότι εμείς ενωμένοι προστατεύουμε τα σύνορά μας. Αυτή η συμπεριφορά πρέπει να σταματήσει άμεσα. Καλό λοιπόν Βεβαίω το να ε, βρεθούν λύσεις μέσω διαλόγου διότι μέσω διαλόγου μόνο μπορούμε να αποφύγουμε περαιτέρω κλιμάκωση την οποία η ιστορία δεν θα συγχωρήσει η Μεσόγειος παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Είναι μια παγκόσμια κληρονομιά. Πρέπει να ασπαστεί τι ευρωπαϊκέ αξίε τη Τουρκία εάν θέλουμε να έχουμε ένα κοινό μέλλον. Ευχαριστούμε κύριε Ζόφκο. Ένα λεπτό σύντερ να επόμενος ομιλητής. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, να καλωσορίσω και τον κύριο είπατε εκπρόσωπο Ερντογάν με πολύ μεγάλα βήματα που μακρύνεται από τις ευρωπαϊκές αξίες ή μάλλον όχι ήταν πολύ μακριά από την αρχή και από τις ευρωπαϊκές αξίες και από τα ανθρώπινα δικαιώματα και από το διεθνές δίκαιο. Βλέπουμε ότι καθερούνται δημοκρατικά εκλεγμένοι δήμαρχοι, διώκονται ε, για πολιτικούς λόγους και κρατούν φυλακές πάρα πολλοί δημοσιογράφοι και άλλοι. Και βλέπουμε τι γίνεται όμως όπως τη Βιέννη για παράδειγμα ε, που ε, ουσιαστικά υποκινεί η Τουρκία ταραχές και και σε πόλεις της Ευρώπης. Βλέπουμε τι έκανε το τοκικό ναυτικό, πώς επιθετικά κινείται απέναντι και στην Κύπρο, στη Λιβύη και ε, παρόλα αυτά πρέπει κυρίες και κύριοι να διερωτηθούμε τελικά. Η Τουρκία μπορεί να είναι ένας εταίρος μας ε, ε, στο Συμβουλίο της Ευρώπης, στο ΝΑΤΟ. Ε, οι κυρώσεις έχουν φέρει κάτι ή πρέπει να προχωρήσουμε στη διακοπή της τελευταίας της Σύνδεσης. Ευχαριστώ πολύ κύριε Σίτερ. Μπαρντέλα είναι επόμενος για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ένα πολεμικό τουρκικό το οποίο επιτίθεται σε ένα γαλλικό πολιτικό που επιτίθεται, σε ελληνικά ελικόπτερα επιθέσεις στη Συρία, στην Τουρκία, στο Ιράκ συμμαχία με τον Άισις θέλουν να κάνουν την Αγία Σοφία τζαμί όλοι καταλαβαίνουμε την στάση του Ερντογάν και την τακτική του. Φαίνεται όμως να μην το καταλαβαίνουν οι Ευρωπαίοι θύνοντες. Ήμουν στα σύνορα με την Ελλάδα ε, πρόσφατα και είδα αυτή την επιθετικότητα του Τούρκου Σουλτάνου απέναντι στην πυρό μα, απέναντι σε μια χώρα, ε, την Ελλάδα, την οποία έχετε εγκαταλείψει απέναντι στον εκβιασμό τη Τουρκία, ε, το μεταναστευτικό. Έχετε συνθηκολογήσει. Πρέπει να μπει τέλος σε αυτό το κρυφτούλι με τον Ερντογάν. Αυτές οι επιθέσεις στα σύνορά μας, στο στρατό μας δεν είναι αποδεκτοί. Πρέπει να υπάρξουν κυρώσεις οικονομικές, να σταματήσουν όλες οι οικονομικές ενισχύσεις απέναντι στην Άγκυρα με χρήματα των Ευγάλων φορολογουμένων και των υπόλοιπων Ευρωπαίων. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και Μπαντελά. Ένα λεπτό ο κ. Μπελαμή. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Το 1935 ο Μουσταφά Κεμάλ δημιούργησε ένα μουσείο από την Αγία Σοφία και έδειξε πόσο καθολικό είναι αυτό, αυτή η κληρονομιά, πόσο οικουμενικό. Είναι σαφές το μήνυμα του Ερντογάν σήμερα, να να ανακάνει τζαμί. Αυτό που κάνει η Τουρκία, το να αλλοιώνει την ιστορία, ε, για το μικρασιατικό, για την αρμενική γενοκτονία, όλα αυτά δημιουργούν ένα προηγούμενο επικίνδυνο. Πρέπει να σταματήσουμε να αρνούμαστε την πραγματικότητα. Ο δρόμο που έχει πάρει η Τουρκία είναι ενισχυτικό, όχι μόνο για τη Μέση Ανατολή, για τον ολόκληρο τον κόσμο και για την Ευρώπη όλο ιδιαίτερο. Είχαμε τι πρόσφατε εντάσει στη Μεσόγειο, οι οποίε είναι σοβαρέ. Θέλω πραγματικά να υποστηρίξω την Ελλάδα, του Έλληνε, του Κύπριου, οι οποίοι βρίσκονται απέναντι στον εκβιασμό αυτό. Απέναντι σε αυτά, η Ευρώπη φαίνεται ανήμπορη. Και πάλι μα προτείνουν σήμερα να στείλουμε χρήματα στου Τούρκου. Χρήματα τα οποία θα μπορούσαν να πάνε στου γεωργού μα, παραδείγματο χάρη. Χρήματα τα οποία δεν ελέγχουμε πλέον. Πρέπει να σταματήσουμε να δούμε στην πραγματικότητα, να μπει τέλο στην ενταξιακή ε, διαδικασία τη Τουρκία που είναι επιστημονική φαντασία. Ευχαριστώ και τον κύριο Μπελαμή. Ένα λεπτό, κύριο Μαγιορίνο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Στην Τουρκία του Ερντογάν έχουμε μία άνοδο του αυταρχισμού Είδα κατήργησαν τους ε, ε, εκλεγμένους δήμαρχους και καταστέλλεται η κοινωνία κόντρα στις αξίες της δικιάς μας. Δεν είναι πρόβλημα ο Ερντογάν μόνο για αυτό που κάνει στην Τουρκία αλλά και για το τι ε, προκαλεί εκτός των ε, συνόντων στη Λιβύη, στη Συρία, τι κάνει κατά των ε, Τούρκων. Είδατε πώς εκμεταλλεύεται τους πρόσφυγες και έναντι των ευρωπαϊκών χωρών. Άρα, ενώπιον αυτών των γεγονότων, πού είναι η δική μας ευθύνη. Φυσικά και πρέπει να τον καταδικάσουμε και να συνεχίζουμε να το κάνουμε και κατηγορηματικά. Όμως να γνωρίζουμε ότι εκμεταλλεύτηκε καταστάσεις ο Ερντογάν, εκμεταλλεύτηκε τις δικέ μας στρατηγικές επιλογές ε, και ενεργεί έτσι στην ε, Μεσόγειο γιατί ε, έτσι καταπατήθηκε τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ευχαριστώ κύριε Μαγιορίνο. Για ένα λεπτό το λόγο ο κύριος Μημαράκης. Μικρό, Μικρόφωνο, παρακαλούμε. Όλοι θέλουμε καλέ σχέσει με την Τουρκία υπό την προϋπόθεση ότι αυτή θα μας σέβεται, θα σέβεται τους κανόνες του διεθνού δικαίου, δεν θα τους καταπατά όπως προκλητικότητα συμπεριφέρεται τελευταία. Αλλιώς δεν έχει νόημα αυτός ο διάλογος γιατί αυτή η χαλαρή συμπεριφορά δίνει στον Ερντογάν χώρο να προκαλεί, να εκβιάζει, να αυθαιρετεί μέχρι και την αγία σοφία. το παγκόσμιο αυτό μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς θέλει να μετατρέψει σε τζαμί. μας προκαλεί διότι δεν είναι στρατιωτική επιχείρηση αυτό είναι χτύπημα στον πολιτισμό μας είναι χτύπημα στον χριστιανισμό και για μας τους έλληνες είναι χτύπημα στην καρδιά μας γι' αυτό εξεπλάγημεν όλοι από τις εικόνες που είδε ο πλανήτης στο πλαίσιο της επίσκεψής σας κύριε μπορέλ στην τουρκία αφού αρνήθηκε να σας συναντήσει ο ερντογάν ταπεινώνοντας για άλλη μια φορά την ευρωπαϊκή ένωση στο πρόσωπό σας όπως είχε κάνει και στην κοινή συνέντευξη τύπου με τον κύριο μισελ και την κυρία ούρσουλα φον λάιεν και έφυγε επιδεικτικά και δεν πήγε τον ακούσατε τον υπουργό να υβρίζει τρία κράτη της ευρωπαϊκής ένωσης και δεν του απαντήσατε και δεν είχατε την αντίδραση την οποία έπρεπε να είχατε και ήταν σαν να δίνετε άφεση αμαρτιών στην τουρκία. εσείς όμως έπρεπε να αναφέρετε τα συμπεράσματα του συμβουλίου Ευχαριστούμε κύριε Μημαράκη. Για ένα λεπτό το λόγο έχει κυρία Σιμακοπούλου. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Μπορέλ, μόλι χθε εδώ σε αυτή την αίθουσα η καγκελάριο Μέρκελ εξήρε το ρόλο μα ω ευρωβουλευτέ στο να εξηγούμε στου πολίτε τι πολιτικέ τη Ένωση. Σα ρωτώ λοιπόν κύριε Μπορέλ, πώ να εξηγήσω εγώ στου συμπολίτε μου στη Ρόδο, στην Κάρπαθο, στην Κάσο και στην Κρήτη τι παράνομε τουρκικέ γεωτρήσει που παροβιάζουν κατάφορα το διεθνέ δίκαιο πώς να εξηγήσω στους συμπολίτες μου στον εύρο στη λέσβο στη χίο στη σάμο που υποδέχονται χιλιάδες πρόσφυγες και μετανάστες δείχνοντας πρωτοφανή αλληλεγγύη τα fake news των τούρκων που τους παρουσιάζουν ως δολοφόνους μικρών παιδιών και πώς να εξηγήσω στους χριστιανούς συμπολίτες μου ότι η αγία σοφιά μπορεί να μετατραπεί σε τζαμί και πώς μα πώς να εξηγήσω στους συμπολίτες μου ότι όταν ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών απειλεί απροκάλυπτα την Ένωση και αρνείται να αναγνωρίσει ένα κράτος μέλος μας την Κύπρο εσείς ο ύπατος ε, ε, μας χαμογελάτε δεχόμενος δώρο ένα απολυμαντικό για τα χέρια. Αν μετά από όλα αυτά, κύριε Μπορέλ, καλούμε να εξηγήσω στους συμπολίτε μου ότι αυτό που χρειαζόμαστε αντί για κυρώσεις είναι επικοδομητικός διάλογος με την Τουρκία, τότε τουλάχιστον ως ένδειξη σεβασμού να λείπουν τα χαμόγελα. Σας ευχαριστούμε κυρία Σιμακοπούλου. Ένα λεπτό κύριος Κέλλη έχει τώρα το λόγο. Όταν πρώτο ξεκίνησα το Brexit πολύ στην Ιρλανδία ένιωσαν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπάθησε να λύσει τα θέματα με το Ολλανδικό σύνορο για να καθησυχάσει τους Βρετανούς και νομίζαμε ότι θα, θα υποκύψει μάλλον στο, στους Βρετανούς για να τους δείξει καλή θέληση και δεν έγινε αυτό, μας υποστήριξε, έδειξε αλληλεγγύη. Το ίδιο θέλουμε για την Ελλάδα και την ε, Κύπρο, ε, διότι ε, δεν είναι μόνο οι κακές σχέσεις γειτονίας, αλλά είναι η παραβίαση των εθνικών συνόρων που επιχειρείται και η παραβίαση τη εθνική κυριαρχία. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να παραβιάσει την εθνική κυριαρχία των κρατών μελών τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλα τα κράτη-μέλη τη Ένωση είναι σημαντικά για εμά. Και αν δεν αντιδράσουμε με το σωστό τρόπο, τότε θα πρέπει να κάνουμε εμείς ό,τι μπορούμε για να σταθούμε ε, στο ανάστημά μας. Ε, ε, και όπως υπήρξε αλληλεγγύη προς την Ιρλανδία απέναντι στο Brexit και τη Συμφωνία Αποχώρησης, το ίδιο πρέπει να δείξουμε την ίδια αλληλεγγύη απέναντι στην Ελλάδα και την Κύπρο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ η κυρία Σπυράκη έχει το λόγο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είπατε εκπρόσωπο κύριε Μπορέλ, όπως γνωρίζετε η Ελλάδα συνομολόγησε ήδη τη συμφωνία για τα όρια της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης με την Ιταλία και εργάζεται σε αυτή την κατεύθυνση και με την αίγυπτο. στόχος της ελλάδος είναι η διαπραγμάτευση με την τουρκία για την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης και σε περίπτωση μη συμφωνίας η προσφυγή από κοινού στο διεθνές δικαστήριο της χάιγης. η τουρκία απειλεί επισήμως την εδαφική ακεραιότητα της ελλάδος και αμφισβητεί τις διεθνείς συμφωνίες. ξέρετε η οριοθέτηση τη σαός της ελλάδος με την τουρκία δεν είναι μια διμερής υπόθεση. η ελλάδα θα έχει τη δυνατότητα να συμβάλει στη διαφοροποίηση των προμηθευτών ενέργειας στην ευρωπαϊκή ένωση αυξάνοντας την αυτονομία της. γι' αυτό η ευρωπαϊκή ένωση έχει κάθε συμφέρον όχι μόνο να επαναλαμβάνει τυπικά και φραστικά τη θέση της για την ΑΟΣ αλλά κυρίως να οθήσει την τουρκία ώστε να καταστεί υποχρεωτική για αυτή η διευθέτηση της ΑΟΣ είτε με διαπραγμάτευση είτε μέσω της αμοιβαίας προσφυγής στη χάγη. σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε και την κυρία Σπυράκη και η συζήτηση, το κομμάτι αυτό τη κοινή συζήτηση ολοκληρώνεται με την κυρία Ζωξία Βιτσιένη. Για ένα λεπτό ευχαριστώ πολύ. Η κατάσταση στη νότια γειτονία τη Ευρωπαϊκή Ένωση είναι επικίνδυνη και αυτό θα πρέπει να ειδωθεί στο ευρύτερο πλέξιο και όχι μόνο σε σχέση με την ε, Τουρκία. Υπάρχουν ε, πολλέ συζητήσει σε σχέση με τη στρατηγική αυτονομία τη Ευρωπαϊκή Ένωση στον τομέα τη άμυνα. Οι διάφορε αυτέ διεργασίε στη γειτονία τη Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ και σειρά ετών δείχνουν πλέον ότι είναι ανάγκη να μην μείνουμε στα λόγια, αλλά περάσουμε στα έργα. Διότι όταν παραμένουμε εμεί αδρανεί, παίρνουν άλλη τη σκητάλη. Στην προκειμένη περίπτωση η Τουρκία και η Ρωσία. Και ακόμα χειρότερα, υπάρχουν αρκετά κράτη-μέλη που ε, υποστηρίζουν διαφορετικέ πλευρέ, διαφορετικά στρατόπεδα επίπεδα τη ε, ε, αντιπαράθεση στη Λιβύη. Πού είναι εδώ η ευρωπαϊκή στρατηγική. Πρέπει να μιλήσουμε για την δυνατότητα τη Ευρωπαϊκή Ένωση να δρά κοντά στα σύνορά τη σε συντονισμό με τον ΝΑΤΟ. Αυτό θα είναι το είδο μια στρατηγική αυτονομία τη Ένωση, την οποία θα μπορούσαν να πιστέψουν οι ψηφοφόροι μα. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ πολύ και την ε, κυρία Γιουκνε Βιτσιέν. Ολοκληρώθηκε λοιπόν για το δεύτερο τμήμα τη κοινή συζήτηση σε ό,τι αφορά τη σταθερότητα στη Μεσόγειο και την, ε, τον αρνητικό ρόλο της Τουρκίας και προχωρούμε στο τρίτο τμήμα της κοινή συζήτησης που ε, θα αφορά την κατάσταση στη Λευκορωσία. Ο κύριος Κουμπίλιους είναι ο πρώτος ομιλητής. Για 1,5 λεπτό έχετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Παντεκπρόσωπε, μετά από 26 χρόνια αυταρχικής κυβέρνησης του Λουκασένκο ζητούν οι πολίτες της Λευκορωσίας μια δημοκρατική αλλαγή και αυτό μπορεί να γίνει στις 9 Αυγούστου στις προεδρικές εκλογές. Τα πράγματα έχουν αλλάξει σε σχέση με το παρελθόν. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι πάνω από 5% των Λευκορώσων θέλουν πραγματική αλλαγή και μόνο μια μειοψηφία θέλει να παραμείνει Λουκασένκο. Αυτό θυμίζει ε, την ε, ε βελούδινη επανάσταση στη Βαλτική στη δεκαετία του 90 ε, αρχίζουν ε, άτομα της πολιτιστικής ελίτ να μιλούν στο ραδιόφωνο κατά του καθεστώτος ε, επιγραμμικά δημιουργούνται δίκτυα αντίστασης και όλοι αυτοί βεβαίως διώκονται από το καθεστώς ο σημαντικός σημαντική της αντιπολίτευσης είναι στη φυλακή μεταξύ των οποίων ο Παύλος Ευρένιες θέλουμε να στείλουμε τρία σαφή μηνύματα. Πρώτον, προ του πολίτε τη Λευκορωσία. Είμαστε αλληλέγγυοι στο αίτημα αλλαγή του λαού τη Λευκορωσία, στο δικαίωμα να αποφασίσει να αλλάξει, να γίνει μια πραγματική ευρωπαϊκή δημοκρατία. Ένα μήνυμα προ προς τον κύριο Λουκασέγκο. Εάν έω 14 Ιουλίου ε, ε, δεν απελευθερωθούν οι πολιτικοί κρατούμενοι, δεν επιτραπεί στου ηγέτε τη να συμμετάσχουν στι εκλογέ, θα υπάρξουν κυρώσει και τρίτο μήνυμα προς εμάς. Πρέπει να υπερασπιστούμε τα δικαιώματα των γειτόνων μας. Σας ευχαριστούμε κύριε Κουμπίλιος. Ένα λεπτό ο κύριος Μπιεντρών. Just on our border, in the heart of... Εδώ στα σύνορά μας, στην καρδιά της Ευρώπης, είναι οι γείτονές μας. Ο λαός της Λευκορωσίας που στερείται τα θεμελιώδη τους. Είμαστε στο πλάι τους. Μήνυμα ξεκάθαρα πρέπει να στείλουμε προς τον Λουκασέγκο. Καταδικάζουμε με αποφασιστικότητα όλα αυτά. Θα πρέπει άμεσα να αποφυλακιστούν όλοι οι αδίκως συλληφθέντες. 26 χρόνια είναι στην εξουσία. Αλλά δεν υπάρχει πολιτικός βίος εκεί. Υπό αυτές τις συνθήκες η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αποκτήσει μια υπεύθυνη στρατηγική και πολιτική προς τη χώρα εκείνη. Ξεκάθαρη πολιτική με προϋποθέσεις και αιρεσιμότητα. Να δούμε πώς δικαιολογείται αυτή μας η στάση. Τι θα γίνει στο μέλλον, χωρίς στρατηγική. Πέστε μας. με έγγραφη δήλωση, αν θέλετε, τις ε, επόμενες εβδομάδες. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Μπιεντρών. Για δυόμιση λεπτά έχει το λόγο και ο Στρεβίτσιους. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πέντε εκπρόσωπε, κυρίες και κύριοι, σήμερα στην χώρα διαπιστώνουμε διαδικασίες που αποτελούν κάποιες ε, νόθες εκλογές, εκλογές μόνο προσχηματικές. Οι διεθνεί παρατηρητές κατέγραψαν όλες αυτές τις εκλογικές ε, παραβάσεις ε, για αυτές τι προεδρικές εκλογές. Το καθεστώ της χώρας έχει αποτύχει να καλύψει τον λαό. Δυσαρέσκεια. Έχει εξαντληθεί η υπομονή του κόσμου. Υπάρχει τώρα μια ε, ακτίδα ελπίδας από αυτές τις εκλογές αλλά ο πρόεδρος της χώρας συνεχίζει εκφοβισμούς, καταστολή, ε, δικαστήρια και συλλήψεις, απαγωγές και ξυλοδαρμός από την Καγκεμπέ. Ο Κομπορίκα και ο Τσιχανόφσκι είναι ακτιβιστές που είναι ακόμη στη φυλακή. Υπάρχουν κρατούμενοι συνείδησης πριν από τρία χρόνια ο Νικόλαη Στατικέβιτ είχε απελευθερωθεί ένα άλλο αρνητή συνείδηση και τώρα ξαναφυλακίστηκε ο Σεβερίνατ. Επίση, άλλο κρατούμενο ε, υπέστη παράταση τη απόφαση φυλάκιση. Έχουμε και το Οστροβέτς, το οποίο είναι πυρηνικές εγκαταστάσεις που δεν συμμορφώνται προς τις διεθνείς ε, ε, προδιαγραφές ασφαλεία, δίπλα στα σύνορά μα. Το κατασκεύασαν οι Ρώσοι και το χρηματοδοτούν. Πρόκειται ουσιαστικά για έναν δούριο ύπο ει βάρο τη ασφάλεια τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Απευθύνω έκκληση στα θεσμικά όργανα να υπάρξει μια ολοκληρωμένη στρατηγική εναντί τη χώρα. Θα πρέπει να βασίζεται σε ευρωπαϊκή προοπτική, ε, με σεβασμό τη ε, κυριαρχία, τη δημοκρατία. να υπάρχουν ελεύθερε εκλογέ, πλουραλισμό και θα πρέπει να σεβαστούν τις διεθνείς προδιαγραφές ασφαλείας για τα πυρηνικά. Δεν θα πρέπει η βοήθεια μας για την πανδημία προς τη χώρα να μην ε, καταλήξει να είναι υποστήριξη στο καθεστώς της χώρας. Θα πρέπει να αντλήσουμε συμπεράσματα από το ότι σταματήσαμε τις κυρώσεις το 2016 είδατε τι έγινε. Να αντλήσουμε συμπεράσματα από αυτό. Ζήτω η χώρα, ζήτω η Λευκορωσία. Ευχαριστώ πολύ για δύο λεπτά κύριε Φων Κράμον Ταουμπάντλ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πατεκπρόσωπε, αξιότιμοι συνάδελφοι, σε πολλά κράτη της ανατολικής γειτονίας έχουμε να κάνουμε με αυταρχικά καθεστώτα και αποτυχημένη δημοκρατία. Αλλά η απόκληση ε, δεν είναι πουθενά εντονότερη όταν έχουμε αυτό τον πρόεδρο στη ε, Λευκορωσία με αυτή την καταστολή, με αυτή την πίεση. Σχεδόν τραγικό είναι να παρακολουθεί κανείς αυτή τη χώρα που είναι στα μέσα από γεωγραφικής πλευράς της Ευρωπαϊκή Υπήρους ε, να έχει μια τέτοια κυβέρνηση που τόσο πολύ μακριά βρίσκεται από τις δικές μας αξίες Υπάρχει ακόμη θανατική ποινή σε αυτή τη χώρα, στο Μίνσκ. Δεν έχουμε να κάνουμε μόνο ε, πρόεδρο που αρνείται τον ε, κορονοϊό, αλλά ε, και έναν άνθρωπο που θέλει να παραμείνει στην εξουσία. 26 χρόνια είναι εκεί ο Λουκασέγκο και ε, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να τον ανταγωνιστούν. Αυτός φοβάται τον ανταγωνισμό, δεν θέλει να δεχτεί κανέναν ε, άλλο υποψήφιο, παρότι μπορεί να στέκονται στις ουρές ε, ώρες οι άνθρωποι για να προτείνουν κάποιον υποψήφιο. Πράγματι, με την δράση της μάθαμε πρόσφατα στοιχεία. Μέσα στην Ευρώπη γίνονται αυτά τα πράγματα. υπάρχουν σίγουρα αυτά τα οποία πρέπει να έχει κάνει το μήνυμα, όπως ο κ. Μπόρελ. Πρώτα απ' όλα, να υπάρχει αυτή η αποστολή παρατήρησης. Επίσης, σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να τολμά ε, τους υποψηφίους ε, για την ε, θέση του να μην τους καταχωρίζει, να μην τους δέχεται ο Λουκασίνκο. Τρίτον, όλοι οι πολιτικοί κρατούμενοι πρέπει άμεσα να φεθούν ελεύθερα και αλεύθεροι και άνευ όρων και προποθέσεων. Θα πρέπει επίσης και εμείς από τις Βρυξέλλες αλλά και από τους θεσμούς που εκπροσωπούνται εκεί να, ε, και με τη βοήθεια των κρατών μελών να προσπαθήσουμε να επιβληθούν αυτοί οι όροι γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι ένα τεστ αξιοπιστία μας ε, προ τα έξω. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρο, σα ευχαριστώ πολύ κυρία Φονκράμον. Ε, τώρα ένα λεπτό έχει το λόγο και ο Σπινέδ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ας μιλήσουμε καθαρά Γίνεται αυτή η συζήτηση σήμερα για τη Λευκορωσία διότι πλησιάζουν εκλογές και θέλετε να επηρεάσετε τις εκλογές. Ουσιαστικά εφαρμόζεται την ανάμειξη ιστορικά μιας άλλης χώρας. Αυτά έχουν γίνει και στο παρελθόν και είναι επικίνδυνα. Όταν προωθούμε αλλαγή καθεστώτος και κυβερνήσεων με κάθε κόστος, μπορούμε να βρεθούμε ξαφνικά με ναζιστικές κυβερνήσεις, όπως γίνει στο παρελθόν. Τα ανατολικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ένα έδαφος το οποίο είναι εξαιρετικά στρατικοποιημένο. Είχαμε ασκήσεις, γυμνάσια του του ΝΑΤΟ με 35.000 στρατιώτες που υποστηρίζουν Αμερικανοί στα σύνορα με τη Λευκορωσία. Αυτό είναι καλό για τους λαούς της Ευρώπης. Όχι. Είναι καλό για να τροφοδοτούμε το νέο ε, ψυχρό πόλεμο του κυρίου Τραμπ. Πρέπει να βάλουμε τέλος στο παρελθόν. Χρειαζόμαστε μια αυτόνομη, ανεξάρτητη, κυρια... Ε, κυρίαρχη εξωτερική πολιτική υπέρ ε, της ειρήνης στην Ήπειρό μα και όχι υπέρ της έντασης. Ευχαριστούμε κύριε Πινέδα. Ένα λεπτό κύριος Γκάλερ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αυτό που είπε ο ε, προλαλής σας ε, ήταν ε, εντυπωσιακό. Σαν να μίλαγε υπέρ του Λουκασέγκο. Μα έχετε υπόψη σας τι γίνεται στη Λευκορωσία. Μετά από 26 χρόνια έχουν μπουχτίσει, για να μην πω τίποτε χειρότερο, από αυτό το καθεστώς οι Λευκορώσοι και θέλουν αλλαγή. Δεν το θέλουμε εμείς. Οι ίδιοι το απαιτούν. Οι Λευκορώσοι. Είναι σημαντικό η ε, πρόσκληση αυτή ε, να ε, γίνει και να υπάρξει αποστολή της επιτήρησης παρακολούθησης εκλογών εκεί. Και σίγουρα πρέπει να καταχωριστούν όλοι οι υποψήφοι, να είναι δυνατόν να συμμετέχουν και άλλοι υποψήφοι σε εκλογές. Είναι καλό που υπάρχει συνένεση ακόμη και από την αριστερά ως προς αυτό και είναι καλό να γίνουν αυτές οι προεδρικές εκλογές Υπάρχουν διάφορες τακτικές ε, για το πώς θα διεξαχθούν και οι εκλογές και, ε, τα, και η προεκλογική. Εντάξει, η προεκλογική Εντάξει, σταματώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Ε, κύριος Νόιζερ έχει τώρα το λόγο για ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, κύριε είπατε εκπρόσωπε, πιστεύω ότι είναι άκρος ανησυχητική η κατάσταση στη Λευκορωσία μέχρι την ημέρα των εκλογών την 9η Αυγούστου θα επιδεινωθεί ακόμη περισσότερο. Βλέπουμε αυθαιρεσίε, βλέπουμε αποκλεισμό ε, της αντιπολίτευσης, των αντιφρονούτων, ε, το ίδιο για του ακτιβιστέ και την κοινωνία των πολιτών, απαγόρευση ειρηνικών διαδηλώσεων κτλ. Τι μπορούμε εμεί να κάνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω ότι αυτό το οποίο χρειάζεται είναι να δοθεί μια πιο ισχυρή κοινή απάντηση. Απάντηση από πλευρά ε, τη ε, Κομισιόν αλλά και της Γερμανικής Προεδρίας Νομίζω ότι θα πρέπει να επηρεάσει το Βερολίνο. Είναι σημαντική η επιρροή του Βερολίνου σε αυτή την περίπτωση. Και επίσης χρειαζόμαστε εταιρικέ σχέσεις και επαφές προσωπικές με αυτούς τους οποίους προσπαθεί να καταστήλει και καταστέλει το καθεστώ Λουκασέγκο αυτή τη στιγμή. Γιατί όλα αυτά ε, έχουν να κάνουν με, ε, με το ίδιο ε, τις αξίες μας και στις οποίες σα Ευχαριστώ πολύ. Κάλλος μπορεί η επόμενη μιλητρία. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε είπατε εκπρόσωπε. Πρόεδρος, δικτάτορας είναι ο Λουκασέγκο. 26 χρόνια τώρα κυβερνά. Κατάχρηση εξουσίας, ψέματα και καταπάτηση ελευθεριών και δικαιωμάτων. Είναι η μόνη ευρωπαϊκή χώρα που έχει την θανατική ποινή. Χειρότερα γίνονται τα πράγματα κάθε μέρα. Συλλαμβάνουν τον κόσμο, τον φυλακίζουν, αν διαμαρτύρεται και τώρα χρησιμοποιούν και τα όπλα για νόμιμες ενέργειες, δηλαδή για το αίτημα εκλογών. Εμείς έχουμε απευθυνθεί στην ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ούτως ώστε να υπάρξουν κάποιες κυρώσεις κατά του Λουκασέγκο. Να μην του λέμε και μπράβο. Επιβολή κυρώσεων, αυτό θέλουμε. Πρόκειται για ένα σκάνδαλο να επιτρέπονται τέτοια πράγματα και να συνεχίζονται στην Ευρώπη. Ο φουντώνει, φουσκώνει η δυσαρέσκεια στη χώρα έχουμε την ευκαιρία να τον καταδικάσουμε και να στηρίξουμε τους δημοκράτες. Όλους που έχουν φυλακιστεί για πολιτικούς λόγους που πρέπει άμεσα να αποφυλακιστούν, να υποστηρίξουμε με έναν δημοκρατικό μετασχηματισμό στη χώρα. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Τόμακ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Χτες ήταν εδώ η καγκελαρία Μέρκελ, κύριε Μπορέλ, και έλεγε ότι είναι προτεραιότητά μα η προστασία των αξιών μα τα θεμελιώδη δικαιώματα. Όλα αυτά είναι αδιαπραγμάτευτα. Είναι απαράδεκτο στα σύνορα μας δίπλα να υπάρχει ένας δικτάτορας που διώκει τον λαό του και καταπατά αυτές τις αξίες μας. Γι' αυτό σας λέω κύριε είπατε εκπρόσωπε θα πρέπει να κάνετε κάτι, να υπάρξουν κυρώσεις κατά αυτού του καθεστώτος. Να ε, υπερασπιστούμε ε, την δημοκρατία και το κράτος δικαίου. Να προσέξουμε αυτή την κατάσταση. Το αξίζει ο λαός της χώρας. Σας ευχαριστώ πολύ. Για ένα λεπτό, κύριος Όλεκας. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, το 2020 θα είναι μια χρονιά που θα τη θυμόμαστε. Μια χρονιά με πολλές αλλαγές. Σε ό,τι τη Λευκορωσία όμως δεν βλέπουμε τόσες αλλαγές. Ο πρόεδρος Λουκασένκο έχει ουσιαστικά εξολοθρεύσει όλους τους ε, υποψήφιους εκλογές. Έχουμε αυθαίρετες συλλήψεις, κρατήσεις. Θα πρέπει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση να επιβάλλει κυρώσεις, να ενισχύσει τις κυρώσεις απέναντι στο καθεστώς Λουκασένκο. Ταυτόχρονα δεν μπορούμε οι κυρώσεις αυτές, δεν πρέπει οι κυρώσεις αυτές να πλήξουν τον λαό της Λευκορωσίας. Πρέπει να ενισχύσουμε τους δεσμούς μας με την κοινωνία των πολιτών της Λευκορωσίας, να τους φέρουμε στην Ευρώπη, ε, να δείξουμε ότι δεν τους ξεχνάμε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Όλεκας. Ε, για να ολοκληρωθεί αυτή η κοινή συζήτηση θα πάρει το λόγο για μια ακόμη φορά ο κύριος Μπορέλος, εκπρόσωπος ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αντιπρόεδρος αλλά και από τους εκπρόσωπους του Ευχαριστώ. Δεν ξέρω πόσο χρόνο έχω στη διάθεσή μου, Πρόεδρε. Δεν είστε πλέον Ευρωβουλευτή, άρα δεν έχετε κάποιο περιορισμό στο χρόνο αγόρευση. Μπορείτε να μιλήσετε όσο θέλετε, κύριε Μπορέλ. Α, πολύ ωραία. Πολύ ωραία, λέει ο κ. Μπορέλ. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, θα απαντήσω στη γλώσσα μου, στα ισπανικά, για να εκφραστώ έτσι και πιο ευθέως. Το να συνδέσουμε τρεις συζητήσεις για τρία τόσο σημαντικά ζητήματα ε, κάπως ε, μπερδεύει τα πράγματα. Η έκθεση για ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο, παραδείγματο χάρη, από μόνη τη ε, θα ήθελε, θα χρειαζόταν μια συζήτηση. Διότι το εύρος που καλύπτει αυτή η έκθεση είναι τεράστιο. Δεν είναι βέβαια ένα κείμενο το οποίο <laughs> επιλύει τα προβλήματα δεν επιλύονται προβλήματα διαβάζοντα κείμενα, τέτοιου είδου προβλήματα. Είναι μόνο σημαντική, μια σημαντική έκθεση. Είναι σημαντικό επίσης να έχουμε κατά νου ότι πέρα από το να εξηγούμε τι συμβαίνει πρέπει και να δράσουμε. Εξού και το νέο σχέδιο δράσης για την επόμενη τετραετία έτσι ώστε η δραστηριότητά μας ε, να μην είναι μόνο αυτή του επεξηγητή αλλά αυτού που προσπαθεί να διορθώσει, να παρέμβει. Βεβαίως και ε, δίνουμε πολύ μεγάλη έμφαση στα ανθρώπινα δικαιώματα και έχουμε ένα μηχανισμό που θα παίξει ένα πολύ σημαντικό ρόλο για να εφαρμοστεί το σχέδιο αυτό. Υπάρχουν και περιορισμοί, το γνωρίζω. Βεβαίω κάποιοι από εσά ε, ε, έχουν μεταφέρει τη συζήτηση για την έκθεση αυτή με τα που συμβαίνουν στο εσωτερικό της Ένωσης ε, έχουν αλλοιώσει δηλαδή κάπως το περιεχόμενο της συζήτησης έγιναν κάποιες αρκετά συγκεκριμένες αναφορές ε, έγινε αναφορά στη συμμετοχή, στη μας ε, στη δημιουργία ενός ε, οργάνου σε επίπεδο ενωμένων Εθνών που να είναι νομικός δεσμευτικό για την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, δυστυχώς δεν υπάρχει εντολή από το Συμβούλιο για να συμμετάσχουμε στη δημιουργία αυτού του μέσου εμείς θεωρούμε ότι είναι αναγκαίο και συμμετέχουμε στις διαβουλεύσεις ε, ατύπως όπως πρόσφατα τον Μάιο στο Εκουαδόρ στον Ισημερινό και θα συμμετάσχουμε και στην επόμενη συνάντηση τον Οκτώβριο εξεκολουθούν να θεωρούμε την απαραίτητο ένα τέτοιο όργανο, ένα τέτοιο μέσο δεν έχουμε όμως δυστυχώς επαναλαμβάνω λάβει εντολή από το Συμβούλιο για να συμμετάσχουμε επισήμω. αποφασίσαμε να ανανεώσουμε την ε, θητεία του ειδικού εκπρόσωπου που ε, υπερασπίζεται την ελευθερία του θρησκεύματος υπάρχει και πάντως εκπρόσωπος για τα ανθρώπινα δικαιώματα συνεργάζονται ε, είναι και αυτό μια προτεραιότητα σε ό,τι αφορά την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων η ελευθερία του θρησκεύματος η οποία απειλείται σε πολλές περιοχές του κόσμου και σε κάποιες περιπτώσεις αυτό βεβαίως πλήττει Ευρωπαίους πολίτες πολλούς ε, χριστιανούς. Σε ό,τι αφορά τώρα την χορήγηση θεωρήσεων σε υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, το ερώτημα αυτό είναι εξαιρετικά ε, κέριο. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι τις θεωρήσεις δεν τις, δίνουν, δεν τις δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τις δίνουν τα κράτη-μέλη. Και η άρνηση εισόδου στο έδαφος ε, ναι, ναι, βεβαίω. Τι θεωρίε δεν τι δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, επαναλαμβάνω. Τι δίνουν τα κράτη-μέλη. Ε, να το θέλουν. Εμεί αυτό που κάνουμε με τι αντιπροσωπείε μα είναι να φέρνουμε σε επαφή συνεχώ τις πρεσβείες των κρατών μελών με τους υπερασπιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων που βρίσκονται σε κάποια ε, κατάσταση κινδύνου που απειλούνται για να μπορέσουν να σχολιαστούν θεωρήσεις. Από τα κράτη-μέλη όμως. Θα εξετάσω την απάντηση που λάβατε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που μου είπατε για να δω επακριβώς ε, ε, ποια ήταν η διατύπωση και κατά πόσο ε, αντικατοπτρίζει τη βούλησή μας να υποστηρίξουμε τους υπερασπιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων όσο μπορούμε. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να πω πολλά για όλα τα ζητήματα που αναφέρει η έκθεση, αλλά δεν θα μπορέσω να το πράξω και θα περάσω ευθύς αμέσως ε, στο επόμενο ε, θέμα που μας απασχολεί σήμερα χωρίς βεβαίως να ξεχάσω να πω ότι το θέμα της προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας ανά τον κόσμο έχει τεράστιο εύρος, τεράστια έκταση. Διότι διαπιστώνουμε βεβαίως ανθρώπινα δικαιώματα απειλούνται απειλούνται όλο και περισσότερο. Γνωρίζουμε ότι η αυταρχικότητα ε, αναζωογονείται ε, σε πολλές περιοχές του κόσμου, ορισμένες φορές μάλιστα με προσωπείο δημοκρατίας που χρησιμοποιούν τις διαδικασίες δημοκρατικές που δεν είναι όμως πραγματικά δημοκρατικές διαδικασίες. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό που κάνουμε και ακόμα περισσότερα με τη βοήθεια των βουλευτών και γι' αυτό η έκθεση αυτή θα έπρεπε να έχει συζητηθεί επιμέρους, αποκλειστικά σε μια συζήτηση. Τώρα, για το θέμα της Τουρκίας. Ακούστε, εγώ αντιλαμβάνομαι πολλά από τα επιχειρήματα τα οποία ακούστηκαν. Όμως, ε, εδώ σήμερα ε, στη συζήτηση υπήρχε έτσι μια διάσταση σχεδόν εμπόλεμη, πολεμική. Είχα την εντύπωση ότι εμφανίστηκε ξαφνικά ο ο Πάπας ε, Πίος 15ος, ο οποίος ε, ζητούσε ιερά συμμαχία κατά της Τουρκίας, ε, κινητοποιώντας ε, τον στόλο του χριστιανισμού για να βάλει φρένο στην Οθωμανική εισβολή. Εγώ δεν είμαι ούτε Τσάμπερλεν βεβαίω, ούτε Νταλαντιέ, αλλά ούτε ο, ο Ιωάννης της έτσι. Διότι αυτά αφορούν άλλες ιστορικές περιόδους δεν ψάχνουμε την αντιπαράθεση. Θέλουμε να αποφύγουμε την αντιπαράθεση. Και γι' αυτό πολλάκις έχω εκφραστεί επί του στήματος και πιο πρόσφατα στην ίδια την Τουρκία, στην Άγκυρα, εκφράζοντας στεναρά την υπεράσπιση τη δραστηριοτική κυριαρχία των συμφερόντων των κρατών μελών που πλήττονται από δραστηριότητε που θεωρούμε ότι είναι παράνομε τη Τουρκία σε ό,τι αφορά τι γεωτρήσει. Ταυτόχρονα εγώ πρέπει να πω ότι η γεωγραφία δεν θα αλλάξει. Εκεί θα είναι η Τουρκία και θα πρέπει να έχουμε μια επικοδομητική σχέση μαζί της. Και αυτό σημαίνει ότι δεν πρέπει να υπάρξει κλιμάκωση της έντασης, η οποία δυστυχώς πήρε και τη μορφή επεισοδίων με ε, πολεμικά πλοία, ε, ευρωπαϊκά, τουρκικά, που είναι και μέλη της ίδιας ε, συμμαχίας στρατιωτικής ε, του ΝΑΤΟ και βεβαίως ε, λαμβάνει έρευνα για το θέμα αυτό, έτσι, σε επίπεδο ΝΑΤΟ. Λαμβάνει χώρα έρευνα. Αυτό που πρέπει να αποφύγουμε βεβαίως είναι να επαναληφθούν τέτοια φαινόμενα. Επαναλαμβάνω, εδώ δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε μια ιερή συμμαχία κατά της Οθωμανικής εισβολής, διότι αυτό φάνηκε να προτείνουν κάποιοι εδώ θέλουμε με επικοδομητικό τρόπο απέναντι σε μια περίπλοκη πραγματικότητα το είπαν και κάποιοι από τους ε, ε ομιλητές η κυρία Ζώου, ο Σάντσες Αμόρ να αναζητήσουμε μια διαδικασία που θα συμπεριλαμβάνει μια διαπραγμάτευση για τα ζητήματα που δημιουργούν αυτή τη στιγμή ένταση μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας διότι είναι πολλά τα προβλήματα αυτά προς επίλυση και είναι αναγκαίο να επιληθούν. Και αυτό μπορεί να συμβεί μόνο μέσα από τη διαπραγμάτευση και τον διάλογο. Με μια αποφασιστική στάση, αλλά αποφεύγοντας μια κλιμάκωση της έντοσης. Της έντασης διότι αυτό δεν συμβάλλει στην επίλυση των προβλημάτων. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε εμείς. Αυτό προσπαθώ να κάνω εγώ και θα συνεχίσω να προσπαθώ με την υποστήριξη των συναδέλφων ε, στο Συμβούλιο Πονών Εξωτερικών. Την επόμενη Δευτέρα, άλλωστε, θα συζητηθεί το θέμα αυτό. Είναι στη μέση διάταξη του Συμβούλιου Υπουργών Εξωτερικών και για την προπαρασκευή μάλιστα αυτής της συνάντησης ε, μετέβη και στην Ελλάδα και στην Κύπρο και στην Τουρκία. Σε ό,τι αφορά τώρα τη Λευκορωσία, Πρόεδρε, δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω με αυτά που ελέγχθησαν. Το έχουμε πει από την αρχή της εκλογικής διαδικασίας εκεί. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή συνθήκες στη χώρα αυτή εξαιρετικά ανησυχητικέ καταστολή, παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τις αρχές της Λευκορωσίας Έχουμε στείλει πολύ σοβαρά προειδοποιητικά μηνύματα. Υπάρχει κατάλογος με αυτά που έχουμε πει και επισήμως ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Ταυτόχρονα θα πρέπει να είμαστε σε συνεχή επαφή με την κοινωνία των πολιτών, με τη Λευκορωσία, έτσι ώστε να μπορούμε να επηρεάσουμε την πραγματικότητα ε, και να βελτιώσουμε την κατάσταση για τους πολίτες της Λευκορωσίας σε αφορά τη σχέση τους με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τα δύο αυτά στοιχεία δεν είναι αλληλοαποκλειόμενα, δεν είναι ασύμβατα. Μπορούμε κάλλιστα να υπερασπιστούμε ε, τα δικαιώματα των πολιτών της Λευκορωσίας, την ανεξαρτησία, την κυριαρχία της χώρας και ταυτόχρονα να συμμετάσχουμε σε επαφές με την κοινωνία των πολιτών να αφήσουμε ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας. Κάτι παρεμφερές θα μπορούσε να υποθεί και για τη Ρωσία. Πολλοί από εσά αναφέρθηκαν στην χρηματοδότηση της Τουρκίας ε, με κονδύλια προενταξιακά. Πρέπει να ξέρετε ότι από το 2017 αυτά τα κονδύλια έχουν περικοπεί κατά 1,3 δις. Και αυτή τη στιγμή τα χρήματα που διατίθενται έχουν να κάνουν με τον τομέα της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την υποστήριξη της κοινωνίας των πολιτών και 160 εκατομμύρια για την ανάπτυξη μάλλον 18 εκατομμύρια συγγνώμη 18 εκατομμύρια για την ανάπτυξη της υπαίθρου δεν υπάρχουν χρήματα προενταξιακά τα οποία να δίνονται στον οικονομικό τομέα διότι τα χρήματα αυτά όπως σας είπα έχουν μειωθεί πολύ σημαντικά λόγω ακριβώς της τάσης της Τουρκίας την οποία το Συμβούλιο θεώρησε μη συμβατή με τη στάση μιας υποψήφιας χώρας. Είναι προφανές λοιπόν ότι χρησιμοποιήσαμε τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας. Μην τα μπερδεύουμε όμως όλα. Μην μπερδεύουμε τα προταξιακά κονδύλια με τα κονδύλια που διαθέτουμε για να υποστηρίξουμε ε, τους ε, ε, Σύριους εξόριστους που βρίσκονται στην Τουρκία. 3,5 εκατομμύρια άνθρωποι. Βεβαίως και είναι σημαντική η επιβάρυνση για τη χώρα που τις υποδέχεται. Το να δίνουμε χρήματα για να διευκολύνουμε την ε, υποδοχή των ανθρώπων αυτών για σχολεία, για υγειονομική περίθαλψη, τι κακό έχει αυτό. Πώς να σταματήσουμε να το κάνουμε αυτό. Πρέπει να συνεχίσουμε να το κάνουμε. Πρόσφατα αποφασίστηκε να διατηρηθούν 500 εκατομμύρια ακόμα για την υποστήριξη των Σύριων προσφύγων. Δεν είναι χρήματα για την Τουρκία αυτά. Αυτά τα χρήματα πάνε απευθείας στην βοήθεια μέσω μη κυβερνητικών οργανώσεων που εργάζονται στην περιοχή και μέσω των οργανισμών των ΗΕ Εθνών για να βοηθηθεί, να βοηθούν οι άνθρωποι στην απελπιστική κατάσταση στην οποία βρίσκονται. Οι Σύριοι πρόσφυγες. Δεν μπορείτε να το επικρίνετε αυτό. Δεν μπορείτε να λέτε ότι εδώ ε, τα έχουμε βρει με την Τουρκία ας πούμε και τους δίνουμε χρήματα. Όχι. Είναι αναγκαίο να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε την προσπάθεια βοήθειας, ανίσχυσης προς ανθρώπους αυτούς όπως το κάνουμε στην Ιορδανία, όπως το κάνουμε στο Λίβανο. Τώρα, για τη Λευκορωσία επανέρχομαι. Ε, Όντω τα πράγματα μπορεί να χειροτερέψουν. Και εμείς έχουμε μέσα δράσεις περιορισμένα μεν. Ε, εμείς ε, έχουμε κάνει ό,τι παίρνουμε από το χέρι μας και με βάση τις εξελίξεις βεβαίως το Συμβουλίο Εξωτερικών θα εξετάσει το ζήτημα και θα πάρει τα μέτρα που θα θεωρήσει σκόπιμα. Γι' αυτό το τρίτο σημείο της μέσης διάταξης ε, θα ήθελα πραγματικά να πω ότι συμφωνώ απολύτως με τους ομιλητές ε, σε ό,τι φορά αυτά που είπαν για την κατάσταση στη Λευκορωσία. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ για το γενναιόδωρο χρόνο που μου χαρίσατε. Θα ήθελα να έχω και περισσότερο, αλλά νομίζω πως ε, απάντησα συνθετικά στις παρεμβάσεις ε, ε, των συναδέλφων για τρία τόσο σημαντικά ζητήματα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Αντιπρόεδρε της Κομισιόν και έπατε εκπρόσωπε. Ολοκληρώνεται λοιπόν εδώ εκείνη συζήτηση και διακόπτεται η σύνοδος ε, μέχρι τις 14 και 15. Καλή όρεξη. Υπότιτλοι

Tag, liebe Kolleginnen und Kollegen. Επανάληψη τη Συνόδου. Ανακοινώσει από την ε, σύσταση τη Επιτροπή ε, Επιτροπής ΕΚΟΝ. Ε, αν δεν υπάρχουν αντιρρήσει, ε, ε όπω δημοσιεύτηκε στην αρχή τη ε, χθεσινή συνεδρίαση και ε, δεν ε, εκφράστηκαν σαν συστάσει. Ε, μέσα στι 24 ώρε και έτσι εγκρίνεται η σύσταση αυτή μαζί με τα συγκριτικά κείμενα. Πρωτού ξεκινήσουμε με τι συζητήσει να ανακοινώσω τα αποτελέσματα του πρώτου γύρου ψηφοφοριών ε, και, του και να ξεκινήσουμε με το δεύτερο γύρο ψηφοφορία. Τα αποτέλεσματα του πρώτου γύρου για την ανθρωπιστική ε, κατάσταση στην Βενεζουέλα και η κατάσταση η ανθρωπιστική. Απορρίφθηκε η πρώτη τροπολογία, η δεύτερη τροπολογία απορρίφθηκε, τροπολογία 3 Απορρίφθηκε. Μια πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση για την ε, καταπολέμηση του ξεπλήματο χρήματο, σχετικά δράση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άλλε εξελίξει. Τροπολογία 1. Απορρίπτεται. Ε, Παράγραφο 3, πρώτο τμήμα εγκρίνεται, δεύτερο τμήμα εγκρίνεται, Παράγραφο 3, τρίτο τμήμα εγκρίνεται. Τροπολογία 6, πρώτο τμήμα απορρίπτεται. Τροπολογία 6, δεύτερο τμήμα απορρίπτεται. Τροπολογία 14 απορρίπτεται. Τροπολογία 15 επίση απορρίπτεται. Παράγραφος 6. Πρώτο τμήμα εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα εγκρίνεται. Παράγραφος 6. Τρίτο τμήμα εγκρίνεται. Παράγραφος 8. Πρώτο τμήμα εγκρίνεται. Παράγραφος 8. Δεύτερο τμήμα εγκρίνεται. Παράγραφο 9 εγκρίνεται. Παράγραφο 13 πρώτο τμήμα εγκρίνεται. Παράγραφο 13 δεύτερο τμήμα εγκρίνεται. Τροπολογία 2 εγκρίνεται. Τροπολογία 16 απορρίπτεται. Τροπολογία 18 εγκρίνεται. Τροπολογία 17, συγγνώμη, εγκρίνεται. 23 παραγραφός πρώτο τμήμα εγκρίνεται. 23 παραγραφός δεύτερο τμήμα εγκρίνεται. Τροπολογία 3 απορρίπτεται. Τροπολογία 8 απορρίπτεται. Παραγραφός 24 πρώτο τμήμα εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα εγκρίνεται. Παραγραφός 27 πρώτο τμήμα εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα εγκρίνεται. Τροπολογία 9 απορρίπτεται. Τροπολογία 10 απορρίπτεται. Παραγραφός 30 πρώτο τμήμα εγκρίνεται. Παραγραφός 30 δεύτερο τμήμα εγκρίνεται. Τροπολογία 11 απορρίπτεται. Τροπολογία 12 απορρίπτεται. Τροπολογία 13 πρώτο τμήμα εγκρίνεται. 13 δεύτερο τμήμα απορρίπτεται. Παράγραφος 40 πρώτο τμήμα καταπίπτει. Επίσης το δεύτερο τμήμα και το τρίτο τμήμα. Τροπολογία 4 απορρίπτεται ε, τη λογική σκέψη ΚΑΠΑ εγκρίνεται και ε, ΧΑ, ε, εγκρίνεται. Και περνάμε τώρα στη δεύτερο γύρο ψηφοφοριών. Τα θέματα που θα ψηφίσουμε θα τα δείτε από την ημερήσια διάταξη και πρώτου ξεκινήσουμε θα ήθελα να δώσω το λόγο στον ε, κύριο Κουσμάρ, ο οποίος το ζήτησε βάσει του 159 άρθρου 4 για την ε, έκθεση του για τα μέτρα για την ε, απασχόληση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για δύο λεπτά έχετε το λόγο. Και από τις 2.30 μέχρι τις 15.45 έχουμε το δεύτερο γύρο ψηφοφοριών. Κύριε Κουσμάου, έχετε το λόγο. Πού βρίσκεται? Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η κρίση COVID-19 είναι μια κρίση που έχει επιπτώσεις πολύ σοβαρές στη δημόσια υγεία, αλλά έχει ήδη ε, επιπτώσεις, ήδη αρχίζουμε να τις νιώθουμε, από την άποψη την οικονομική και την κοινωνική. Και γι' αυτό η έκθεση για τις κατευθύνσεις των πολιτικών απασχόλησης για φέτος έχει μεγάλη διτηρότητα, γιατί στόχο έχει να αρχίσει ήδη να απαντά σε μια οικονομική και κοινωνική κρίση που ήδη γίνεται αισθητή και που ξέρουμε ότι θα επιδεινωθεί στη διάρκεια των επόμενων είναι λοιπόν γι' αυτό πάρα πολύ σημαντικό, εφόσον γνωρίζουμε ότι υπάρχουν αποκλήσει σημαντικέ ανάμεσα στι διάφορε ομάδε όσον αφορά τη λειτουργία τη αγορά-εργασία, αλλά και όσον αφορά τι δημόσιε υπηρεσίε και τι οικονομικέ πολιτικέ, το να έχουμε φτάσει σε τόσο μεγάλη πλειοψηφία και συνένεση για να στηρίξουμε πολιτικές οι οποίες είναι θεμελιώδεις ώστε να προστατευτεί η επασχόληση των όσων έχουν ακόμα απασχόληση αλλά για να προστατευτούν και δημόσιες υπηρεσίες και κοινωνικές υπηρεσίες, κοινωνική πρόνοια για όσους θα χάσουν τη δουλειά τους ε, ε, λόγω αυτής της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης. Γι' αυτό και θέλω να ευχαριστήσω τους συζητητές και συνεισηγητές αυτής της έκθεσης το πνεύμα συνένεσης και συμβιβασμού που επικράτησε και τη συνεργασία των Ευρωπαϊκών, ε, της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Συνδικάτων ε, που θα μπορέσει να συμβάλλει στο να μπορέσει και η Ευρωπαϊκή Ένωση να ανταποκριθεί σε αυτή την κρίση, πράγμα το οποίο έχουμε εκδηλώσει ως επιθυμία μας επανελειμμένα σε αυτή την Ολομέλεια, να μην αφήσουμε κανέναν πίσω. Αυτό ήταν το πνεύμα νομίζω που κίνησε όλους όσους στήριξαν αυτή την έκθεση. Σας ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ, συνάδελφε Μάου Και όπω σα είπα, ξεκινάει ε, ο δεύτερο γύρο ψηφοφορία από 14.30 μέχρι 15.45 με την ε, ίδια διαδικασία που ακολουθήσαμε και σήμερα το πρωί. Και έτσι λοιπόν ξεκινάει ο δεύτερο γύρο ψηφοφορία. Μπορείτε να ψηφίσετε μέχρι 15.45. Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στι 18 και 15. Περνάμε λοιπόν τώρα στις συζητήσεις ε, και επόμενο θέμα στην ημερήσια διατάξη. και ερώτηση προ την ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη στρατηγική για τι χημικέ ουσίε. Με στόχο τη βιωσιμότητα, να σα ε, επισημάνω ότι στη συζήτηση αυτή θα ακούσουμε μόνο του ε, ομιλητέ που έχουν διοριστεί από τι πολιτικέ ομάδε. Και πρώτη έχει το λόγο η συνάδελφο κυρία Σπυράκη. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ελπίζω να είναι εδώ παρούσα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μήπως να περιμένουμε λίγα λεπτά. Ναι, θα περιμένουμε λίγα λεπτά γιατί από ό,τι φαίνεται φτάνει.

Right. Thank Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ για την υπομονή σας. Καλώς ήρθατε, κύριε Επίτροπε. Θα ακούσουμε όμως πρώτα την κυρία Σπυράκη, τη συνάδελφό μας. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε Σεκεβίτσιος, με αυτό το ψήφισμα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητάει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συνεχίσει τις μελέτες για τα χημικά. Τα χημικά βρίσκονται παντού. Βρίσκονται στα τρόφιμα, στο νερό μας, στα ρούχα μας, στα καλλιντικά μας. Βρίσκονται στον ίδιο τον αέρα που αναπνέουμε. Με άλλα λόγια δηλαδή, επηρεάζουν την καθημερινότητά μας. Πρώτη μας προτεραιότητα λοιπόν είναι να αναβαθμίσουμε την προστασία του περιβάλλοντος και των πολιτών. Και γι' αυτό ακριβώς ζητάμε να απαλληφθούν αυτές οι ουσίες που είναι επικίνδυνες για την υγεία και να βρεθούν εναλλακτικά εφόσον αυτό είναι εφικτό. Και ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να φροντίσει να κάνει την αξιολόγηση που χρειάζεται για τους ενδοκρινικούς διαταράκτες. Εμείς επικεντρωνόμαστε εδώ, κύριε Επίτροπε, σε κάτι πάρα πολύ φιλόδοξο να αναβαθμιστεί η ασφάλειά μας από τα χημικά σε ολόκληρο τον κόσμο. Και η ΕΚΑ θα πρέπει να στηρίξει αυτή την πολιτική, καθορίζοντας προδιαγραφές και αριθμιστικά συστήματα με υψηλές προδιαγραφές όσον αφορά την ασφάλεια από τα χημικά. Έτσι θα ενισχυθεί η προστασία και πέρα από τα ευρωπαϊκά σύνορα. Τα χημικά είναι και η βιομηχανία της βιομηχανίας. Υπάρχουν διάφοροι όμιλοι και Γι' αυτό εμείς πρέπει να βοηθήσουμε και να υιοθετήσουμε τη στρατηγική μία ουσία, μία αξιολόγηση επικινδυνότητας και να δώσουμε χρόνο στις βιομηχανίες ώστε να μας προσφέρουν ασφαλή προϊόντα και να δώσουμε επίσης και κίνητρα έτσι στην παραγωγή και την ευρωπαϊκή οικονομία. Να υπάρχει αξιοπρεπής χρηματοδότηση και για να επιταχύνουμε επίσης εναλλακτικές και καινοτόμες λύσεις. Η στρατηγική αυτή θα πρέπει επίσης να διασφαλίσει ότι δεν θα γίνονται χωρίς σοβαρό λόγο δοκιμές στα ζώα πλέον. Όμως, δεν εξαρτώνται όλα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δεν εξαρτώνται όλα από τις Βρυξέλλες ή από την πολιτική βούληση των Βρυξελών. Γι' αυτό και πρέπει να αυξήσουμε και τον βαθμό συμμόρφωσης στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία όσον αφορά τα χημικά και να ζητήσουμε από τις χώρες μέλη να εφαρμόσουν πλήρως το τρέχον πλαίσιο για να προσφέρουν ένα ασφαλές περιβάλλον στους πολίτες, αλλά και με ανταγωνιστικότητα. Χρειαζόμαστε συμμαχίες. Η ΕΚΑ, η ΕΦΣΑ και η ΕΜΑ. Πρώτα απ' όλα λοιπόν πρέπει να αποφύγουμε την επικάλυψη μεταξύ των διαφόρων αυτών ευρωπαϊκών οργανισμών και πρέπει επίσης να διασφαλίσουμε και την κατάλληλη χρηματοδότηση προσφέροντας επιπλέον πόρους. Θα ολοκληρώσω λέγοντας ότι η χημική στρατηγική για τη βιωσιμότητα πρέπει να ευθυγραμμίζεται με τους στόχους της πράσινης ε, ανάπτυξης, το περιβάλλον και τα ψηφιακά. Ενισχύουμε λοιπόν την στρατηγική της ΕΚΑ, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού δηλαδή Χημικών Προϊόντων, προκειμένου να υπάρχει μια πλατφόρμα με τα χημικά και να μπορούμε να ανταλλάσσουμε δεδομένα, οι διάφορες αρχές δηλαδή, και να ενημερώνονται έτσι οι ρυθμιστές, νομοθέτες και οι Επίτροπε, κυρία Πρόεδρε, η στρατηγική για τα βιώσιμα χημικά μπορεί να οδηγήσει τη γενιά μας και τα παιδιά μας σε ένα μέλλον με λιγότερα προβλήματα. Μπορεί να οδηγήσει τη βιομηχανία σε βιώσιμες λύσεις με πολύ χαμηλότερες επιπτώσεις στο περιβάλλον αρκεί τα χημικά προϊόντα που εισάγονται από τρίτε χώρε στην ευρωπαϊκή ένωση να έχουν τι ίδιε. Ακριβώ τι ίδιε προδιαγραφέ με αυτά που παρασκευάζονται και καταναλώνονται στην ευρωπαϊκή ένωση. η αγορά είναι παγκόσμια και το στίχημα για τα βιώσιμα χημικά αφορά τον πλανήτη αφορά τη ζωή μας. ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ. Ε, και τώρα εξ ονόματος της ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπής το λόγο έχει ο Επίτροπος Σιγκεβίτσιος. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμοι Ευρωβουλευτές. Αγαπητοί συνάδελφοι, η σημερινή συζήτηση και το ψήφισμα που θα ψηφίσετε αύριο για την μελλοντική στρατηγική και για τη βιωσιμότητα όσον αφορά τα χημικά είναι κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνετε την ευκαιρία να απαντήσω στα όσα θέτετε στην προφορική σας ερώτηση και να σας ενημερώσω για το πού βρισκόμαστε όσον αφορά τη στρατηγική αυτή. Όπως ανακοινώθηκε στο πρόγραμμα εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2020, έχουμε ενημερώσει πρόσφατα την στρατηγική μας για τα χημικά στα πλαίσια του COVID-19 και συνεχίζουμε να εργαζόμαστε για να εγκριθεί η στρατηγική μας το τρίτο τρίμηνο του, της χρονιάς. Οι πληροφορίες που σας δίνω σήμερα Βέβαια παραμένουν γενικές. Δεν μπορώ ακόμα να μπω σε λεπτομέρειες όσον αφορά την επερχόμενη αυτή στρατηγική. Η χηγημική στρατηγική ενισχύει την βιωσιμότητα και αυτό είναι το πιο βασικό που αναφέρεται στην Πράσινη Συμφωνία και μία από τις κύριες προτεραιότητες του δικού μου χαρτοφυλακίου για φέτος. Όταν εγκρίναμε την Πράσινη Συμφωνία το Δεκέμβριο που μας πέρασε, όλοι συμφωνήσαμε να απαλλαγούμε από το τοξικό περιβάλλον. Η στρατηγική μας ακριβώς ακολουθεί διτή προσέγγιση. Πρώτον, πρέπει να βοηθήσει ώστε να προστατευθούν οι πολίτες και το περιβάλλον καλύτερα απέναντι σε ε, βλαβερά χημικά και δεύτερον, να ενισχύσουμε την καινοτομία ακριβώς υπέρ της ασφάλειας και υπέρ εναλλακτικών λύσεων. Αυτή λοιπόν η διτή προσέγγιση ε, προχωρά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αυτήν ακριβώς έχουν ακολουθήσει οι εργασίες μας από την αρχή όταν αποσαφηνίσαμε ότι θέλουμε να συνδυάσουμε την προστασία του περιβάλλοντος με την υγεία αλλά και να ενισχύσουμε την αντιγωνιστικότητά μας. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συνεργαστούν μεταξύ τους. Αυτό ισχύει βέβαια και για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγώ, οι υπηρεσίες μου, οι συνεργάτες μου ετοιμάζουμε τη στρατηγική αυτή σε στενή συνεργασία με άλλες γενικές διευθύνσεις, με επιτρόπους, τις υπηρεσίες τους, για αυτό το οριζόντιο θα έλεγα θέμα. Στο ψήφισμα το οποίο θα εγκρίνετε εσείς αύριο, επίσης αναγνωρίσετε τον οριζόντιο χαρακτήρα των χημικών. Τονίζετε την ανάγκη για δράση, για ένα ασφαλές περιβάλλον, ασφαλές από τα χημικά, και δεύτερον τονίζεται το σημαντικό ρόλο που παίζει ο τομέας των χημικών προκειμένου να επιτευθούν οι στόχοι της Πράσινης Συμφωνίας, που είναι η κλιματική ουδετερότητα, η ενεργειακή μετάβαση, η πρόθεση ε, της ασφάλειας στον ενεργειακό ε, εφοδιασμό, ψηφιακή οικονομία κτλ. Για άλλη μια φορά θέλω να σας ευχαριστήσω για το έργο σας, για τις τεράστιες προσπάθειες που έχετε κάνει στην εκπόνηση του ψηφίσματος αυτού το οποίο μάλιστα έρχεται σε μια πολύ σωστή στιγμή, γιατί εφόσον εγκριθεί θα μελετήσουμε πάρα πολύ προσεκτικά το περιεχόμενο και θα το λάβουμε υπόψη μας όταν ε, καταλήξουμε όσον αφορά τη στρατηγική μας μέσα τις επόμενες εβδομάδες. Θα λάβουμε επίσης υπόψη μας και τα 400 σχόλια και τις συνεισφορές που έχουμε πάρει από διάφορους φορείς και από πολίτες ε, σε σχέση με τον χάρτη πορεία μας για την στρατηγική μας για τα χημικά. Ε, ξεκίνησε η διαβούλευση ήδη από τις 9 Μαΐου και ολοκληρώνεται αυτό το μήνα. Τώρα θέλω να σα δώσω και κάποια ακόμα στοιχεία όσον αφορά τη στρατηγική μα για τα χημικά και τη βιωσιμότητα. Η στρατηγική μα βασίζεται και θα χτιστεί πάνω σε διάφορε αξιολογήσει ε, για πολιτικέ που έχουν να κάνουν με την νομοθεσία τη Ευρωπαϊκή Ένωση για τα χημικά και, η και κυρίως ε, την ε, δεύτερη απόφαση για το REACH όπως επίσης τις αποφάσεις μας του 19, την ανακοίνωση του 2020 για τους ενδοκρινικούς σου διαταράκτες και τις διάφορες επιλογές που έχουμε για να αντιμετωπίσουμε το θέμα της διεπαφής. Για να πετύχουμε τους κύριους στόχους μας βασιζόμαστε στα εξής στοιχεία. Πρώτον, την ενίσχυση της νομοθεσίας για υψηλής ποιότητας υγεία και προστασία από τα χημικά που προκαλούν βλάβη η ευρωπαϊκή νομοθεσία θα πρέπει να ενισχυθεί και να προστατεύσουμε καλύτερα τις πιο ευάλωτες ομάδες. Να λάβουμε υπόψη μας την συνδυαστική δράση των χημικών και την αντίστασή τους. Δεύτερον, να υπογραμμίσουμε την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα. Πρέπει να δώσουμε κίνητρα για την ανάπτυξη αυτού του παράγοντα ασφάλειας όσον αφορά τη χρήση των χημικών και να περάσουμε σε ένα περιβάλλον με ασφάλεια που να βασίζεται σε νέο σχεδιασμό των χημικών ουσιών. Συγχρόνως, χρειάζεται και είναι πολύ σημαντικό στοιχείο για μας να έχουμε μια ισχυρή ευρωπαϊκή βιομηχανία, έναν βιομηχανικό κλάδο χημικών ισχυρό. Μην ξεχνάμε ότι περιμένουμε και την ανάκαμψη. Έπειτα, πρέπει να υπάρχει στρατηγική αυτονομία στην προμήθεια, τον εφοδιασμό βασικών χημικών που είναι πολύ βασικές τέτοιες χημικές ουσίες πολλές φορές για την υγεία και να λάβουμε υπόψη μας και την ε, πράσινη μετάβαση και τα μηδενικά απόβλητα. Τρίτον, το νομοθετικό μας πλαίσιο είναι μεν ικανοποιητικό για το σκοπό για τον οποίο έχει φτιαχτεί, αλλά είναι περίπλοκο. Και πρόκειται εδώ πέρα για μια πρόκληση που έχουν και οι αρχέ για να το ελέγξουν, αλλά και ο κλάδο για να εφαρμόσει όλε αυτέ τι ρυθμίσει. Πρέπει λοιπόν να απλοποιηθεί και να είναι πιο αποτελεσματικό αυτό το νομοθετικό πλαίσιο. Να ακολουθήσουμε λοιπόν την αρχή που λέει μία ουσία, μία αξιολόγηση επικινδυνότητας και να προσέξουμε και ε, τις αδυναμίες που εντοπίζονται εκεί που διάφοροι κανονισμοί μπερδεύονται μεταξύ τους πρέπει να ενισχυθεί η γνώση όσον αφορά τις χημικές ουσίες που επηρεάζουν την υγεία αλλά και που δημιουργούν απόβλητα. Να ανταλλάσσουμε δεδομένα, πληροφορίες μεταξύ μας αλλά να προσφέρουμε και πληροφορίες ε, στην αλυσίδα εφοδιασμού και για την βιομηχανία. Να φροντίσουμε να καταλήξουμε σε ένα κύκλο χωρίς τοξικές ουσίες. Τέλος, πρέπει να ενισχυθεί η παγκόσμια διάσταση. Είναι πολύ σημαντικό η Ευρωπαϊκή Ένωση να αποτελεί πρότυπο όλο και περισσότερο όσον αφορά την σωστή διαχείριση των χημικών και να ανεβάσει τις προδιαγραφές ασφάλειας για τα χημικά στον κόσμο, την παραγωγή τους και τη χρήση τους. Τέλος, η βιωσιμότητα και η στρατηγική μας αυτή, εφόσον εγκριθεί από το Σώμα των Επιτρόπων, θα επανέλθω και θα σας την παρουσιάσω και προσβλέπω σε στενή συνεργασία μαζί της, προκειμένου να ε, τεθεί σε εφαρμογή αυτή. Γιατί το έργο μας βέβαια δεν ολοκληρώνεται με την έγκριση της στρατηγικής αυτής, Κάθε άλλο. Προς το παρόν θέλω να σας ευχαριστήσω για την προσοχή σας και περιμένω τις απόψεις των πολιτικών σας ομάδων. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε τον Επιτροπό και τώρα να πάρει το λόγο καταρχάς ο συνάδελφος Βάης από το ΕΛΕΚ. Η συνάδελφος Βάης. Το περιβάλλον δεν μπορεί πλέον να αντέξει άλλο. Και ο πληθυσμός αυξάνεται. Θα πρέπει λοιπόν να ρυθμιστούν κάποια πράγματα και εδώ η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μεγάλο ρόλο να παίξει ως παράγοντας για τη βιώσιμη παραγωγή φυτοπροστατευτικών. Αυτό το επεσήμανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο Πράσινο Σύμφωνο. Δεν το ξεχάσαμε από πλευρά του ΕΛΚ. Γι' αυτό λοιπόν στο ψήφισμα αυτό ζητούμε μια στρατηγική για τα χημικά υπέρ της βιωσιμότητας και μάλιστα το συντομότερο δυνατόν. Υπάρχει μια αξιολόγηση ταχαίας ε, ε, εκτήρηξης fast track και θα πρέπει λοιπόν να κινηθούμε με γρήγορους ρυθμούς γιατί οι επιχειρήσεις εξελίσσονται και αναπτύσσουν διάφορα φύτα προστατευτικά και αυτό ωφελεί φυσικά τον κόσμο αλλά η αξιολόγηση και η καταχώρηση γίνεται εκ των υστέρων και έτσι θα πρέπει αυτό το fast track να είναι όντως fast track αυτό το οφείλουμε στον κόσμο Και τα χημικά πάντα κατηγορούνται. Αυτό δεν είναι ούτε σωστό ούτε Ορθό. Η συνάδελφο η κυρία Μαρία Ρένα για 1,5 λεπτό. Στην ανακοίνωση για το Green Deal, η Κομισιόν ανακοίνωσε τη φιλοδοξία τη για μηδενική ρήπανση για ένα περιβάλλον χωρί τοξικέ ουσίε. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ε, ο περιορισμό τη έκθεση σε επικίνδυνε χημικέ ουσίε είναι μεγάλη πρόκληση και ένα κανονισμό σχετικό θα μπορεί να προστατέψει του ε, πολίτε αλλά και το περιβάλλον του κινδύνου που αντιπροσωπούν κάποιε τέτοιε ουσίε. Το Κοινοβούλιο έχει δώσει σαφέ και φιλόδοξο μήνυμα για πλήρη εφαρμογή τη ισχύουσα νομοθεσία καταρχά, αλλά και για μια εξέλιξη τη νομοθεσία σε διάφορε πτυχέ. Είναι αλήθεια πω ε, ισχυρά μέτρα υπέρ τη υγεία και του περιβάλλοντο είναι απαραίτητα και πρέπει οπωσδήποτε να λάβουμε τι ευθύνε μα στο θέμα αυτό. Επιθυμούμε η υγεία να περάσει πριν από τα οικονομικά συμφέροντα ορισμένων βιομηχανιών. Βιώσιμη η η χημεία. Τι σημαίνει αυτό. Συγκεκριμένα κριτήρια για την ορίσουμε. Ε, Αν άνευ αυτών θα είναι μόνο μια έννοια για την οποία θα, την οποία θα χρησιμοποιήσουν οι βιομηχανίε για να υποτίθεται πρασινίσουν την παραγωγή τους εις βάρος των πολιτών. Μια χημική χημεία μάλλον βιώσιμη δεν είναι αυτή που αποδίδει πάντοτε περισσότερα ε, το, ε, μερίδια στους ε, μετόχους, αλλά είναι μια που προστατεύει την βιοπικιλότητα. Περιορισμός των κινδύνων μέσω της αντικατάστασης των πιο επικίνδυνων ουσιών από ασφαλείς εναλλακτικέ λύσεις. Επίσης, θα πρέπει να ενταχθούν εκεί τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά κόστη για τα χημικά που χρησιμοποιούνται. Το κόστος της χημικής βιομηχανίας σε σχέση με την Υγεία είναι 160 δι ετησίω. Εάν αυτό το κόστος το αναλάμβανε η βιομηχανία, μπορώ να σα διαβεβαιώσω πως η αντικατάσταση με εναλλακτικέ ουσίες θα προχωρούσε πολύ πιο γρήγορα. Και προς αυτό πρέπει να κινηθούμε. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ και το... Η κυρία Ρένα μίλησε εξ ονόματο των Σοσιαλιστών και τώρα η κυρία Ρή εξ ονόματο του Ρινιού. Σα ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, το ψήφισμά μα ορίζει ε, το γνώμονα για την ε, βιώσιμη στρατηγική για τα χημικά προϊόντα και γι' αυτό θα περιμένουμε νέα σα πριν το τέλο του χρόνου. Με κοινό στόχο βέβαια, ενίσχυση τη προστασία τη υγεία των πολιτών και του περιβάλλοντο, ένα στόχο ο οποίο είναι φιλόδοξο 71% των χημικών προϊόντων που παράγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρούνται, είναι μάλλον ταξινομημένα στα επικίνδυνα. Ε, επειδή έχουμε ακούσει διάφορα, ξέρουμε πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να ενισχύσει το ρυθμιστικό πλαίσιο, το σε πιο συγκεκριμένα και αυτό είναι καλό νέο. Με ομαδοποιημένη ε, αξιολόγηση των επικινδύνων ουσιών ώστε να επιταχυνθεί η διαδικασία. Κάτι σύντομο. Αυτή η λογική ανά οικογένεια θα πρέπει να εφαρμοστεί και στη διαδικασία περιορισμού για τις επικίνδυνες ουσίες φθαλάτες για παράδειγμα που απαγορεύονται ας πούμε στα παιδικά παιχνίδια αλλά επιτρέπονται αλλού. Επίσης ε, ακούσαμε ότι θα προβλέπονται νέα κριτήρια για τη διαχείριση του κινδύνου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να προστατέψει από του ενδοκρινικού διαταράκτε τα νευροτοξικέ ουσίε, πολλοί εργαζόμενοι καθημερινά εκτίθενται σε διάφορους ε, διαλυτέ ή σε ε, βαρέα μέταλλα. Θα πρέπει επίση να μιλήσουμε για το περφλουάριο που βρίσκουμε στι Ε, ε, στους διάφορους αφρούς ε, ε, είναι ιδιαίτερα επίμονες και αθεκτικές αυτές οι ουσίες είναι πάρα πολύ επικίνδυνες και πρέπει να επιμείνουμε εδώ. Πρόκειται για 5.000 χημικά προϊόντα που ανήκουν σε αυτή τη κλάση. Τον περασμένο Δεκέμβριο η Ολλανδική κυβέρνηση, να θυμίσω, πίεσε για τη συζήτηση αυτή στο Συμβούλιο. Υπάρχει ένα παράθυρο, υπάρχει μια ευκαιρία, πρέπει να την αδράξουμε. Ευχαριστώ. Κύριο Στοβαλιέρη, εξ ονόματος του ε, ID. Κυρία, με συγχωρείτε το Βαλιέρη. Ευχαριστώ. Εγώ βλέπω εδώ διάφορε κρίσιμε ε, σε φάσεις. Πρώτον, ιδεολογική προσέγγιση. Αν θέλουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα για το περιβάλλον, δεν μπορούμε απλώ να δαιμονοποιούμε έναν τομέα ολόκληρο όπω η χημεία, η χημική βιομηχανία που έχει μεγάλη αριστεία, ιδιαίτερα η Ιταλική χημική βιομηχανία και οδηγεί προ βιώσιμε λύσει. Χωρί ρεαλιστική προσέγγιση μπορεί να πλήξουμε την Ευρωπαϊκή και χημική βιομηχανία, όπου απλά θα σημαίνει αυτό μεταφορά τη παραγωγή εκτό Ευρώπη, όπου δεν τηρούνται ούτω ή άλλω τα στάνταρ τα οποία εμεί θέλουμε. Είναι μια μειοπική ε, αντιμετώπιση ει βάρο των εταιριών μα και των εργαζόμενων σε αυτέ. Στόχος ε, ο οποίος θα πρέπει να επιδιωχθεί είναι η στήριξη του τομέα αυτά, όχι μόνο επιβάλλοντας πράσινους φόρους, αλλά και μέσω ε, ε, διαφόρων μέσων που ευνοούν την επιστροφή στην Ευρώπη διαφόρων δυνατοτήτων που έχουμε απλά μεταφέρει εκτός Ευρώπης. Δεν θέλουμε λοιπόν να πλήξουμε ένα στρατηγικό τομέα για ολόκληρη την Ευρώπη, έναν τομέα που αντίθετα θα έπρεπε να στηριχθεί ώστε να μετακινηθεί προς μια παραγωγή ακόμα πιο βιώσιμη. Ευχαριστώ. Επόμενος από τους πράσινους είναι ο συνάδελφος ο κ. Γκίκολτ. Για ένα λεπτό έχει το λόγο. Κυρία Πρόεδρε, Επίτροπε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εδώ δεν ζητάει τίποτα λιγότερο παρά να αλλάξει το παράδειγμα σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Χημική Βιομηχανία για την ε, υγεία μας, για ένα περιβάλλον χωρίς ε, δηλητηρίο και για να υπάρξει αναμόρφωση τη χημική βιομηχανία θα πρέπει να υπάρχει μηδενική ανοχή από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ό,τι αφορά τα επικίνδυνα χημικά. Την εβδομάδα αυτή, κύριε Επίτροπε, δημοσιεύτηκαν αριθμητικά στοιχεία στην Γερμανία. Κάθε πέμπτο παιδί, και αυτό μα ανησυχεί, επιβαρύνεται στην υγεία του από τα χημικά στην καθημερινή του ζωή. Και κάθε ένα παιδί, λοιπόν, στα πέντε επιβαρύνεται σε βάθο χρόνου και ιδιαίτερα χημικά που επιβαρύνουν ε, τις ορμόνες όπως η βυσφενόλη κτλ. θα πρέπει να απαγορευτούν. Θα πρέπει να υπάρχει μια φιλόδοξη τέτοια πολιτική, όχι μόνο για τα παιδιά μας, αλλά γιατί αποτελεί και μια ευκαιρία για την ευρωπαϊκή χημική βιομηχανία. Η καθαρή λοιπόν χημεία τα καθαρά χημικά θα σημαίνουν όχι μόνο καθαρό περιβάλλον και για τη φύση και για τον άνθρωπο, αλλά 1,2 εκατομμύρια δουλειέ στον τομέα τη χημική βιομηχανία. Κύριε Επίτροπε, αναμένουμε λοιπόν μια φιλοδοξή στρατηγική από πλευρά σα. Ευχαριστώ πολύ. Φίωκη, για ένα λεπτό από το ECR. Κυρία Πρόεδρε, ω κοιόδη συζητητή, πρέπει να σα πω ότι δεν συμφωνώ με πολλέ από τι συμβαστικέ τροπολογίε. Ο κανονισμό θα είναι τιμωρητικό, κυρίω για τι μικρέ και μεσαίε επιχειρήσει στα 35 χρόνια που είμαι επιχειρηματίας, ξέρω ότι πρέπει να έχουμε κανονισμούς με υπευθυνότητα που να προστατεύουν την υγεία. Υπάρχουν πολλά επίμαχα ζητήματα. Το νομικό σκέλος, ο κανονισμός θα αλλάξει άλλους κανονισμούς. Το CLP, για παράδειγμα, εκείνο είναι για την ασφάλεια. Κάτι το οποίο θα βάλει τεράστιο βάρος, ιδίως αν συμπεριλάβουμε τις ε, προδιαγραφές για τον συνδυασμό στην ε, επίδραση των χημικών, τον συνδυασμό των χημικών ουσιών. Μερικές φορές δεν μπορούμε να βρούμε βραχυπρόθεσμα εναλλακτικές λύσεις. Γι' αυτό πρέπει να το προσέξουμε πάρα πολύ. Δεν λέω να μην απαγορεύσουμε τις επικίνδυνες ουσίες, αλλά να λάβουμε υπόψη μας ότι πρόκειται για ένα μεγάλο μειονέκτημα σε βάρος των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων πρέπει να βάλουμε στο κέντρο τις επιχειρήσεις. Ενώ δεν λέμε τίποτα, ούτε λέμε τίποτα τι γίνεται για τους ιδιώτες. Η κυρία Χάζελκαμπ. 1,5 λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Επίτροπε, δικαιούμαστε ένα μη τοξικό περιβάλλον. Τι θα κάνουμε όμως για να το πετύχουμε αυτό. Πάρα πολλοί άνθρωποι πεθαίνουν νέοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι μόνο, επειδή είναι θύματα των χημικών ουσιών. Εκτίθεται δηλαδή σε επικίνδυνες χημικές ουσίες στην εργασία τους. Υπάρχουν στοιχεία στο οικοσύστημά μας, υπάρχουν τα φυτοφάρμακα, τα οποία πολλές φορές οδηγούν στο θάνατο. Επίσης υπάρχει έκθεση στους ενδοκρινικούς διαταράκτες τα παιδιά παίζουν με παιχνίδια τα οποία περιέχουν επικίνδυνες ουσίες, τοξικές. Στα εργαστήρια επίσης χρησιμοποιούνται πολλές φορές ε, φτηνές και παροχημένες πρακτικές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση βέβαια έχει αξιοπρεπή νομοθεσία για την προστασία από τις πιο επικίνδυνες χημικές ουσίες. Παρόλα αυτά, ε, τέτοιες χημικές ουσίες εξάγονται σε άλλα μέρη του κόσμου. Χαίρομαι που μας υποσχέθηκε η Επιτροπή μηδενικές ε, εκπομπές ε, ρηπογόνων ουσιών. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σας ζητάει να κάνετε κι άλλα, να φροντίσετε για τη βιωσιμότητα των ε, χημικών και να μας ακούσετε δεν περισσεύει χρόνος. Σας παρακαλούμε να μας προσφέρετε αυτόν τον ε, ελεύθερο από τοξικά, από τοξικές ουσίες κόσμο όσο γίνεται πιο γρήγορα. Ευχαριστώ πολύ. Και στο τέλος έχει πάλι το λόγο ο κύριος Επιτραπός, ο κύριος Σιγκεβίτσιος. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αξιότιμοι βουλευτές, συνάδελφοι, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τις παρεμβάσεις σας. Να σας ευχαριστήσω και για τα πολύ σημαντικά στοιχεία τα οποία θέσατε, πολλά εκ των οποίων αποτυπώνονται και στο ψήφισμα, το οποίο θα εγκρίνεται αύριο. Σημειώνω. Σημειώνω δεόντως όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία μου δώσατε και όλε τι απόψει που εκφράσατε και τα οποία θα τα λάβετε υπόψη, θα τα λάβουμε και εμεί υπόψη όταν θα οριστικοποιήσουμε τη στρατηγική τις επόμενες εβδομάδες. Ο στόχο που έχω θέσει είναι σαφέστατο. είναι να δημιουργήσουμε ένα όραμα για ένα συνεκτικό πλαίσιο, ένα πολύ συγκεκριμένο σχέδιο δράση για τη συνεργασία όλων των εμπλεκομένων φορέων. Η κρίση COVID-19 έχει καταδείξει σαφώς την ανάγκη να δράσουμε πιο γρήγορα στον τομέα των χημικών. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε την προστασία των πολιτών μας, να υποστηρίξουμε την κοινωνικο-οικονομική ανάκαμψη της ευρωπαϊκής Βιομηχανία και να προωθήσουμε τη στρατηγική πολιτική μας για τους τομείς εκείνους και τα χημικά εκείνα τα οποία είναι σημαντικά για την κοινωνία και την υγεία. Αυτή η στρατηγική θα αποτελέσει ένα πρώτο βήμα για την φιλοδοξία μηδενική ε, ρήπανση. Ε, θα ακολουθούν και το σχέδιο δράση το 2021. Θα συμπληρωθεί και με άλλε δράσει από το Πράσινο Σύμφωνο, την προστασία τη βιοπικιλότητα και στην τελική ανάλυση το μέλλον και την ε, συνεισφορά που θα είναι τεράστια στην κυκλική οικονομία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει τονίσει ότι την απασχολούν το θέμα της ψηφιακής μετάβασης, η καταπολέμηση του καρκίνου και αυτό έχει οριζόντιο χαρακτήρα. Θα χρειαστούν λοιπόν κοινέ προσπάθειε και επικοδομητική συνεργασία από όλου του πλευ... Ε, φορεί. Υπολογίζω στην υποστήριξή σα και προσβλέπω στην ε, συνεχή στενή συνεργασία μαζί σα σε ό,τι αφορά την πολιτική αυτή. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Επίτροπο και έτσι ολοκληρώθηκε η συζήτηση αυτή, η ψηφοφορία για τις ε, τροπολογίες θα λάβει χώρα σήμερα και το τελικό κείμενο θα ψηφιστεί αύριο. Περνάμε στο επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη λοιπόν. Η δήλωση του Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, για την ενίσχυση ε, τη πολιτική για τη διαδικασία ένταξη των Ρωμά στην Ευρώπη για την επόμενη δεκαετία δεν επιτρέπονται μπλε κάρτε. Να σα επισημάνω, ούτε μπορεί να ζητήσουμε το λόγο οι συνάδελφοι. Να δώσουμε το χρόνο που χρειάζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να πάρει τη θέση της. Um... Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, λέει η πρόεδρο, όλου εκείνου που καθαρίζουν και απολυμμένουν το χώρο εργασία μα καθ' όλη τη διάρκεια τη ε, συνεδρίαση τη Ολομέλεια. Και θα ήθελα στο σημείο αυτό να δώσω το λόγο στο Συμβούλιο, στον κύριο Υπουργό, κύριο Αξιότιμη κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές. Σήμερα που μιλάμε για την κοινωνική κατάσταση των Ρωμά, μιλάμε για 10 12 εκατομμύρια ανθρώπους στην Ευρώπη. Μιλάμε για 6 εκατομμύρια πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πολλοί, υπερβολικά πολλοί από αυτούς ζουν σε καθεστώς ε, φτώχειας, απόλυτης ένδυας και βρίσκονται υπό τραγικούς όρους. Ε, έχουν περάσει περίπου 10 χρόνια από τότε που καταρτήσαμε και συμφωνήσαμε τη στρατηγική για τους Ρωμά και κάποιοι από εσά ήδη τότε συμμετείχαν στη διαδικασία αυτή όταν ξεκίνησε αυτή η διαδικασία το 2011 και μάλιστα με μεγάλη υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έκτοτε κυρίες και κύριοι βουλευτές, έχουν περάσει περίπου 10 χρόνια, σχεδόν 10 χρόνια και δυστυχώς διαπιστώνουμε ότι τα αποτελέσματα τα οποία θέλαμε να έχουμε πετύχει ως τώρα μας έχουν απογοητεύσει. Αυτά μας αναφέρει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό τονίζετε και εσείς στα ψηφίσματά σας, ε, στο ψήφισμά σας της προηγούμενης χρονιάς, αγαπητοί βουλευτές. Α, διαπιστώνουμε δυστυχώς ότι τα πράγματα πάνε αργά πολύ αργά, υπερβολικά αργά. Και αυτή η καταπολέμηση της φτώχειας η οποία μαστίζει γενιά, γενιές ολόκληρες ε, των Ρωμά και σε ό,τι αφορά την περιθεωποίηση των Ρωμά και των Σύντη. Το λέω αυτό και ως εκπρόσωπος μιας χώρας η οποία πριν από δεκαετίες ε, σε καθεστώς φασισμού Ε, προκάλεσε θύματα, 500.000 θύματα, αθώους, άνδρες, γυναίκες και παιδιά. Το θέμα λοιπόν της ε, ίσης ε, συμμετοχή στην κοινωνία των Ρωμά είναι ένα θέμα που παίρνει χρόνο. Και ναι, θα έπρεπε να έχουμε πετύχει πολλά παραπάνω τώρα. Και ναι, δίχως αμφιβολία. Και μπορούμε και πρέπει στο μέλλον να καταβάλουμε μεγαλύτερες προσπάθειες. Ωστόσο, κυρίες και κύριοι βουλευτές, έχουμε και καλές ειδήσει να αναφέρουμε. Όπως αναφέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στον τομέα της εκπαίδευσης ε, έχουμε σημειώσει τη μεγαλύτερη πρόοδο. Για παράδειγμα, τα κρατημέλη λαμβάνουν μέτρα προκειμένου να εγκαταλείπουν όλο και λιγότερα παιδιά Ρωμά το σχολείο και να υπάρχει όλο και πιο πολύ πρόσβαση των ε, Ρωμά και των μικρών παιδιών στη φύλαξη και σε ό,τι αφορά την υποχρεωτική εκπαίδευση. Προφανώς και αυτό έχει τεράστια σημασία, αγαπητοί βουλευτέ Τον 21ο αιώνα η διακριτική μεταχείριση και τα ρατσιστικά σχόλια και προκαταλήψεις θα πρέπει να πάρουν ένα τέλος. Η διακριτική μεταχείριση και η ρατσισμός κατά των Αθηγανών θα πρέπει να σταματήσει. Αν θέλουμε να κοιτάμε τον εαυτό μας στον καθρέφτη και αν θέλουμε να γινόμαστε αντιληπτοί ως ε, δίκαιοι πολιτικοί Χρειαζόμαστε όμως και μια συνεκτική πολιτική για την καταπολέμηση των κοινωνικών ανισοτήτων. Η ακραία φτώχεια η οποία μας θέσει γενιάς μετά και γενιές έχει πραγματικά πολύ σοβαρέ συνέπειε σε ό,τι αφορά την υγεία, σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση, σε ό,τι αφορά τη στέγαση και την απασχόληση. Χρειαζόμαστε επιτέλου ένα σχέδιο που θα καλύψει όλου αυτού του τομέ παράλληλα. Μόνο έτσι θα σταματήσει ο φαύλο κύκλο τη περιθωριοποίηση και φυσικά θα πρέπει οι εκπρόσωποι των Ρωμά να συμμετέχουν στη διαδικασία αυτή. Όχι όμως κάπου στο περιθώριο, επίσης όρις, με ένα διάλογο σεβασμού, χωρίς προκαταλήψεις. Όταν δεν έχει κανείς πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη, σε ένα κανονικό σχολείο, αν κανείς ε, δεν έχει ε, στέγαση, δεν έχει δουλειά, πώς αυτός ο άνθρωπος μπορούμε να φανταστούμε ότι μπορεί να εκπληρώσει τα όνειρά του, πώς μπορεί να αναπτύξει τις ικανότητές του, τα ταλέντα του στην κοινωνία μας. Το θέμα της υγείας, του καιρού της πανδημίας COVID-19 προφανώς είναι όλο και πιο σημαντικό. Και οι Ρωμά, όπως και όλοι οι υπόλοιποι, θα πρέπει να έχουν ίση πρόσβαση στις βασικές υπηρεσίες υγειονομικής περιθαλψη και σε ειδικέ υπηρεσίες υγείας. Σε ό,τι αφορά τις νέες πρωτοβουλίες της οποίας ε, εξήγηλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Οκτώβριο, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γιατί το θέμα αυτό πάντα το βάζετε στην ημερήσια διάταξη. Διαρκώ. Και έτσι όχι μόνο συμβάλατε τότε το 2011 στην κατάρτιση του δεκαετούς αυτού σχεδίου και πλαισίου, αλλά και τα τελευταία χρόνια καταφέρατε τακτικά να επισημαίνετε το θέμα αυτό το οποίο χρήζει περαιτέρω προσπάθειας και προσοχής. Αγαπητοί, αξιότιμοι κύριοι βουλευτές, ε, αγαπητή κυρία Επίτροπε, φανταστείτε ένα παιδί, Ρωμά, το οποίο γεννήθηκε τότε, όταν αποφασίστηκε το πλαίσιο αυτό για τους Ρωμά, το 2011 δηλαδή. Σε ένα έτος ε, μεγάλων σχεδίων, μεγαλοπίβολων και μεγάλης ελπίδας. Σήμερα αυτό το παιδί θα έχει κλείσει τα εννιά Και δυστυχώς κατά πάσα πιθανότητα δεν έλαβε την ευκαιρία την οποία εμείς οι πιο πολλοί τη θεωρούμε αυτονόητη. Την οποία τη θέλουμε για τα παιδιά μας για τα εγγόνια μας. Η ακραία φτώχεια, η διακριτική μεταχείριση, ο κοινωνικός αποκλεισμός δεν είναι μόνο λέξεις και αφηρημένες έννοιες. Είναι η πραγματικότητα, η τραγική πραγματικότητα που ζουν στην Ευρώπη και σε όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι άνθρωποι αυτοί. Πρόκειται για άδικα εμπόδια τα οποία εμποδίζουν και αφαιρούν την ευκαιρία για αξιόπρεπη διαβίωση από όλους τους Ρωμά. Ας σκεφτούμε λοιπόν αυτό το 9χρονο παιδί Ας σκεφτούμε τα 6 εκατομμύρια πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενήλικοι και παιδιά. Αγόρια και κορίτσια. Γυναίκες και άντρες. Τι προοπτικές θα έχουν τα επόμενα χρόνια αυτοί οι άνθρωποι. Δεν μπορούμε να τους αφήσουμε ξεκρέμαστούς. Το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι σύμμαχοι σε ό,τι αφορά την συμπερίληψη των Ρωμά στην κοινωνία και είμαι πεπισμένος ότι αυτή η συμμαχία θα συνεχιστεί. Τα κράτη-μέλη διαθέτουν τις βασικές ικανότητες που χρειάζονται, αλλά εμείς ως όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούμε να συνδράμουμε, μπορούμε να βοηθήσουμε προκειμένου αυτός ο μακρύς και δύσβατος δρόμος να έχει επιτυχή έκβαση. Έχουμε και νομικέ διατάξει σε ευρωπαϊκό επίπεδο που απαγορεύουν την διακριτική μεταχείριση όλων των εθνοτικών ομάδων και το Ρωμά προφανώ. Αγαπητοί βουλευτέ. Πρόκειται για ένα έτος κλειδί για την στρατηγική για τη συμπερίληψη των Ρωμά και πολύ φοβάμαι ότι αυτό το έχετε ακούσει πολλέ φορέ. Δεν είναι όμω και ένα λόγια. Το θέμα είναι να υπάρξει συγκεκριμένη δράση. Και αν υπομονώ να ακούσω αγάπητη Ελένα Ντάλι πώ θα διαμορφωθεί το πακέτο το οποίο θα προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και προτείνω να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μα προκειμένου στην Προεδρία μα να ψηφιστεί το πακέτο αυτό. Ας ε, αντλήσουμε δύναμη λοιπόν από τις ευρωπαϊκές αξίες της δικαιοσύνης και της αλληλεγγύης. Η Ευρώπη ήταν, είναι και θα είναι το όνειρο της αλληλεγγύης, το όριμο της αξιοπρέπειας και της ισότητας και της δικαιοσύνης, αλλά πάνω απ' όλα για τους Σύντη και τους Ρωμά, τους οποίους ε, τιμούμε με τέτοιο τρόπο σήμερα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Υπουργέ Ρότ. Και τώρα το λόγο έχει εξ ονόματο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή η Επιτροπή κυρία Τάλη. Ευχαριστώ, Υπουργέ Ρότ, για αυτήν την ε, ε, συναισθηματική εισήγηση σε αυτή την πολύ σημαντική συζήτηση. Αξιότιμοι κύριε Βερβουλευτέ, σας ευχαριστώ και εσάς που βάλατε αυτό το θέμα στη σημερινή μερίσια διάταξη. Σας ευχαριστώ όλους σήμερα εδώ την κυρία Λίβια Γερόκα, τον Ρωμαίο Βλάνση και τον κύριο Πίτερ Πόλα και όλος ιδιαίτερος για την ορατότητα που παρέχουν στην κοινότητα των Ρωμά, την προσήλωσή τους και το ακούραστο έργο τους ε, για την ε, πολιτική για τους Ρωμά, την ε, συμμετοχή τους και την ένταξή τους, αλλά και για τη διοργάνωση της σημερινής συζήτησης. Επίσης, επαναλαμβάνω τις ευχαριστίες μου στα μέλη που είναι παρόντα σήμερα εδώ για ε, την ε, αδιάλειπτη στήριξη τους ε, προς την ατζέντα της ένταξης των Ρωμά και της ισότιμης συμμετοχής τους. Θα παραθέσω την καγκελάριο Μέρκελ και την ομιλία της τη χθεσινή εδώ στην αίθουσα της Ολομέλειας που είπε «Τα ανθρώπινα και τα πολιτικά δικαιώματα ο απαραβίαστος χαρακτήρας της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, η ελευθερία, η ατομική, η προσωπική, η πολιτική και η κοινωνική ανάπτυξη, η προστασία κατά των διακρίσεων, και της παράβλεψης, η ισότητα, η ισότητα την οποία όχι μόνο κάνεις διεκδικεί αλλά υλοποιείται, μπαίνει σε εφαρμογή. Αυτές είναι, αυτά είναι τα ηθικά και πολιτικά θεμέλια επί των οποίων εδράζεται η Ευρώπη. Αυτά είναι τα δικαιώματα που ισχύουν για όλους δεν ισχύουν σε ορισμένους περισσότερο και σε άλλους λιγότερο δεν ισχύουν σε ορισμένους πάντοτε ενώ σε άλλους που και που ισχύουν τελεία. Αυτή είναι η υπόσχεση της Ευρώπης που πρέπει να εγγυηθούμε ότι οι πολίτες να είναι πραγματικά ελεύθεροι να ζήσουν τις θρησκευτική, τη θρησκευτική τους πίστη, τις πολιτιστικές, οι πολιτικές τους επιπιθήσεις, να μπορούν να τηρούν τις δικές τους ιδέες για την ευτυχία και την καλοζωία. Αξιότιμοι κύριοι βουλευτές λοιπόν, με αυτήν την παράθεση της καγκελαρίου Μέρκελ στην καρδιά μας και στο μυαλό μας θα μιλήσω τώρα για την πραγματικότητα των Ρωμά που είναι το σημερινό αντικείμενο της συζήτησης. Όπως γνωρίζετε, οι Ρωμά που ζουν σε περιθωριοποιημένες κοινωνίες είναι κάποιες από τις πιο ευάλωτες ομάδες που χτυπήθηκαν σκληρότερα από την πανδημία κοροναϊού. Οι ήδη υπάρχουσες ανισότητες ε, επιβεβαιώθηκαν. Διαρκείες ανισότητες, διακρίσεις και αποκλεισμό έχουν καταστεί πιο ορατές. Η Επιτροπή γνωρίζει αυτό το γεγονός ε, και μάλιστα μέσω συγκεκριμένων επικοινωνι... Ε, ανακοινοθέντων έχουμε κάνει ό,τι μπορούμε ώστε να προσφέρουμε ταχεία παρέμβαση. Θα παραμείνουμε σε παγρύπνηση και θα συνεχίσουμε να παρεμβαίνουμε με τη βάση των αναγκών σύμμορφα με το καθήκον μας και την ευθύνη μας. Η Κομισιόν εξ αρχής ανταποκρίθηκε με το ξέσπασμα της κρίσης για, μαζί με τους επιτρόπους Κυριακίδη και Σμιτ έγραψα στους υπολείπους και τόνισα την ανάγκη λήψης ειδικών μέτρων για τις πιο ευάλωτες ομάδες στο πλαίσιο της κρίσης του κοροναϊού. Επίσης είδαμε να δημορφώνονται άμεσα κάποια μέσα για άμεση ανταπόκριση στην κρίση που μπορούν να προσφέρουν στήριξη σε ευάλωτες ομάδες όπως η Ρωμά. Κανείς και σίγουρα όχι οι πιο ευάλωτοι δεν θα πρέπει να φέρουν περισσότερα από το μερίδιο που τις αντιστοιχεί ε, στο πλαίσιο αυτής της πανδημίας. Η κοινότητα των Ρωμά όχι μόνο υποφέρει από τις επιπτώσεις στην υγεία και την οικονομία ε, λόγω αυτής της κρίσης και σε ορισμένα από κράτη-μέλη και πραγματικά με λυπή που το λέω αυτό, οι Ρωμά έχουν επίσης ε, προβληθεί ως απειλή για τη δημόσια υγεία στη διάρκεια της κρίσης και αυτό είναι κάτι ντροπιαστικό. Η πανδημία τόνισε βαθιά ριζωμένες ε, διακρίσεις και μίσος κατά αυτών των κοινοτήτων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταδικάζει στεναρά όλες τις μορφές στιγματισμού, ε, εξωστρακισμού ε, των Ρωμά. Όλα αυτά είναι αντίθετα με τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατά των βασικών αρχών της δημοκρατίας μας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει νομικά δεσμευτικά εργαλεία στη διάθεσή της για να καταπολεμήσει τις διακρίσεις και αυτές που βασίζονται σε φιλετική ή εθνοτική προέλευση η απόφαση του Συμβουλίου για την καταπολέμηση ορισμένων μορφών ρατσισμού και ξενοφοβίας είναι το εργαλείο για να καταπολεμηθεί το έγκλημα μίσους, ε, ο αντιθικανισμός, ε, ο, φιλετικός ε, ρατσισμός και λόγος. Αυτά αντιμετωπίζονται σε βασικές ε, ε, πτυχές της καθημερινής ζωής. Η Ρωμά είναι προστατευόμενη μειονότητα και καλύπτονται από αυτά τα νομικά εργαλεία και έχουμε καθήκον να τα επιβάλλουμε. Γνωρίζουμε όμως επίσης ε, ότι η νομοθεσία είναι θετική. Τώρα, το πόσο αποτελεσματική είναι όμως στην πραγματική ζωή είναι κάτι διαφορετικό. Από μόνη της η νομοθεσία δεν αρκεί ποτέ και σε κανένα τομέα. Και έτσι πρέπει να κάνουμε πολύ περισσότερο περισσότερα. Ε, παρακολουθούμε στενά τη συμμόρφωση των κρατών μελών με την οδηγία. Τρεις διαδικασίες κατά παράβαση είναι υπό εξέλιξη κατά κρατών μελών και σχετίζονται με την ε, διάκριση ενάντια στα παιδιά Ρωμά, στα, στα σχολεία αλλά και ε, ενάντια σε παιδιά Ρωμά με πνευματικές δυσκολίες ή αναπηρίες. Ε, θέλουμε να σταματήσει αυτή η κατάσταση και δεν θα διστάσουμε να ξεκινήσουμε νέες διαδικασίες κατά παράβαση αν διαπιστωθεί τέτοια ανάγκη. Η η υπέρβαση των διακρίσεων και του αποκλεισμού των Ρωμά χρειάζεται μακροπρόθεσμη πολιτική. Όπως ανακοίνωσα, έχουμε προετοιμάσει μια στρατηγική, το στρατηγικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ισότητα, την ένταξη και τη συμμετοχή των Ρωμά μέχρι το 2030. Αυτή η στρατηγική θα αντικατοπτρίζει και τις νέες ανάγκες που προκύπτουν λόγω της κρίσης ε, του κοροναϊού και αφορούν ε, τις περιθωριοποιημένες κοινότητες ε, των Ρωμά. Θα παρουσιαστεί αργότερα φέτος. Θέλουμε ισχυρή, φιλόδοξη και ολοκληρωμένη στρατηγική. Πιστεύω ακράδαντα ότι αν βασιστούμε στα πορίσματα της αξιολόγησης του πλαισίου που πήγαινε μέχρι το 2000 θα μπορέσουμε να προάγουμε την ισότητα για τους Ρωμά καταπολεμώντας το αντιθυγκανισμό και του διακρίσεις ενώ ταυτόχρονα θα προωθούμε την οικονομική και κοινωνική ένταξη των ανθρώπων αυτών. Πρέπει να αντικατοπιστεί καλύτερα η διαφορετικότητα ανάμεσα στους Ρωμά και να δώσουμε ε, δυνατότητες περισσότερες για τη συνεργασία με τις κοινωνίες, κοινότητες των Ρωμά, την, την κοινωνία των πολιτών των Ρωμά και άλλους φορείς. Να προωθήσουμε την ισότητα των Ρωμά και την ένταξή τους σε όλες τις βασικές μας πολιτικές. Το να εργαστούμε προς βελτιωμένη συλλογή στοιχείων και παρακολούθηση της πρόοδου μέσω δικτών και σαφών στόχων ώστε να εξασφαλίσουμε πραγματική πρόοδο και να προωθήσουμε τις πολιτικές αυτές. Οι άμεσες συνέπειες αυτής της πανδημίας στις κοινότητες των Ρωμά έχουν τον, ε, δίνει ακόμη περισσότερο την ανάγκη για ανανεωμένη και ισχυρή ε, δέσμευση από όλου τους φορείς ώστε να προχωρήσουμε περισσότερο από κοινού με πλήρη ε, συμμετοχή και των ίδιων των Ρωμά. Χρειάζονται τη δική σας, τη δική μου και τη δική μας ακούραστη δέσμευση, προσήλωση και σκληρή δουλειά. Είμαι βεβαία ότι από κοινού θα μπορέσουμε να κάνουμε πολλά για να αλλάξουμε και να βελτιώσουμε τις κοινωνίες μας. Από κοινού μπορούμε να πετύχουμε περισσότερα, περισσότερη ένταξη, περισσότερη ισότητα, περισσότερη δικαιοσύνη, περισσότερη συμμετοχή για τις κοινότητες των Ρωμά σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε την κυρία Πετροπό. Και τώρα εξ ονόματος του ΕΛΚ το λόγο έχει ο συνάδελφος κύριος Πόλακ για 1,5 λεπτό. Ε, ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο αξιότιμοι συνάδελφοι. Θα πρέπει να παραδεχτούμε στην παρούσα φάση ότι τα τελευταία, τις τελευταίες δύο προγραμματικές περιόδους ε, έχουμε σημειώσει μόνο περιορισμένη επιτυχία σε ό,τι αφορά και το τεράστιο δαπάνε που έγινε τον Οκτώβριο, εκινήθηκε μια τεράστια πρωτοβουλία σε ό,τι αφορά την πολιτική για τους Ρωμά μέχρι το 2030. Η πρωτοβουλία θα πρέπει να βασίζεται στην επίτευξη αποτελεσμάτων σε ό,τι αφορά και την ε, αποτελεσματικότητα σε σχέση με τα δαπανηθέντα κονδύλια. Θα χρειαστεί να πετύχουμε λοιπόν στόχους ε, στα κράτη-μέλη σε ό,τι αφορά τα προβλήματα οικονομικά τα οποία εμβαθύνονται. Θα πρέπει να επικεντρωθούμε λοιπόν στα κράτη-μέλη με μεγάλο πληθυσμό Ρωμά όπου τον 21ο αιώνα οι Ρωμά βρίσκονται να ζουν υπό θλιβερές συνθήκες. Χρειάζεται λοιπόν διαρκή συμμετοχή των Ρωμά στη διαδικασία αυτή. Όλα αυτά θα πρέπει να είναι βασικό συστατικό οποιασδήποτε πολιτικής. η Ρωμά είναι Ευρωπαίοι πολίτες και αποτελούν τεράστιο οικονομικό και ανθρώπινο δυναμικό. Θα πρέπει να ομολογήσουμε ότι οι Ρωμά στην ε, Ευρώπη αντιμετωπίζουν ένα θεσμικό ρατσισμό, ακόμα και τα παιδιά. Θα πρέπει λοιπόν εξ ονόματος όλων των πολιτικών ομάδων να δραστηριοποιηθούμε. Κάποιες πολιτικές ομάδες μπλόκαραν ε, λοιπόν τη λήψη ε, αποφάσεων. Πρώτο γεγονός ότι ήταν, ε, μιλάμε για τους Αφροαμερικανούς στην Αμερική, καταδικάζουν το ρατσισμό. Θα πρέπει λοιπόν να καταπολεμήσουμε τέτοια φαινόμενα στην Ευρώπη. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πόλεκ. Εκ μέρους των Σοσιαλδημοκρατών τώρα η κυρία Ινσύρ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Πράγματι πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες δεν εφαρμόζουν όλες τις ευρωπαϊκές απαιτήσεις κάθε φορά και η Ευρώπη έχει την ευθύνη να τις πιέσει και να πιέσει την κοινωνία μας. Μιλάμε για διακρίσεις που γίνονται στους χώρους εργασίας, στην στέγαση, στα σχολεία και στο διάλογο με κυβερνητικές αρχές. Οι νέοι και κυρίως οι γυναίκες εκτίθενται συχνά και υποφέρουν στις κοινωνίες μας. Και η κατάσταση βέβαια έχει επιδεινωθεί τώρα με τον κορονοϊό. Πιστεύω ότι οι Ρωμά, γενικά μιλώντας, αξίζουν περισσότερο, αξίζουν καλύτερα, φτάνει πια. Πρέπει να σταματήσει αυτός ο ρατσισμός και να έχουμε μία κοινωνία όπου όλοι να είναι ίσοι. Δεν έχουμε περιθώρια για διακρίσεις στις κοινωνίες μας, φτάνει πια. Είναι σαφές ότι πρέπει να υιοθετήσουμε στρατηγικές, αλλά χρειαζόμαστε και μετρήσιμους στόχους. Πρέπει να αναλάβουμε δράση και όχι να σχεδιάζουμε μόνο και να έχουμε σχέδια προς εφαρμογή. Ευχαριστούμε. Τώρα το λόγο έχει η κυρία Ντόνατ. Η πολιτική αυτή λοιπόν των τελευταίων ε, δεκαετιών κόστησε ολόκληρε δεκαετίε στην Ευρώπη γιατί η στρατηγική δεν συνέβαλε τελικά στη μείωση και στον τερματισμό του ρατσισμού κατά το Ρωμά. αντιθέτω. εξακολουθούν λοιπόν τα παιδιά των Ρωμά να μην μπορούν να βγουν από το τέλμα της φτώχειας. Και πρόκειται αυτό για απώλεια όλων μας. Η διακριτική αυτή μεταχείριση και ο αποκλεισμό στα σχολεία και στην αγορά εργασία οδηγεί στην κατάσταση όπου τελικά εκατοντάδε χιλιάδε βρίσκονται χωρίς δουλειά στην Ευρώπη και αυτό είναι εις βάρος όλης της ε, κοινωνίας. Θεωρήσαμε ότι με τη στρατηγική θα επιληθούν από μόνο τα προβλήματα, αλλά θεωρώ ότι η ένταξη είναι μια στρατηγική η οποία δεν μπορεί να επιτευχθεί μόνο με κονδύλια. Χρειάζεται μια ανθρωπι... ανθρώπινη πολιτική, μια ανθρώπινη στρατηγική, η οποία θα υλοποιηθεί από κοινού με τη Ρωμά η Ουγγρική Προεδρία τότε έθεσε αυτή τη στρατηγική για τους Ρώμα πριν από 9 χρόνια και βλέπουμε σήμερα ότι η Ουγγρική κυβέρνηση κάνει ότι περνάει από το χέρι της για να έχει ίδια κέρδος. Και στην Ουγγαρία λοιπόν είναι τραγική αντιμετώπιση των Ρωμά και αυτό αποτελεί τμήμα των πραγματικών δηλώσεων της κυβέρνησης. Δεν μπορούμε όμως να επιτρέψουμε την περιθωριοποίηση. Θα πρέπει μαζί να προσπιστούμε τους Ρωμά. Ευχαριστούμε την κυρία Ντόνατ. Η Αναλίζα Ταρντίνε τώρα από τους ID. Ευχαριστώ. Η υποδοχή θα πρέπει πάντοτε να γίνεται με βάση του νόμου και να συνδυάζεται όταν αυτό είναι απαραίτητο με την καταστολή των καταχρήσεων. Και με τα λόγια του Πάπα Ιωάννη Παύλου Δευτέρου η αίσθηση ένταξη είναι μια διαδικασία που συναποτελείται από καθήκοντα και από δικαιώματα αλλά και από καθήκοντα. Δυστυχώ, η υποδοχή αυτή τη στιγμή σημαίνει εγκατάλειψη των αρχών μα και του στυλ ζωή μα. Δηλαδή, το να υποδεχτεί τον άλλον να σημαίνει ότι αλλάζει αλλάζεις εσύ ο ίδιος. Αυτό συμβαίνει με τους Ρωμά στη χώρα μας. Έχουν δημιουργήσει εγκληματικά δίκτυα, δεν εγγράφονται πουθενά, εκμεταλλεύονται τα ίδια τους τα παιδιά τους, υποχρεώνουν να ζητιανεύουν και ε, δεν τα στέλνουν ούτε καν στο σχολείο. Εκεί πρέπει να παρέμβει το κράτος ε, καταπολεμώντας την υποβάθμιση των Ρωμά που ζουν στις πόλεις μας. Στάνει η υποκρισία ότι σέβονται τους κανόνες, τους νόμους και τις πολιτιστικές μας αξίες. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Ταρντίνο. Τώρα έχει το λόγο ο κύριος Φράντς. Για δύο λεπτά. Αγαπητοί συνάδελφοι, αυτή η συζήτηση για την κατάσταση των Ρωμά και τη συμπερίληψη αυτών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο χρειάζονται καταπηγόντω. Ο COVID-19 κατέστησε σαφή τα πράγματα σε ό,τι αφορά του ε, Βλέπουμε ε, βία από τους ε, αστυνομικού κατά την Ρώμα στην Σλοβακία και στη Ρωμανία. Βλέπουμε ε, να έχουν άνθρωποι οι οποίοι ήταν σε κλεισμό προηγουμένη ε, πρόσβαση σε τρόφιμα και στην Γερμανία βλέπουμε βία κατά τον Σύντη και τον Ρώμαν και στο Βερλίνο ε, συζητιέται ε, η απόσυρση ενός μνημείου για τον Σύντη και τους Ρώμα λόγω μιας γραμμής τραμ καινούριας. Είμαι εισηγητής για την έκθεση αυτή στο Κοινοβούλιο και εκφράσαμε στην τελευταία μου έκθεση σαφώς τι απαιτήσει μας και τις αξιώσεις μας σε ό,τι αφορά τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν ακόμα οι Ρωμά. Χρειάζεται μια νέα προσέγγιση και θα πρέπει να καταπολεμήσουμε τον ρατσισμό αυτό κατά των Αθήγανων. Χρειάζεται ίση συμμετοχή των Ρώμα σε όλα τα επίπεδα της διακυβέρνηση μέσω νομικά δεσμευτικών νομοθετημάτων σε τοπικό και περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και εθνικό επίπεδο. Και όλα αυτά θα πρέπει να ενσωματωθούν στο επόμενο πλαίσιο. Είμαι γιος ε, επιβιώσαντα του ολοκαυτώματος. Έχω χάσει έξι θείους και θείες στο ολοκαύτωμα. Ξέρω πώς είναι, πώς νιώθει κανείς στο πετσί του τον ρατσισμό και δεν θέλω κανένας να νιώσει αυτό που εγώ και ο λαός μου ζούμε καθημερινά. Δυστυχώς το κοινοβούλιο αυτό έζησε Ομιλίε ρατσισμού, Ρατζαμπάσκι, Ουρίκ. Σας παρακαλώ λοιπόν να σκεφτείτε για μία στιγμή πώς θα ήταν να είστε στη θέση μας. Διερωτηθείτε πώς ε, θα αισθανόσαστε αν αντιμετωπίσατε ρατσισμό και απαξιωτικά σχόλια. Δεν έχουμε μόνο τον COVID-19, αγαπητοί συνάδελφοι, έχουμε και μια πανδημία η οποία είναι ίσως και πιο επικίνδυνη, το ρατσισμό. Είμαστε επιτέλους πρόθυμοι, διατεθειμένοι να αντιμετωπίσουμε αυτή την αδικία. Σου Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Φραντς. Τώρα θα δώσω το λόγο στην κυρία Ραφάλσκα από το ECR. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Επίτροπε, για χρόνια θεωρούσαμε ότι οι Ρωμά ήταν κάτι περίεργο. Δεν τους εμπιστευόμασταν, ζούσαν απομονωμένοι στο περιθώριο των κοινωνιών μας στην Ευρώπη. Παρόλο που συμμετείχαν σε μια πολιτιστική κληρονομιά, τη δικιά τους. Ένας Πολωνός ερευνητής δούλεψε πάνω στους Ρωμά και υποστηρίζει ότι αξίζουν πλήρως την αξιοπρέπειά μας και την βοήθειά μας. Εμείς από εκεί που προέρχομαι τους ξέρουμε τους Ρωμά. Έχουν συγκεκριμένες πολιτιστικές αξίες, έχουμε και πολλές γνωστές οικογένειες που είναι Ρωμά. Στη δικιά μου την περιοχή διοργανώνονται και πολλά διεθνή φεστιβάλ. Και με τον κύριο Έντβαντ Μαντίσκι, ο οποίος πρόσφατα γιόρτασε τη δημιουργία της πολιτιστικής τους κληρονομιάς. Έχουμε Ρωμά δηλαδή και πιστεύω πραγματικά ότι η εφαρμογή ε, προγραμμάτων και για άλλους κλάδους κοινωνικής προστασίας πρέπει να βασίζονται στη γνώση. Αυτό είναι ο καλύτερος τρόπος να βοηθήσουμε και τους Ρωμά σήμερα. Το θέμα λοιπόν δεν είναι να προσπαθούμε να βρούμε μία λύση για τα πάντα, αλλά πρέπει να σεβόμαστε τους Ρωμά και να τους επιτρέψουμε να διατηρήσουν τα δικά τους χαρακτηριστικά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Στη συνέχεια, το λόγο έχει τώρα η κυρία Κλέρ Ντέιλι. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Χαίρομαι που μπορώ να μιλήσω για τους Ρωμά αυτή τη βδομάδα που ο, η πρώτη Ρωμά κατάφερε και πέτυχε έδρα στο Ιρλανδικό Κοινοβούλιο. Θυμάμαι όταν έκανε την εκστρατεία της για την άμβλωση, για τα δικαιώματα των γυναικών στην Ιρλανδία. Έχει περάσει πολύ καιρό από τότε. Είναι τόσο πολύ σημαντικό να έχουν δικαιώματα οι άνθρωποι αυτοί που ταξιδεύουν και που είναι θύματα. Στην Ουγγαρία υπάρχουν διακρίσεις σε βάρος των γυναικών Ρωμά. Ε, στην Ουγγαρία και σε άλλες χώρες δεν μπορούν να προβούν στην ιατρική επιστήμη για αν δεν θέλουν να κάνουν παιδιά, για στήρωση. Η στρατηγική που έχουμε είτε για την υγεία είτε για άλλα δεν εφαρμόζονται στην περίπτωση των Ρωμάν. Μπορούμε λοιπόν να έχουμε ό,τι στρατηγικές θέλουμε, αλλά αυτό που χρειάζεται είναι να εφαρμόζονται σωστά, αν πραγματικά θέλουμε να πετύχουμε την ισότητα μεταξύ όλων. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Τώρα θα δώσω το λόγο, τελειώσανε παρεμβάσει εκ μέρου του πολιτικών ομάδων, στην κυρία Σόντροβα. Ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, αναρωτιέμαι γιατί υπάρχει αυτή η κατάσταση όπου οι Ρωμά ζουν σε γκέτο μέσα σε φτώχεια και σε μεγάλη ανεργία. Νομίζω ότι και οι δύο πλευρές πρέπει να συνεισφέρουν στην αλλαγή, και η κοινωνία δηλαδή, αλλά και η η Ρωμά. Θέλω να ευχαριστήσω λοιπόν τον Κυρούλα που εκπροσωπεί τους Ρώμα και που γνωρίζει πάρα πολύ καλά αυτήν την ε, ευθύνη που έχουν εκεί οι ίδιοι οι Ρωμά. Είναι πολύ σημαντικό πραγματικά να σταματήσει αυτός ο φαύλος κύκλος της φτώχειας με εκπαίδευση. Γιατί έχουμε παραδείγματα ανθρώπων Ρωμά οι οποίοι κατάφεραν και μορφώθηκαν γιατί το θέλαν και γιατί κατάφεραν να πετύχουν και στήριξη από τις κοινότητές τους δεν πρέπει να υπάρχει ρατσισμό. Όχι απλώ να τον περιορίσουμε, αλλά να τον απαλείψουμε πλήρω. Πρέπει να ενθαρρύνουμε τι φιλοδοξίε των ανθρώπων αυτών και η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να βοηθήσει και οι χώρε μέλη φυσικά να δραστηριοποιηθούν προ αυτή την κατεύθυνση. Να στηρίξουμε την εκπαίδευσή του. Οι γονεί πρέπει επίση να δραστηριοποιηθούν. Όλα αυτά μπορούν να βοηθήσουν για να σπάσει αυτό ο φαύλο κύκλο αποκλεισμού και αντίθετα να βοηθήσουμε τη συμμετοχή των ανθρώπων αυτών στην κοινωνία. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ. Έχουμε μείνει λίγο πίσω όσον αφορά το χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας, γι' αυτό σας παρακαλώ να τηρείτε το χρόνο σας. Επόμενος ομιλητής είναι ο Μίλιον Μπρέκλετς. Παρακαλώ, ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Όλοι πρέπει να είναι υπεύθυνοι και να φροντίσουν για την συμμετοχή των Ρωμά στην κοινωνία μας. Όλοι, 80% των ανθρώπων αυτών ζουν σε κάποιο είδους απομόνωση. Όλοι πρέπει να βοηθήσουμε, οι κοινωνίες, οι τοπικές αρχές, όλοι. Και χρειάζεται βέβαια και ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο για την ένταξή τους. Το σημερινό πλαίσιο πέτυχε σε ένα βαθμό, αλλά πρέπει να πάμε ακόμα πιο μακριά. Πρώτα απ' όλα πρέπει να κατανοήσουμε όλοι τις διαφορές που υπάρχουν μέσα στην ίδια την κοινότητα των Ρωμά. Ζουν σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές, περιβάλλον. Πρέπει λοιπόν να βελτιώσουμε την κοινωνική και οικονομική κατάσταση των ανθρώπων αυτών. Να εξασφαλίσουμε ότι έχουν πρόσβαση στην υγεία, ότι η κοινωνική και οικονομική τους κατάσταση δεν εξαρτάται από πολιτιστικά κλητήρια και να φροντίσουμε όλες οι χώρες να έχουν την κατάλληλη εθνική στρατηγική. Στην Σλοβανία έχουμε κάτι τέτοιο για παράδειγμα. Είναι ένα καλό παράδειγμα πιστεύω για όλους. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε κύριε Πλές. Φραντς Ζαμέ, παρακαλώ. Ένα λεπτό. Αγαπητοί συνάδελφοι, σήμερα ζητάμε περισσότερα χρήματα για μια στρατηγική ένταξη των Ρωμά. Μα δεν θα αλλάξετε μια κατάσταση που εξαρτάται από πολλούς λόγους και κυρίως πολιτιστικούς, προσφέροντας περισσότερα χρήματα. Ούτε είναι δικός μας ρόλος να στηρίξουμε οικονομικά ή να αναλάβουμε την ευθύνη για μια επιλογή ζωής που έχουν κάνει οι ίδιοι. Στη Γαλλία έχουμε πάρα πολλού άνεργους και πάρα πολλού στοχούς ανθρώπους. Η οικονομική τους κατάσταση, το επενθυμίσαμε και πριν, επιδεινώθηκε με την κρίση του κορονοϊού. Πώς λοιπόν να εξηγήσουμε στους συμπατριώτε μας ότι επειδή θέλουμε να είμαστε ανθρωπιστές, για κάποιους ε, ανθρώπους αποφασίζουμε να δώσουμε περισσότερα χρήματα, περισσότερο χρόνο, περισσότερα μέσα ώστε να ενταχθούν ενώ δεν το θέλουν. Μέσα στις δυσκολίες και την κρίση που αντιμετωπίζουμε πρέπει να επιλέξουμε να στηρίξουμε τη Γαλλία και τους Γάλλους πρώτα εμείς. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πρόεδρος. Παρακαλώ. Αυτό που κάνει το ID τώρα είναι αυτό που δεν θέλουμε να δούμε. Κάνει διάκριση κατά ανθρώπων. Τους κάνετε να φαίνονται λες και είναι εγκληματίες. Εγώ πιστεύω θα πρέπει να διαγραφούν όλα όσα είπε το ID μέχρι τώρα. So observation... Αυτή η παρατήρηση έχει την αξία της, αλλά θα πρέπει να θυμόμαστε ότι οι ευρωβουλευτές πρέπει να σέβονται αλλήλους και όντως κυρία Ζαμέ είπατε πράγματα τα οποία ίσως να είναι προσβλητικά για τους άλλους. Παρακαλώ να κρατάτε την αξιοπρέπεια Η πρόεδρο συνεχίζει. Θα προχωρήσουμε και θα δώσω το λόγο στον κύριο Τζαμπάσκι. Όταν ακούμε αυτά τα πράγματα να απευθύνονται στους συναδέλφους. Παρακαλώ, σας κάνω έκκληση να τιμωρηθούν, να υπάρξουν κυρώσεις. Τώρα, εσείς συνάδελφοι μας λέτε ότι υπάρχουν διακρίσεις σε αυτή τη χώρα. Εγώ δεν μπορώ να το συζητήσω αυτό, ε, ε, ίσως με ακρίβεια, γιατί ίσως να μην ξέρετε πού πέφτει καν η Βουλγαρία. Αλλά θα ήθελα να σας καλέσω ωστόσο να έρθετε όλοι στη Βουλγαρία και να δείτε πώς ζει ο κόσμος σε μικρούς καταβλισμούς πώς οι ηλικιωμένοι ε, δέχονται την βία από αυτήν την εθνοτική ομάδα. Ελάτε να δείτε με τα ίδια σας τα μάτια για να ξέρετε για τι πράγμα μιλάμε. Συνάδελφοι, τώρα ναι, κουνάτε το κεφάλι σας σε μένα, αλλά εσείς ε, είστε, ε, εσείς μπορείτε να με κατηγορήσετε για κάτι, αν ναι, τότε πρέπει να πάμε στο δικαστήριο. Μάλιστα, εάν δεν το κάνετε αυτό στο δικαστήριο, τότε μάλλον θα πρέπει να ντρέπεστε για τη συμπεριφορά σας. Excuse me, I have to call for... Πρόεδρος, κοιτάξτε, ε, ε ηρεμήστε. Αυτό δεν είναι συζήτηση. Ο καθένας έχει ε, χρόνο ομιλίας. Excuse me, uh, if you have if you have a complaint on the basis of rules. Πρόεδρος, αν έχετε ε, παράπονο όσον αφορά τον κανονισμό λειτουργίας, μπορείτε να διαμαρτυρηθείτε στον Πρόεδρο. Εμείς θα συνεχίσουμε. Συνομιλία εκτός μικροφώνου. Sorry, excuse me. Excuse me, Mr. Κύριε Τζαμπάσκι, παρακαλώ. Δεν μπορείτε να κάνετε, μπορείτε να κάνετε προσωπική δήλωση στο τέλος της συζήτησης, αλλά πρέπει να προχωρήσουμε. Δείξτε σεβασμό στον πρόεδρο της Ολομέλειας. Διαβάζω τον κανονισμό. Πώς έχει ο κανονισμός. Όχι, ακούστε με. Μπορείτε να κάνετε προσωπική δήλωση στο τέλος της συζήτησης, αλλά όχι τώρα. Τώρα συνεχίζεται η συζήτηση και τώρα θα δώσω το λόγο στον κύριο Λοράντ Βίντσεκ για ένα λεπτό. Παρακαλώ κύριε Βίντσεκ. Ευχαριστώ πρόεδρε αγαπητοί συνάδελφοι. Οι πολίτες Ρωμά αναφέρονται συλλογικά μετά από δέκα χρόνια στρατηγικών για τους Ρωμά να θυμάστε ότι κάθε ένα στα τρία παιδιά ζει σε ένα σπίτι και, ε, και πεινά κάθε ε, τουλάχιστον δύο φορές το μήνα. Δεν μπορούμε να το αρνηθούμε αυτό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να παρέχει την ενθάρρυνση και το συντονισμό προς τα κράτη-μέρη για να απομακρυνθούν από την θεσμική και πολιτική αδράνεια. Στην κεντρική Ανατολική Ευρώπη πρέπει να δοθεί μεγάλη προτεραιότητα ώστε να αντιμετωπιστεί η πείνα, η φτώχεια και οι στερήσεις στι κοινότητε των Ρωμά. Έπειτα, στρατηγικέ εκπαίδευση για του Ρωμά, επαγγελματική κατάρτιση και άλλου είδου κατάρτιση επίση. Καλύτερη πρόσβαση είναι το τρίτο στην αγορά εργασία. Στι κοινωνίε μας πρέπει να κάνουμε περισσότερα για να καταπολεμήσουμε τι διακρίσει, να ενημερώσουμε το κοινό για την ευάλωτη κατάσταση των Ρωμά. Όλα αυτά είναι εκπαίδευση. Σας ευχαριστώ. Θα σε ευχαριστώ κύριε Βίνση. Και τώρα θα δώσω το λόγο στην Επίτροπο Έλενα Ντάλι και πάλι. Αξιότιμοι Ευρωβουλευτές, σας ευχαριστώ πολύ που μου είπατε τις απόψεις σας. Σας ευχαριστώ πολύ για την αφοσίωσή σας και για την στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο θέμα που συζητάμε σήμερα. Το νέο πλαίσιο θα προωθήσει την αποτελεσματική ισότητα, την συμμετοχή επίσης των Ρωμά, χωρίς αποκλεισμούς. Θα φροντίσει να μην υπάρχουν τάσεις κατά των ανθρώπων αυτών, θα φροντίσει για την μείωση της φτώχειας και του αποκλεισμού και θα φροντίσει επίσης και για την συμμετοχή των Ρωμά, δίνοντας τους περισσότερες δυνατότητες και εμπιστοσύνη. Είναι πολύ βασικό για να υπάρχει αποτελεσματική πρόσβαση των Ρώμα σε εκπαίδευση που να είναι ποιότητας και χωρίς αποκλεισμούς όπως επίσης σε απασχόληση ποιότητας, σε υγεία ποιότητας και επίσης σε δυνατότητες στέγασης χωρίς διακρίσεις. Ήρθε η στιγμή να κλείσει αυτό το χάσμα κοινωνικό και οικονομικό ανάμεσα στους Ρωμά και τους άλλους. Και από αυτό το πνεύμα χαίρομαι που η Γερμανική Προεδρία βάζει την ισότητα των Ρωμά, την συμμετοχή τους στην ημερήσια διάταξη. Και θέλω να ευχαριστήσω και πάλι την καγκελάριο Μέρκελ, η οποία επανέλαβε τη δέσμευσή της υπέρ της ισότητας με σαφήνια στα πλαίσια της Γερμανικής Προεδρίας και το επανέλαβε χτες εδώ. Βασίζομαι βέβαια και στην στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και στο έργο βέβαια που βρίσκεται μπροστά μας προκειμένου να επιτελεστεί. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Πίτρο Πεντάλη. Το λόγο έχει τώρα ο υπουργό. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Επιτροπέ, αξιότιμοι βουλευτέ Σας ευχαριστώ που συμμετείχα σήμερα στη συζήτηση αυτή και φαίνεται ότι σε μεγάλο βαθμό είμαστε σύμφωνοι και γνωρίζουμε επίσης πόσο δύσκολο είναι το έργο που έχουμε μπροστά μας αλλά από κοινού θα το αναλάβουμε με μεγάλη δέσμευση και μέχρι τέλος του χρόνου θέλουμε να έχουμε μια στρατηγική η οποία θα έχει ως αποτέλεσμα την ενίσχυση όλων μας. Θέλουμε να συμβάλλουμε συγκεκριμένα, θέλουμε μια διάσκεψη να οργανώσουμε και φοβάμαι ότι θα είναι εικονική η διάσκεψη αυτή. Παρ' όλα αυτά θεωρώ ότι θα αποτελέσει μια περαιτέρω ευκαιρία για την ανταλλαγή όχι μόνο εδώ στο Κοινοβούλιο και στα άλλα θεσμικά όργανα, αλλά και με τους άμεσα ενδιαφερόμενους κάτι μου προκαλεί έκπληξη, το οποίο το άκουσα όχι μόνο εδώ, αγαπητοί βουλευτές, σε ό,τι αφορά τους ε, Ρωμά και το πώς θα αντιμετωπίσουμε. Δεν μιλάμε για φιλοξενία. Μιλάμε για πολίτες των ε, πολιτών, των, των χωρών μας. Είναι πολίτες των χωρών μας και έχουν τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες υποχρεώσεις που έχουμε όλοι μας. Δεν είναι φιλοξενούμενοι Και τμήμα λοιπόν της διακριτικής μεταχείρισης είναι το ότι τις αποκλείουμε από μια κοινωνία ελεύθερης και ίσης συμμετοχής. Και επίσης κυρίες και κύριοι δεν μιλάμε για προνόμια. Μιλάμε για κάτι εντελώς απλό. Μιλάμε για τα ίδια δικαιώματα, για την ίση αντιμετώπιση των 6-7 εκατομμυρίων πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωση και θα πρέπει να είναι σαφές ότι μια επίθεση κατά τον Ρωμά αποτελεί πάντα και μια επίθεση κατά των ευρωπαϊκών αρχών, κατά των ίδιων μας των αρχών. και είμαι ευγνώμων για τους βουλευτές εκείνους που επεσήμεναν ότι χρειάζομαστε κυρίως τόλμη και παραδείγματα η Ρωμά δεν είναι μόνο προβληματικός παράγοντας. Αντιθέτως, η Ρωμά ως τμήμα της ε, κοινωνίας μας μας εμπλουτίζουν. Για παράδειγμα, στο Βερολίνο με το ε, Ινστιτούτο το Ίδρυμα Ρωμά για τον πολιτισμό θέλαμε να δείξουμε ακριβώς αυτό, ότι είναι σημαντική και πολύ συγκεκριμένη η συμβολή των Ρωμά στην πολιτιστική ταυτότητα της Υπήρου μας και θα ήθελα στο πλαίσιο της στρατηγικής να καταφέρναμε να ξεκαθαρίσουμε ότι μιλάμε για ένα παράγοντα εμπλουτισμού, για πολλέ ευκαιρίε ε, τις οποίες πρέπει να συνδέσουμε με τον παράγοντα Ρωμά. Και ασφαλώς αγαπητοί συνάδελφοι και δεν πρόκειται μόνο για τα χρήματα. Μιλάμε όχι μόνο για οικονομικά μέσα. Μιλάμε για μία στάση. Πώς θα αντιμετωπίσουμε τη μεγαλύτερη αυτή εθνοτική μειονότητα της Ευρώπης. Και θα ήθελα και στα πλαίσια της συζήτησης κατά του ρατσισμού που γίνεται σε παγκόσμιο επίπεδο. Η... Το Black Lives Matter να γίνει Roma Lives Matters. Ότι μετράνε δηλαδή η ζωή όλων των Ρώμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Υπουργέ Ρότ. Ο κύριος Ζαμπόφσκι τώρα, ο οποίος βάσει του άρθρου του κανονισμού 103 θέλει να παρέμβει για να διαμαρτυρηθεί, να διατηρηθεί για τα σχόλια που έγιναν προηγουμένως. Να ξέρετε όμως ότι δεν θα κάνουμε συζήτηση. Έχετε το λόγο για τρία λεπτά, έτσι όπως προβλέπει ο κανονισμός. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρε, και κύριε Επιτροπέ, όταν ακολουθήσει κανείς ένα είδος ζωής, ένα χρώμα και πει ότι μόνο ένα χρώμα μετράει στη ζωή, αυτό δεν είναι διάκριση. Είναι διάκριση αν λες ότι η μαύρη ζωή αξίζει, όχι υπόλοιπε. Λοιπόν, κυρία Πρόεδρε, θέλω να εξηγήσω και να πω το εξής. Άκουσα από δύο συναδέρφους να λένε ότι είμαι ρατσιστής αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό και αποδεικνύεται στα δικαστήρια. Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα λοιπόν ένα βίντεο με αυτά που είπαν οι συνάδελφοι, αυτοί που αναφέρθηκαν σε μένα και σε αυτούς που βρίσκονται πίσω από μένα και που είπαν ότι είμαστε ρατσιστές και να αποδείξουν στο δικαστήριο ότι έχουν δίκιο. Αυτό πρέπει να γίνει. Επίσης, πρέπει να υπάρξουν κυρώσει σε βάρος των συναδέλφων αυτών, γιατί αυτοί οι συνάδελφοι στην αριστερά ουσιαστικά κάνουν υποθέσεις και μιλάνε για την ελευθερία της έκφρασης και νομίζουν ότι επειδή υποστηρίζουν ελευθερία της έκφρασης μπορούν να πούν ό,τι θέλουν. Όχι λοιπόν. Πρέπει οι απόψεις όλων μας να είναι ισότιμες. Αδικό έχω. Πρέπει να έχουν το ίδιο βάρος. Όλοι. Και αν κάποιος από πίσω πει ότι είμαι ρατσιστής πρέπει να το αποδείξει με όνομα και επίθετο και να αποδείξει ότι όντω ισχύει αυτό που λένε. Λοιπόν, οι αριστεροί, οι μπολσεβίκοι, οι κομμουνιστές, όσοι αγαπούν τον κομμουνισμό, αυτή την κατάχρηση κάνουν. Όχι, πρέπει να λογοδοτήσουν για τις πράξεις τους. Λοιπόν, δεν σέβονται. Εγώ μπορώ να εξηγήσω τι υποστηρίζω. Κάποιοι αναφέρθηκαν στη Βουλγαρία. Και εγώ μπορώ να σας πω ότι δεν ξέρω που βρίσκεται, δεν ε, έχω πάει ποτέ. Μπορώ να σας πω όμως ότι δεκάδες ε, Βούλγαροι, Ρώμα, θα γελάνε μαζί σας και δεν θέλουν να τους εκπροσωπείτε. Δεν τους εκπροσωπείτε εξάλλου, γιατί αποτελούν μέρος της βουλγαρικής κοινωνίας. Είναι εξαίρετοι πολίτες δεν πρέπει να με διακόπτετε. Μη με διακόπτετε. Δεν είναι πολιτισμένο κάτι τέτοιο. Ούτε δείχνετε σεβασμό έτσι όταν με διακόπτετε. Κάθε άποψη μετράει και έχει το ίδιο βάρος. Πιστεύω επίσης ότι οι άνθρωποι πρέπει να έχουν το δικαίωμα να μιλάνε. Αφήστε με να ολοκληρώσω την πρότασή μου. Πρόεδρε, πρέπει να επιβάλλετε κυρώσει στους συναδέλφους. Με διακόπτουν. Να ξέρετε ότι ζητάω το βίντεο να πάω στη δικαιοσύνη και να αποδείξουν οι συνάδελφοι αυτοί αυτά που λένε και ισχυρίζονται για μένα. Πρόεδρος, ωραία. Ο κύριος Τζαμπάφσκι χρησιμοποιήσει το δικαίωμά του να κάνει επιπροσωπικού δήλωση όσον αφορά τις παρατηρήσεις που ακούστηκαν πριν. Και εννοείται ότι θα ζητήσουμε το transcript της συζήτησης αυτής για να εκτιμήσουμε αν πρέπει να υπάρξει κάποια συνέχεια από το Προεδρείο. Ευχαριστώ. Συνεχίζουμε λοιπόν τώρα και περνάμε στο επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη παρακαλώ. Και πρόκειται για την συζήτηση όσον αφορά κανονισμό του Συμβουλίου για την προστασία του προπολογισμού τη Ένωση στην περίπτωση γενικευμένων ελλείψεων όσον αφορά το κράτο δικαίου στα κράτη-μέλη. Και θα δώσω πρώτα το λόγο στο Συμβούλιο. Παρακαλώ, κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο. Ε, Σα ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Πρόεδρε, αξιότιμοι κύριοι βουλευτέ. Θα ήθελα ευθύ εξ αρχή ε, να πω το εξή και να διευκρινίσω το εξή. Κάτι που ακούγεται ενδεχομένω αυτονόητο σε όλου μα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι σε πρώτο επίπεδο μία νομισματική ένωση, μια νέα αγορά. Είμαστε κυρίως μια νομική ένωση, μια ένωση αξιών. Αυτές οι αρχές οι οποίες επηγάζουν από τις συνθήκες μας και οι οποίες κατοχυρώνονται από τις συνθήκες μας είναι αρχές που μας ε, διέπουν όλους μας. Σας ευχαριστώ λοιπόν αγαπητοί βουλευτές που μου δίνετε την ευκαιρία να σας ενημερώσω τι γίνεται με τις διαπραγματεύσεις στο Συμβούλιο σε ό,τι αφορά τον κανονισμό και την προστασία του προπολογισμού τη Ένωση σε περίπτωση γενικευμένων ελλείψεων σε ό,τι αφορά το κρατό δικαίου στα κράτη-μέλη. Η πρόταση αυτή αποτέλεσε ένα απόσπαστο σημείο του πολιτικού συμφώνου, του πολιτικού πακέτου μάλλον, το οποίο πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 2 Μαΐου του 2018 και το Συμβούλιο Αντιμετωπίζεται λοιπόν το θέμα αυτό, την πρόταση αυτή, στα πλαίσια του πολιτισμικού πλαισίου. Τον Νοέμβριο λοιπόν του 2018 εκφράστηκε η επιφύλαξη μελέτη και πλέον έχει περάσει πολλές χρόνος και διαπιστώνουμε ότι δύο είναι τα στοιχεία τα οποία για τις αντιπροσωπείες του Συμβουλίου είναι ιδιαίτερα αμφιλεγόμενα. Καταρχάς η σύνδεση με το κράτος δικαίου και κατά δεύτερο ο τρόπος ψηφοφορίας για την έγκριση των μέτρων. Η Προεδρία θεωρεί ότι χωρίς πολιτικές κατευθυντηρίες γραμμές ε, των αρχηγών ε, κρατών και κυβερνήσεων δεν θα μπορούσε να έχει επιτευχθεί πρόοδος στα θέματα αυτά και ως εκ τούτου τα θέματα αυτά συμπεριλήφθησαν σαν διαπραγματευτικό κοιτίο τα οποία η Αυστριακή Προεδρία τα πρότεινε. Η Ρουμανική Προεδρία συνέχισε τις εξειδικευμένες διαπραγματεύσεις για τα άλλα στοιχεία της πρότασης και υπέβαλε συνολικά πέντε συμβαστικές προτάσεις από πλευράς της Προεδρίας οι οποίες βασίζονταν και σε πολιτικά ζητήματα αλλά και σε τεχνικά ζητήματα. Μια λεπτομερής λοιπόν επισκόπηση για την διαδικασία αυτή και τα βασικά στοιχεία της διαπραγμάτευσης ε, περιλαμβάνονται στην ε, έκθεση πρόοδου της Ρουμανικής Προεδρίας. Ο πρόεδρος ε, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ανέλαβε το καθήκον να σχηματίσει μια σαφή εικόνα για το πώς οι αρχηγοί αρχών και κρατών και κυβερνήσεων ε, τοποθετούνται εναντί του συνολικού πακέτου για το πολιτιστικο δημοσιονομικό πλαίσιο στα πλαίσια της πρότασης ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το Φεβρουάριο λοιπόν του 2020 υποβλήθη μια πρόταση από πλευρά του Συμβουλίου και ξέρετε ότι αυτέ οι εργασίε ακόμα δεν έχουν ολοκληρωθεί. Χωρί κατευθυντήριες γραμμέ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τα πολιτικά στοιχεία, και τον έλεγχο του πακέτου δεν υπάρχει ουσιαστικά δυνατότητα για συνέχιση των εργασιών στο τεχνικό επίπεδο. Μόλις λοιπόν να διαμορφωθούν ε, οι πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές αυτές και ελπίζουμε αυτό να το πετύχουμε σύντομα, η Προεδρία άμεσα πάρα αυτά θα, θα συμπεριλάβει το κείμενο αυτό για να ξεκινήσουν το συντομότερο δυνατόν διαπραγματεύσει με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ο πρόεδρος Μισελ λοιπόν μας ενημέρωσε για τις προετοιμασίες για την επερχόμενη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Οι προτάσεις λοιπόν είναι τμήματα του συνολικού πολιτικού οικονομικού πλαισίου. Θα πρέπει να φροντίσουμε λοιπόν στα πλαίσια της κανονικής ε, διαδικασίας διαπραγματεύσεων να μην υπάρξει οποιαδήποτε καθυστέρηση και να εξασφαλιστεί η έγκριση από πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σα ζητώ συγγνώμη αν είμαι πολύ περίπλοκο, αλλά είναι το θέμα πολύ τεχνικό, πολύ περιπλοκό. Και ήθελα να σα ενημερώσω λοιπόν για το πώ έχουν τα πράγματα στου κόλπου του Συμβουλίου. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον πρόεδρο Ροτ. Και τώρα να δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο κ. Χάνα έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητοί βουλευτέ, η σύνοδο του επόμενη εβδομάδα θα σημειώσει ένα ορόσημο και ξέρουμε όλοι μας το έχουμε ζήσει και στις χώρες μας και στις εκλογικέ μας περιφέρειες. Ο κορονοϊός έχει αλλάξει τον τρόπο ζωής μας και την οικονομία μας. Αυτή η πρόκληση ανεφρεγουμένου είναι η στιγμή όπου η Ευρώπη θα μετρήσει πιο πολύ παραποτέ. Οι ζωές και το μέλλον των ανθρώπων και των επιχειρήσεων και οι προοπτικέ πολλών περιφερειών εξαρτώνται από το πρόγραμμα ανάκαμψής μα. Γι' αυτό λοιπόν είναι ακόμα πιο σημαντικό κάθε ευρώ που θα δαπανηθεί με τον ε, κοινό ευρωπαϊκό προπολογισμό να έχει προστιθέμενη αξία, να αποτελέσει μια πραγματική επένδυση στο μέλλον. Οι Ευρωπαίοι αναμένουν λοιπόν από εμά να προστατεύσουμε τα λεφτά των φορολογουμένων και καλά κάνουν. Όπω και να έχει όμω ε, το πακέτο αυτό έχει τη σημασία του. Γι' αυτό λοιπόν εκτιμώ αυτή τη συζήτηση πριν από τη Συνοδόν. Θα ήθελα να τονίσω τρία σημεία. Καταρχά, όπου τίθεται θέμα ε, γενικευμένων ελλείψεων σε ό,τι αφορά το κράτο δικαίου στα κράτη-μέλη, χρειάζεται ένα αποτελεσματικό εργαλείο για να προστατεύσουμε τα χρήματα των φορολογουμένων. Και έτσι λοιπόν το κράτο δικαίου αποτελεί ένα αυθεντικό μηχανισμό προστασία του προπολογισμού. Κατά δεύτερον, θα πρέπει να προστατεύσουμε τον προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση σύμφωνα με τι ε, συνθήκε, σύμφωνα με το άρθρο 7 των συνθήκων. Τρίτον, πρόκειται για ένα στόχο, ένα αντικειμενικό μάλλον ε, και διαφανή μηχανισμό για να προστατεύσουμε σωστά και καλά μέτρα για την χάραξη του προπολογισμού. Το βάρος της ευθύνης θα το φέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο. Τα μέτρα θα πρέπει να βασίζονται σε συγκεκριμένα περιστατικά και γεγονότα και αριθμητικά στοιχεία. Θα ήθελα να ευχαριστήσω λοιπόν το Κοινοβούλιο Αρχνέου για την υποστήριξή του για την πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την νομοθετικό ψήφισμα τη 4η Απριλίου του 2019. Τα θέματα που έθεσε το Κοινοβούλιο σημειώθηκαν όντω Η ανάγκη λοιπόν να εξασφαλίσουμε την προστασία των τελετικών δικαιούχων είναι σημαντικό να μην πληρώσουν τελικά τα σπασμένα για τις ελλείψεις σε ό,τι αφορά το κράτος δικαίου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα θέσει το θέμα αυτό στους τριμερείς διαλόγους, γιατί στόχος μας είναι σαφής. Θέλουμε ένα μηχανισμό, γενικό μηχανισμό για την προστασία του ευρωπαϊκού προπολογισμού και να εξασφαλίσουμε τα χρηστά δημοσιονομικά μέτρα. Το Νοέμβριο του 2019 η Επιτροπή του Κοινοβουλίου αποφάσισε να ξεκινήσει τις διαθεσμικές διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο και ελπίζω να ξεκινήσει γρήγορα ο διάλογο υπό την αιγύδα τη γερμανική Προεδρίας. Σημειώσαμε και χαρήκαμε με τι δηλώσει του Συμβουλίου άλλωστε. Υπολογίζω στην συνεχιζόμενη υποστήριξη από πλευρά του Κοινοβουλίου για να εξευρεθεί μια λύση η οποία θα προστατεύσει την αποτελεσματικότητα και τη φιλοδοξία του σημαντικού αυτού μηχανισμού για την προστασία του προπολογισμού. Είναι κοινό μα στόχο. Και το κράτο δικαίου είναι βασικό στοιχείο σε ό,τι αφορά την διαπραγμάτευση του πολιτισμού δημοσιονομικού πλαισίου. Ο χρόνο πιέζει, αγαπητοί βουλευτέ. Μόνο αν όλοι μα ε, καταφέρουμε να πετύχουμε συμφωνία μέσα στο καλοκαίρι, έχουμε μια ευκαιρία να πετύχουμε αυτά που θέλουμε. Ξέρω ότι είναι πολύ φιλοδόξο όλα αυτά και θα ήταν μια ταχύτητα άνευ προηγουμένου. Μα και οι εποχές που ζούμε είναι ανευπροηγουμένου και νομίζω ότι οι πολίτες και οι επιχειρήσεις ε, θεωρούν ότι κάθε μέρα μετράει. Γι' αυτό λοιπόν δρούμε προς το κοινό μας συμφέρον. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Χάν. Κύριε Επίτροπε, θα δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Σάρβαμα. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, ήδη πριν από πάνω από ένα χρόνο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, εξέφρασε τις απόψεις του για την ρύθμιση όταν υπάρχει ανεπάρκεια όσον αφορά την εφαρμογή του κράτους δικαίου. Ο μηχανισμός αυτός ο κράτους δικαίου θα βοηθήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση να στηρίξει τις αξίες μας και να προστατεύσει τα χρήματα των Ευρωπαίων φορολογούμενων και τον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό από καταχρήσεις. Και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει στέρες απόψεις. Χρειαζόμαστε πράγματι ένα μηχανισμό ισχυρό για το κράτος δικαίου. Και είναι κάπως ανησυχητικό που οι πληροφορίες που έχουμε από το Συμβούλιο μέχρι τώρα δείχνουν ότι εξακολουθούν να υπάρχουν διαφωνίες στους κύκλους του Συμβουλίου, ακόμα και για βασικά στοιχεία του κανονισμού αυτού. Ζητήσαμε από το Συμβούλιο να κάνει ουσιαστικές συζητήσεις και διαπραγματεύσεις και να συμμετέχουμε να μην είμαστε απλώς για να βάλουμε τη σφραγίδα μας σε μια απόφαση που έχει ήδη ληφθεί, αλλά να συμμετέχουμε και εμείς στις διαπραγματεύσεις. Οπότε παραμένει το ερώτημα προς το Συμβούλιο. Ποιο είναι το επίπεδο φιλοδοξιών σας. Είναι αντίστοιχο των δικών μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Σάρβαμα. Τώρα εκ μέρου των σοσιαλδημοκρατών το λόγο έχει η κυρία Καρδιαθαμπάλ Ρούμπιαλ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε Χάν, κύριε Υπουργέ Ροτ, χαίρομαι και χτες χάρηκα που άκουσα ότι η Προεδρία μεταξύ των προτεραιοτήτων της έχει τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και συμφωνούμε ότι έχει πολύ μεγάλη ε, σημασία η τήρηση του κράτους δικαίου. Είναι βασικό στοιχείο του ευρωπαϊκού οικοδομήματος και βασικό ευρωπαϊκό κεκτημένο. Είμαστε μια ένωση δικαίου και αξιών. Και αν σήμερα κάνουμε αυτή τη συζήτηση, είναι ακριβώ επειδή θέλουμε να υπογραμμίσουμε ότι για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αυτό δεν αποτελεί απλώ μια προτεραιότητα, πρόκειται για μια προπόθεση αναγκαία για να προχωρήσουν οι διαπραγματεύσει επί του προπολογισμού που θα έχουμε του επόμενου μήνε. Και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει εκφράσει με σαφήνεια τη θέση του απέναντι στην πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Χρειάζεται τήρηση ανθρωπίνου δικαίου, αλλά επίση να προσέχουμε ότι θα τηρούνται όλε οι πτυχέ που έχουν να κάνουν με το κράτο δικαίου και που συνυπογράφουν ουσιαστικά όλε οι χώρε μέλη όταν εντάσσονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή να αντιμετωπίζονται οι φορολογικέ απάτε, δημοσιονομικέ απάτε και χτε ήδη εδώ είπε ότι πρέπει να υπάρχει συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να προστατεύσουμε την κοινή μας Ευρώπη. Μαζί θα ενισχύσουμε την Ευρώπη. Και εσείς το υπογραμμίσατε. Οπότε είμαστε έτοιμοι για διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο. Διαπραγματεύσεις, το τονίζω αυτό, γιατί διαπραγματεύσεις πρέπει να γίνουν. Εμείς δεν είμαστε εδώ απλώς για να βάλουμε πλάτη σε μια συμφωνία στην οποία θα καταλήξει το Συμβούλιο. Όχι, διαπραγματεύσεις μαζί μας, ώστε μαζί να χτίσουμε αυτή την κοινή Ευρώπη που θα είναι πρότυπο στον κόσμο όσον αφορά την τήρηξη των αξιών και του κράτους δικαίου. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, κύριε κυρία Θαμπάλου Ρουμπιάλ. Τώρα, θα δώσω το λόγο στον κύριο Κέρνερ. μισή λεπτό παρακαλώ. Κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, η Καγελάριος χθε στην ομιλία της ε, απέθυνε μια έντονη έκκληση για τα θεμελιώδη δικαιώματα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξεκίνησε μάλιστα την ομιλία τη έτσι και ήταν καλό αυτό και απαραίτητο. Αλλά αυτό σημαίνει ότι θέλουμε συνέπεια από πλευρά τη ε, ε, Καγκελαρίου για τον μηχανισμό για τα θεμελιώδη δικαιώματα. Γιατί όντω η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κάτι παραπάνω από μια νέα αγορά. Είναι μια κοινότητα αξιών. Και με τι διαπραγματεύσει στο Συμβούλιο, όπου έχουμε σημειώσει τέλμα στο σημείο αυτό. Καταδικάζεται αυτή η κοινότητα αξιών. Μας παρουσίασε ο Υπουργός πολύ καλά τι γίνεται στο Συμβούλιο. Διαπιστώνουμε ότι τα κράτη-μέλη ουσιαστικά σε ό,τι αφορά τον μηχανισμό του κράτους δικαίου δεν συμφωνούν για δύο σημεία. Για το μηχανισμό και για το κράτος δικαίου. Αυτή είναι η κατάσταση στο Συμβούλιο. Χρειάζεται μια συνέπεια. Δεν μπορούν να δεχόμαστε. Δεν μπορεί να δεχόμαστε τα κόντυλα τη Ευρωπαϊκή Ένωση και να καταπατάμε τι αξίε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θέλουμε να τιμωρήσουμε κανέναν. Θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα δαπανούνται ευρωπαϊκοί πόροι σε... να καταλήγουν στις τσέπε σκοτεινών δυνάμεων που καταπολεμούν τελικά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό θα πρέπει να εξασφαλίσουμε και εκεί ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέλουμε να θέσουμε ένα σαφές μήνυμα προς το Συμβούλιο. Είναι τεράστια ευθύνη να βγάλει κόκκινη κάρτα σε αυτούς που αγνοούν το κράτος δικαίου στην Ευρώπη. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Κέρνερ και τώρα από την ομάδα των ID να πάρει το λόγο ο Νίκολας Μπέι. Αναφέροντα τι απειλέ για το κράτο δικαίου, θα πρέπει να αναφερθούμε στη συζήτηση στη Μάλτα ή στη Σλοβακία, όπου δημοσιογράφοι έχουν δολοφονηθεί μέσα σε πλαίσιο πολιτικό, ε, διεφθαρμένο, σοσιαλιστικό. Ακόμα και σήμερα όμω, αυτοί που στοχεύουμε και θέλουμε να του στερήσουμε από τα ευρωπαϊκά κονδύλια είναι πάλι και ξανά η Πολωνία και η Ουγγαρία. Είναι δημοφιλείς κυβερνήσεις που χαίρουν ε, ε, μεγάλης ε, δημοκρατικής θεμητότητας και που έχουν καλύτερα εκλεγεί από ό,τι εσείς όλοι εδώ. Πολύ καλύτερα έχουν εκλεγεί από όλους όσους θέλουν να τους κάνουν ε, μαθήματα. Εσείς χρησιμοποιείτε το τον εκβιασμό, τον μεταναστευτικό, αλλά και το γεγονό ότι δεν θέλουν να δεχτούν τις ομάδες LGBTQI και διάφορου άλλου ακραίου. Και μιλάμε για δίκαιο, αλλά κανεί δεν μιλά για τον διορισμό του κ. Ντυπό Μορετή ω Υπουργό Δικαιοσύνη του κ. Μακρόν πριν από λίγε μέρε. Αυτό ο ίδιο κύριος είχε ζητήσει την απαγόρευση του κυρίου κόμματο αντιπολίτευσης στη Γαλλία. Ε, άρα λοιπόν το δίκαιο χρησιμοποιείται πολιτικά να επιβληθούν άνθρωποι κατά ενάντια στη βούληση των λαών. Όμως όσο θέλουμε να τους υποτάξουμε τους λαούς τόσο περισσότερο αντιδρούν και θα αντιδράσουν. Ευχαριστώ κύριε Μπέι. Και τώρα αξιονόματος των Πρασίνων ο κύριος Φρόιντ, δύο λεπτά. Αγαπητέ Μιχαλ Ρότ, την προηγούμενη εβδομάδα ήμουν στην Ποταπέστη και συναντήθηκα με ε, τους αντιπολιτευτές του Βίκτορ Όρμπαν που βοηθάνε τους ε, πιο αδύναμους, τους άστεγους. Ο Ιβάνε λοιπόν ε, προασπίζεται τους αδύναμους. Και τον καταστρέφει λοιπόν ο Ορμπάν. Του κατάργησε τους δημόσιους πόρους τους, προσπαθεί να καταστρέψει και το έργο μιας ολόκληρης ζωής σαν μαφιόζος. Και ο Ιβάνη δεν είναι και ο μόνος. Οποιοςδήποτε ασκεί κριτική αντιμετωπίζει τα ίδια. Τους α, απειλούν να τους καταστρέψουν, να τους απολύσουν. Δεν έχει πλέον χώρο η αντιπολίτευση στο καθεστώς του Ορμπάν. Την προηγούμενη χρονιά δεν υπήρξε ούτε ένα τόξο, ούτε μία συνέντευξη με εκπροσώπους της αντιπολίτευσης. Και στο μεταξύ βγάζουν όλο και πιο πολλά οι κοντινοί του Ορμπάν. Ο πατέρας του, ο κουνιάδος του. Πρόκειται λοιπόν για μια οικογένεια εκατομμυριούχων σήμερα. Την προηγούμενη εβδομάδα λοιπόν ήμουνα ο μόνος που ταξίδεψε προς την Ουγγαρία. Είναι πραγματικά παραλογισμός. Ο, λό, ρόλος λοιπόν της Γερμανίας είναι επονίδιστος. Η κυβέρνηση για παράδειγμα έχει μειο νοτικό μόνο συμμετοχή στην ε, γερμανική εταιρεία τηλεπικοινωνιών στην Ουγγαρία. Αυτέ οι διαπραγματεύσει λοιπόν για το πολιτικό δημοσιονομικό πλαίσιο είναι η τελευταία ευκαιρία για να καταδείξουμε ότι αυτοί οι κανόνε, αυτέ οι αξίε δεν είναι διαπραγματεύσιμε για μα, είναι αναπαλωτρίωτε, ότι δεν μπορούμε να πατάμε δισεκατομμύρια χωρί έλεγχο, χωρί κυρώσει. Σα παρακαλώ λοιπόν αυτά μην τα θυσιάσετε την επόμενη εβδομάδα. Kiitos Σας ευχαριστώ. Τώρα, εξ ονόματος του ECR, θα δώσω το λόγο στην κυρία Βυσνιεύσκα. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, είναι αλήθεια ότι οι συνθήκε είναι η πηγή τη νομοθεσία. Στηρίζουμε τέτοιε πρωτοβουλίε περί κράτου δικαίου που αναλαμβάνονται σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση όταν αυτέ συμφωνούν με, το πνεύμα και το γράμμα των συνθήκων. Και αναλαμβάνοντα υπόψη ότι σύμφωνα με τι αρχέ τη η Ευρωπαϊκή Ένωση εργάζεται με, τις με βάση τι αρμοδιότητε που τη χορηγούνται από τα κράτη-μέλη με βάση τις συνθήκες για την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων. Οποιαδήποτε αρμοδιότητα δεν χορηγείται στην Ένωση από τις συνθήκες παραμένει στο επίπεδο των κρατών μελών. Δυστυχώς αυτός ο συνδυασμός, ε, αυτός ο νέος μηχανισμός μάλλον που συνδυάζει τον προπολογισμό με ε, το δίκαιο δεν εγγυάται την νομική ασφάλεια των κρατών μελών. Η αιρεσιμότητα περί ε, των κονδυλίων που θα πανώνται θα πρέπει να βασίζεται σε συγκεκριμένους στόχους με και στα κατάλληλα κριτήρια. Δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει σε μη συγκεκριμένες απειλές ή φοβίες της αριστεράς όπως αυτές παρουσιάζονται εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο. Το προτινόμενο σχέδιο του κειμένου δεν πληρεί τα απαραίτητα κριτήρια, δίνει υπερβολικά ε, ε, μεγάλη λαβή δεν είναι πολιτικής φύσης και δεν είναι και ούτε και οικονομικής φύσης. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Και θα δώσω το λόγο στην κυρία Σίλβια Μόντι και τώρα. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το αντίθετο του κράτους δικαίου είναι η δικτατορία. Γι' αυτό και το κράτο δικαίου είναι μία από τι θεμελιώδει αξίε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Χρειαζόμαστε έναν μηχανισμό μέσω του οποίου να εγγυόμαστε ότι δεν δίνουμε χρήματα σε χώρε που δεν σέβονται το κράτο δικαίου. Αυτό είναι καθήκον μα απέναντι στου φορολογούμενου πολίτε. Εάν δεν υπάρχει πραγματικό ε, και ισχυρό νομικό ε, κράτος, κράτος δικαίου, δεν είμαστε βέβαιοι ότι θα τιμωρηθούν αδικήματα ή και εγκλήματα. Τώρα που υιοθετούμε το Ταμείο Ανάκαμψης, το Κονδύλι Ανάπαξης, ορισμένα χρήματα από αυτά θα πάνε σε χώρες όπου το κράτος δικαίου δεν ανθεί. Πρέπει να ζητήσουμε, απαιτήσουμε από τα κράτη που παίρνουν χρήματα να σέβονται τις αρχές του κράτους δικαίου. Αν η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν δεν επιμείνει στην αρχή του κράτους δικαίου, τότε δεν είμαστε πλέον η κοινότητα των αξιών που επιθυμούσαν οι ιδρυτικοί πατέρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Τώρα το λόγο θα πάρει ο κύριος Μάριο Φουρόρε. Grazie, Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η Ευρώπη πρέπει να επιμείνει στην εγγύηση του κράτους δικαίου μέσω βέβαιων και σταθερών κανόνων που δεν επιτρέπουν διακρίσεις ή διακριτική ευχέρεια. Δεν θέλουμε αυτά όλα να χρησιμοποιηθούν για πολιτικούς λόγους. Γι' αυτό καλώ το Συμβούλιο και την Κομισιόν να προβλέψει συγκεκριμένους κανόνες και ξεκάθαρους κανόνες για να οριστεί το κράτος δικαίου συγκεκριμένα, ξεκάθαρα και θα βασίζεται σε μετρήσιμου και παληθεύσιμους δείκτες. Προληπτική παρακολουθήση παρακολούθηση των προβλημάτων που βασίζεται σε αιτήσια ε, ανάλυση. Δεν θέλουμε να επιβληθούν επιπλέον ε, περιορισμοί που θα βασίζονται σε μακροαιρεσιμότητα, αλλά πρέπει να εγγυηθούμε τις αρχές της νομιμότητας και την εξαρτησία του δικαστικού σώματος. Και γι' αυτό θέλουμε να υπάρξει ένα κείμενο το οποίο θα είναι ένα αποτελεσματικό μέσο ώστε να εγγυηθούμε πως η Ευρώπη και οι πολίτες τους προστατεύονται. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Τώρα συνεχίζουμε στις ατομικές παρεμβάσεις των Ευρωβουλευτών. Ο Τόμας Τσεχόφσκι είναι ο επόμενος. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε που μου δίνετε το λόγο. Δεν θα καταχραστώ το ένα μου λεφτό για να επιτεθώ σε κάποιον είτε από τη δεξιά είτε από την αριστερά, γιατί δεν πρόκειται περί αυτού αγαπητοί συνάδελφοι εδώ. πάντα είμαστε κατά κάποιου, του Φιντές, ε, των Σελιστών, δεν ξέρω τι. Όχι, εδώ πέρα ε, πρόκειται για κάτι άλλο. Πρέπει να είμαστε ενωμένοι απέναντι σε μια αρχή. Σε κάθε χώρα, όποια χώρα κι αν είναι αυτή, δεν θα τους υποστηρίζουμε, όποιο κόμμα κι αν κυριαρχεί, αν δεν τηρούν κάποιες αρχές. Όταν μια χώρα πάβει να σέβεται τα οικουμενικά ανθρώπινα δικαιώματα δεν είναι δυνατόν να στηρίζεται από μας οικονομικά. Με ευρωπαϊκούς πόρους δηλαδή και κονδύλια. Εξού και μιλάμε για διαπραγματεύσεις. Να ενώσουμε τις δυνάμεις μας απέναντι στο Συμβούλιο, να καθίσουμε κάτω στο τραπέζι, να συζητήσουμε μαζί όποιος και αν έχει την εξουσία στη μία ή στην άλλη χώρα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Επόμενος ομιλητή είναι η κυρία Φεραίρα Μάρκε. Σα ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ήθελα να ξεκινήσω χαιρετίζοντα τον Υπουργό Ροτ. Ξέρω πω το θέμα αυτό του είναι ιδιαίτερα προσφυλέ και γι' αυτό και βασιζόμαστε ε, σε εσά για την περάσπιση του κράτου δικαίου. Οποιαδήποτε χώρα θέλει να είναι υποψήφια για να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να τηρεί τα κριτήρια τη Κοπεχάγη και άρα να σέβεται το κράτο δικαίου. Δεν μπορεί να εγκαταλείψει αυτό, ε, αυτά τα κριτήρια όταν γίνει κράτος μέλος πια. Ε, έτσι έχει σταθεί και δημιουργηθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να διευκρινίσουμε ότι η οικονομική συμβολή των ε, Ευρωπαίων πολιτών για την οικοδόμηση του ίδιου του ευρωπαϊκού οράματος ε, συμβάλλει στην οικοδόμηση αυτού του ίδιου. Γι' αυτό και έχουμε φτιάξει έναν ισχυρό μηχανισμό που επιτρέπει να ενεργήσει κανείς όταν υπάρχει παραβίαση του κράτους δικαίου που προστατεύει τους δικαιούχους και σέβεται τις αρχές και τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε θέματα προπολογισμού. Τέλος, πρέπει να προστατεύσουμε τη δημοκρατία και το κράτος του δικαίου και να εγγυήσουμε ότι τα χρήματα των Ευρωπαίων φορολογούμενων χρησιμοποιούνται σωστά υπέρ των ευρωπαϊκών αξιών. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Μάρκες τώρα. Η κυρία Τσε έχει το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ο νέο προπολογισμό αποτελεί μια εξαιρετική ευκαιρία για την Ευρωπαϊκή Ένωση να προχωρήσει. Να βάλουμε τα χρήματά μα εκεί που πραγματικά χρειάζονται, στι ευρωπαϊκέ αξίε. Αυτέ πρέπει να είναι στο κέντρο του προπολογισμού μα. Ο μηχανισμός μας για προϋποθέσεις είναι ο κατάλληλος τρόπος να διασφαλίσουμε ότι οι κυβερνήσεις οι οποίες παραβιάζουν το δίκαιο θα τιμωρούνται. Όχι όμως ο κόσμος. Οπότε υπάρχει το θέμα των ε, δημεύσεων, των ε, κατασχέσεων, αλλά χρειάζεται φυσικά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Όταν γίνονται τέτοιες δημεύσεις θα πρέπει τα χρήματα να πηγαίνουν αλλού. Και επιτρέψτε μου τώρα να αναφερθώ στις πολιτικές δυσκολίες που πολύ συχνά συζητάει το Συμβούλιο. Ακούμε ότι υπάρχει θέμα συμφερόντων στις χώρες μέλη. Βεβαίως υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων. Αλλά μιλάμε για επικεφαλής κατών και κυβερνήσεων. Ο κύριος Ορμπάν δεν είναι ολόκληρη Ουγγαρία, οπότε εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να ακούσω τι πιστεύει γι' αυτό το Συμβούλιο. Το Συμβούλιο πρέπει να εκπροσωπεί τον κόσμο, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις και γι' αυτό να προστατεύει τη χρηματοδότηση. Πώς να υποχρεώσουμε τις κυβερνήσεις που δεν τηρούν τους κανόνες, όπου υπάρχει διαφθορά, να σταματήσουν να το κάνουν. Νομίζω ότι η απάντηση είναι σαφής. Δεν πρέπει να το επιτρέπουμε αυτό. Ευχαριστούμε πολύ. Επόμενος μιλητής, ο κύριος Γιώχαν Κούς. Ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι. Πιστεύω ότι κανείς εδώ στην αίθουσα δεν αμφισβητεί το κράτος δικαίου. Το κράτο δικαίου λοιπόν είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να τηρηθεί. Αυτό που παρουσιάζεται όμως ως πρόβλημα είναι η σύνδεση του κράτου δικαίου με ένα μηχανισμό ο οποίο ε, ενδεχομένω δεν θα ισχύει επίση όρους για όλους. Αυτό θεωρώ ότι αποτελεί προβληματικό σημείο και αμφισβητεί και την αρχή της δημοκρατίας ή για παράδειγμα την αρχή της επικουρικότητας. Θα πρέπει να προσέξουμε στον αγώνα κατά ενός κακού και έχουμε εδώ την Όλαφ και την ΕΠΟ και άλλες αρχές, το ελεκτικό συνέδριο για παράδειγμα για το κακό αυτό, στον αγώνα αυτό να μην καταλήξουμε σε ένα Lex όρμπαν που θα δεσμεύσει όλους τους υπόλοιπους και τελικά δεν θα πετύχει και το στόχο που έχει δημιουργηθεί, για τον οποίο έχει δημιουργηθεί. Γι' αυτό λοιπόν ας προσέξουμε να μην ξεπεράσουμε το στόχο τον οποίο έχουμε θέσει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και τώρα το λόγο έχει η κυρία Ποντσάντη Ομπιόρ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Πρέπει να προστατεύεται ο ευρωπαϊκό προπολογισμό από παραβιάσει κράτου δικαίου. Αλλά το να είμαστε άδικοι ή να μεροληπτούμε σε βάρο κάποια χώρα, αυτό δεν είναι σωστό. Οι παραβιάσει στο κράτο δικαίου έχουν πολλέ διαστάσει. Αλλά πρέπει να υπάρχει ένα αντικειμενικό κριτήριο ελάχιστο που να αναγνωρίζουν όλοι. Και αυτό είναι το να υπάρχουν πολιτικοί κρατούμενοι. Αυτό είναι κάτι ασύμβατο με το κράτος δικαίου. Οπότε όταν υπάρχουν τέτοιες αυθαίρετες κρατήσεις όπως συμβαίνει με τους Καταλανούς ηγέτες που η Ισπανία ε, κρατά στις φυλακές, αυτό είναι παραβίαση του κράτους δικαίου. Οι Ισπανικές αρχές δεν έχουν υπακούσει. Η Ισπανία εξακολουθεί να παραβιάζει τις αρχές αυτές και να ε, μην ακούει τις μειονότητες εκεί. Παραβιάζεται και στη Δύση το κράτος δικαίου. Αν σας ενδιαφέρει το κράτος δικαίου και η δημοκρατία, στρέψτε το βλέμμα προς την Ισπανία παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Θα δώσω τώρα το λόγο στην κυρία Χολμάιερ. Ένα λεπτό παρακαλώ. Κυρία Πρόεδρε, αγαπητέ Επιτροπέ, αγαπητοί συνάδελφοι, αυτό που μου κάνει εντύπωση στην παρούσα φάση είναι ότι μιλάμε για μια χώρα που ο καθένα μιλάει για μια χώρα που τον προβληματίζει. Αυτό όμω θεωρώ ότι είναι αντιφατικό με την έννοια του κράτου δικαίου. Το κράτο δικαίου προϋποθέτει ενιαία πρότυπα και θα πρέπει λοιπόν αυτά τα πρότυπα να τηρούνται σε όλους χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη τη χώρα ή το κόμμα τότε θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για κυρώσει και για μέτρα δεν με νοιάζει ποιος είναι ο Μισκάτο, ο Όρμπαν, ο έχουμε κάποιες προβληματικές περιπτώσεις σε διάφορες πολιτικές οικογένειες και έχουμε προβλήματα σε ό,τι αφορά το κράτος δικαίου και αυτό θέλω να το πω ευθαρσό. Θα πρέπει να κάνουμε συστημικούς ελέγχους. Να ελέγχουμε συστηματικά λοιπόν κατά πόσο λειτουργούν οι μηχανισμοί κράτου δικαίου. Να ελέγχουμε συστηματικά, για παράδειγμα, πώς γίνονται οι δημόσιες ε, δημόσιοι διαγωνισμοί για προμήθειες, δημόσιες προμήθειες, πώς θα πάνονται τα δημόσια χρήματα. Θα πρέπει να υπάρχει και ένα έγκαιρο σύστημα πληροφόρηση για να έχει νόημα να μπορούμε να ελέγχουμε τι γίνεται ανά πάσα στιγμή, να μην χρειάζεται να περιμένουμε μήνες και μήνες. Θα ήθελα να μην κοιτάξουμε λοιπόν τι γίνεται από πλευρά πολιτικών οικογενειών, όχι να κοιτάξουμε μόνο πρότυπα και μέτρα. Τότε μόνο θα είμαστε αξιόπιστοι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα, αντιπρόεδρος Μπαρλή. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Το θέμα αυτό το σημαντικό για την προστασία των, του κράτους δικαίου με κυρώσεις. Γιατί είναι σημαντικό αυτό. Γιατί καταρχάς έχουμε δεσμευτεί ε, όλοι μας όσοι έχουμε μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε ό,τι αφορά την κοινότητα αυτή αξιών. Και κατά δεύτερον γιατί δεν είναι πλέον κάτι αυτονόητο. Δυστυχώ, όλο και πιο πολλοί παίρνουν ε, πόρους από την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά δεν ε, τηρούν τις υποχρεώσεις τους τρίτων γιατί χωρίς σεβασμό των αρχών αυτών δεν μπορεί να λειτουργήσει τίποτα. Ούτε η ενιαία αγορά, ούτε τα δικαστήρια και τίποτα άλλο. Κατά τέταρτον, γιατί όλοι οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν την, το δικαίωμα να μην καταλήγουν σε παράνομες δραστηριότητες στα χρήματα τους. Και κατά πέμπτον, γιατί δεν καταλαβαίνουν αυτές οι κυβερνήσεις άλλη γλώσσα πέρα από τη γλώσσα του χρήματος. Αγαπητό Συμβούλιο και αγαπητή Επιτροπή, έχετε στο πλευρό σας το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε ό,τι αφορά την προστασία των χρήματων αυτών και για ένα σύστημα παρακολουθήσει, Αλλά να είστε βέβαιοι ότι θα υπάρχει αντίσταση από πλευρά μας αν αποδυναμώσετε ε, και ουσιαστικά αχρηστεύσετε αυτόν τον μηχανισμό γιατί ένας μηχανισμός προστασίας είναι προς το συμφέρον όλων των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ την Αντιπρόεδρο Μπάρλεϊ. Κρίστοφ Χάνσεν. Ένα λεπτό από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, κύριε ε, Υπουργέ Ρότ, κύριε Ρέιντερ. Πριν από δύο χρόνια υποβλήθη αυτή η πρόταση και εδώ και ένα χρόνο και παραπένω είναι γνωστή η άποψη του Κοινοβουλίου. Φαίνεται όμως το Συμβούλιο κύματα τον ύπνο του δικαίου. Ποτέ δεν υπήρχαν τόσο πολλέ προβληματικέ εγκαταστάσει σε τόσο πολλά κράτη-μέλη και ποτέ δεν διακυβεύονταν τόσο πολλά χρήματα. Οι αυτοκράτε, ε, τα αυτοκρατικά αυτά καθεστώτα γεμίζουν ε, τι τσέπε του με τα χρήματα αυτά και καταπατούν τι βασικέ μα αξίε το κράτος δικαίου δεν είναι κάτι το οποίο θα διαπραγματευτούμε στα πλαίσια του ΔΠ Και υπολογίζω και περιμένω από τη Γερμανική Προεδρία να προστατεύσει τους πολίτες και τις επιχειρήσεις εκεί που τη χρειάζονται πιο πολύ, όχι εκεί που καταπατώνται τα δικαιώματα της πιο ξεδιάτροπα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και τώρα να δώσω το λόγο στην κυρία Βόλτερς για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η ευρωπαϊκή μας δημοκρατία ε, είναι ευαίσθητη. Έχουμε κάποιους ολιγάρχες εδώ στην Ευρώπη που ε, προσπαθούν να καταστρέψουν την Ευρώπη και αποδυναμώνουν και τα θεσμικά εκείνα όργανα στις χώρες τους που ουσιαστικά ε, ποπτεύουν την ανάθεση των ευρωπαϊκών πόρων. Ξέρουν φυσικά τα κόλπα και δεν είναι τυχαίο αυτό, γιατί οι ολιγάρχε και οι λαϊκιστές, δεν χρειάζονται να πω ονόματα, κάνουν ό,τι μπορούν για να φροντίσουν ότι οι Ευρωπαϊκέ αυτέ επιδοτήσει θα καταλήξουν στι τσέπε τη κλικά του και των συμμοριών του. Και λε και δεν τις βλέπει κανεί. Ο μηχανισμό λοιπόν κράτο δικαίου είναι πάρα πολύ σημαντική πρόταση για μένα. τέτοιο μηχανισμό. Θα μπορέσουμε να επιβάλλουμε κυρώσει αν υπάρχουν αμφιβολίες για τον εθνικό έλεγχο και καλό τα κράτη-μέλη να μιλήσουν ξεκάθαρα, να υποστηρίξουν αυτές τις προτάσεις, ό,τι και να γίνει την επόμενη εβδομάδα, να υποστηρίξουν την Ευρωπαϊκή Δημοκρατία και το κράτος δικαίου και να προασπιστούν και τους Ευρωπαίους φορολογούμενους που ποτέ δεν συμφώνησαν με όποια έκφανση της διαφθοράς. Ευχαριστούμε την κυρία Βόλτερς. Επόμενος μελτής. Ο κύριος Οτμαρκάρας. Κυρία Πρόεδρε, επειδή η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ακριβώς ε, κοινότητα αξιών, είναι ντροπή το γεγονός ότι ως τώρα τα κρατη δεν έχουν συμφωνήσει για ένα μηχανισμό επιβολής κυρώσεων. Μπορεί να μην το ήθελαν και τον μπλόκαραν οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς έχουμε απλές αξιώσεις και έχουν βαρεθεί πλέον με υποσχέσεις. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να είναι αποφασιστικά γιατί μόνο έτσι με αποφασιστικότητα θα μπορέσουν να ανακτήσουν την εμπιστοσύνη των πολιτών. Και το λέω από πλευρά μα ξεκάθαρα. Δεν μπορεί να χορηγούνται κονδύλια σε χώρες και σε άτομα που καταπατούν τις ευρωπαϊκές ε, αξίες. Ο μηχανισμός του κράτους δικαίου θα πρέπει να είναι τμήμα του Next Generation EU και του επόμενου πολιτικού δημοσιονομικού πλαισίου. Θα πρέπει να είναι τμήμα του συνολικού πακέτου γιατί η τήρηση του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων αποτελεί προτεραιότητα όχι μόνο για τη Γερμανική Προεδρία, όχι μόνο για την Αυστριακή κυβέρνηση, αλλά για όλους μας, για όλους μας, γιατί είναι η βάση της κοινότητάς μας. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κάρας. Τώρα θα δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία εκπροσωπείται από τον κύριο Ρέιντερς. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, ε, κυρίες και κύριοι Ευρωβουλευτές. Πρώτα απ' όλα σας ευχαριστώ πολύ για τη σημερινή συζήτηση. Πολύ χαίρομαι που ακούω ότι συμφωνούμε πλήρως για τη σημασία που έχει η προστασία του προπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ξέρετε ότι η δικιά σας στήριξη είναι βασική. Ο σεβασμός του κράτους δικαίου αποτελεί προϋπόθεση, βασική προϋπόθεση μάλιστα, προκειμένου να τηρείται η χρηστή διαχείριση των οικονομικών μας. Και οι αρχές είναι απλές, προκειμένου να ελέγξουμε τη χρήση των δημοσιονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των κονδυλίων μάλλον που δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, γι' αυτό χρειαζόμαστε σε κάθε χώρα μέλος συστήματα ε, καλά δικαιοσύνης, να υπάρχουν υπηρεσίες διερεύνησης και εισαγγελία και συνεργασία των ε, αρχών όταν πρόκειται για χρήση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Όταν ε, κάτι τέτοιο όμως τίθεται σε κίνδυνο εξαιτία αδυναμιών στο κράτος δικαίου, τότε η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορεί, βάσει του μηχανισμού μας, να σταματήσει την πρόσβαση σε ευρωπαϊκή χρηματοδότηση με αναλογικό τρόπο. Επιτρέψτε μου εδώ να τονίσω ότι ο προτινόμενος μηχανισμός διασφαλίζει τη δικαιοσύνη και την αντικειμενικότητα της διαδικασίας, διότι ακούει πρώτα ε, τις απόψεις του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους και μετά αποφασίζει για την αναλογικότητα των μέτρων που θα ληφθούν. Επιπλέον, τα μέτρα τα οποία θα εγκριθούν εξαρτώνται από ε, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο επίσης. Ο μηχανισμός αυτός πρέπει να είναι γρήγορος και αποτελεσματικός. Η ψηφοφορία στο Συμβούλιο πρέπει να γίνεται με την αντιστραμμένη δική πλειοψηφία, έτσι όπως προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κάτι το οποίο διασφαλίζει να εγκρίνονται τα προτινόμενα μέτρα γρήγορα. Αξιότιμοι Ευρωβουλευτέ, σήμερα δεν έχουμε τέτοιον μηχανισμό για να προστατεύουμε τον ευρωπαϊκό προπολογισμό από γενικευμένε αδυναμίε ω πρωτοκράτο δικαίου στι χώρε μέλη. Ο μηχανισμό αυτό λοιπόν θα βελτιώσει την προστασία του ευρωπαϊκού προπολογισμού και θα καλύψει αυτό το σημαντικό κενό και υπάρχει μεγάλη ανάγκη σήμερα δεδομένου ότι υπάρχει αυξανόμενη χρηματοδότηση και ευελιξία από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Ένωση όπω έχει προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια του COVID-19. Και αυτή την ευελιξία πρέπει να την προστατεύσουμε με κάθε τρόπο υπέρ των Ευρωπαίων πολιτών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν είναι αποφασισμένη να συνεισφέρει στην εξέβρεση συμβιβασμού και καλεί το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να καταλήξουν γρήγορα σε συμφωνία όσον αφορά αυτή τη σημαντική πρόταση, αλλά και για ένα νέο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Γιατί είναι προς το συμφέρον όλων μας να καταλήξουμε γρήγορα σε μια συμφωνία προκειμένου ο νέος πολιετής δημοσιονομικός προϋπολογισμός να μπορέσει να τεθεί σε ισχύ ήδη από την 1η Ιανουαρίου του 2021. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να έχει στη διάθεσή της τα μέσα που χρειάζεται για ανάκαμψη διαρκείας για να στηρίξει τις επιχειρήσεις, τις περιφέρειες που έχουν πληγεί περισσότερο από την κρίση. Επίσης, το οφείλουμε στις επόμενες γενιές το σχέδιο ανάκαμψη ε, που έχουμε, θα έχουμε στη διάθεσή μας πρέπει να βοηθήσει να έχουμε μια Ευρωπαϊκή Ένωση περισσότερο πράσινη, περισσότερο ψηφιακή, αλλά και με μεγαλύτερη αντοχή που να συνάδει με τις αξίες της. Η Επιτροπή θα κάνει ό,τι μπορεί ώστε γρήγορα να υπάρξει συμφωνία φιλόδοξη ανάμεσα στους συνομοθέτες. Το Συμβούλιο να ξέρετε, ρώτη ότι είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε τις συζητήσεις στον τριμερή διάλογο προκειμένου να προοδεύσουμε και να προστατεύσουμε τον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποστηρίζοντας πάντα τις αξίες μας. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε. Τώρα θα δώσω το λόγο στον Υπουργό, τον κύριο Ρότ. Α, ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ρέιντερ, κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι βουλευτές. Ε, φοβόμαστε... Ε... Δεν φοβόμαστε μάλλον τις ε, αντίθετε απόψει, ούτε εμεί ούτε εσεί, γιατί η Ευρώπη βασίστηκε σε τέτοιε αντιπαλότητε. Πριν από δεκαετίε, οι προπάτορε τη Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορούσαν να φανταστούν ότι θα βρισκόμαστε κάποια στιγμή σε μια κατάσταση όπου στα σοβαρά θα πρέπει να καθόμασταν να ελέγξουμε κατά πόσον τηρούνται σε ίδιο βαθμό οι αρχέ και διατάξει των κράτου δικαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό που είπε η εκπρόσωπο του Ρωμά, θα ήθελα να επαναλάβω, ότι το θέμα είναι να υπάρχει ίση ε, μεταχείριση ε, παντού, σε όλα τα κράτη-μέλη, παντού να ελέγχεται αυτό. Ο Ντανιλ είναι. άμα αμφισβητεί την δικαιοσύνη της Προέδρου, θα ήθελα να πω το εξή. Όχι μόνο αυτά που είπε χθε ε, η καγκελάριο, αλλά και το πρόγραμμα της Προεδρίας που περιλαμβάνει μια πρόταση, η οποία φαντάζομαι θα χαροποιήσει τον κύριο Φρόιντ. Υποστηρίζουμε την πρόταση Ευρωπαϊκή Επιτροπή για σύνδεση των ε, πόρων τη Ευρωπαϊκή Ένωση με την τήρηση του κρατών δικαίου στα κράτη-μέλη. Αυτό λοιπόν είναι το θέμα, αγαπητέ κυρίε και κύριοι. Και πολύ απλά δεν μα φτάνει, δεν μα αρκεί. Γι' αυτό λοιπόν να σα πω ότι δεν κοιμόμαστε καθόλου τον ύπνο του δικαίου. Είμαστε ξύπνοι και άγρυπνοι. Σας το λέω αυτό, αυτή είναι η πρόταση της Προεδρίας. Στο Συμβούλιο, σε κάθε σχεδόν συνεδρίαση θα θέτουμε το θέμα του κράτους δικαίου. Η προγραμματιζόμενη έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το θέμα του κράτους δικαίου θα τη χρησιμοποιήσουμε για μία αντικειμενική ανταλλαγή απόψεων που σίγουρα όμως θα έχει και διαφορετικές απόψεις. Σας ευχαριστώ λοιπόν αγαπητοί βουλευτές για την ενθάρρυνση που μας δίνατε γιατί βλέπω ότι υπάρχει σε μεγάλο βαθμό συμφωνία αλλά μιας και όλα αυτά είναι ενταγμένα στα πλαίσια των διαπραγματεύσεων για το πολιτές δημοσιονομικών πλαίσιο ξέρετε ότι όλα συσχετίζονται. Δεν μιλάμε για ένα και μόνο τομέα. Παρόλα αυτά, να υπολογίσετε ότι ο ρόλος της καγκελαρίου θα και ο λόγος της καγκελαρίου θα συνεχίσει να ακούγονται. Δεν είναι μόνο τα χρήματα που μας ενώνουν και γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να απαντήσω στον κύριο Σαβαμά και στον κύριο Κόρνερ για το κατά πόσον έχουμε επαρκή φιλοδοξία. Θα ήθελα να απαντήσω με ένα εχειρό ναι πολιτικές εκπτώσεις δεν κάνουμε σε κανέναν. Και γι' αυτό λοιπόν προσλέπω στις μελλοντικές ε, διαπραγματεύσεις μαζί σας. Ε, πολλά διακυβεύονται, αλλά και η ενότητα της ε, ευρωπαϊκής κοινότητας που βασίζεται σε κοινέ αξίες. Και εδώ συγκαταλέγεται το κράτος δικαίου. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, Υπουργέ Ρώτα. Σας εύχομαι κάθε επιτυχία στις διαπραγματεύσεις. Και εδώ ολοκληρώνεται η σημερινή μας συζήτηση και διακόπτεται η συνεδρίαση μέχρι τις 6 και 4.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 Αγαπητοί συνάδελφοι, επανάληψη των εργασιών της Συνόδου της Ολομέλειας. Θα ήθελα να σας ανακοινώσω τα αποτελέσματα της δεύτερης ψηφοφορίας. Πρωτοβουλία των Ευρωπαίων Πολιτών για τα προσωρινά μέτρα ε, σε ό,τι αφορά τι προθεσμίε των σταδίων συγκέντρωση, επαλήθευση και εξέταση λόγω τη ε, της νόσου COVID-19. 19 15 τροπολογία εγκρίνεται. Η πρώτη ανάγνωση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ολοκληρωθεί. Κατευθυντήριες γραμμές ε, για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών. Ε, ομαδών ε, οι τροπολογίες εγκρίνονται. Τρία ξεχωριστή τροπολογία εγκρίνεται. Πρώτο τμήμα. Δεύτερο τμήμα της τρία εγκρίνεται. Τέσσερα πρώτο τμήμα εγκρίνεται. Τέσσερα δεύτερο τμήμα εγκρίνεται. Πέντε πρώτο τμήμα εγκρίνεται. Πέντε δεύτερο τμήμα εγκρίνεται. 5 τρίτο τμήμα εγκρίνεται, 6 σε τρία τμήματα, πρώτο τμήμα εγκρίνεται, δεύτερο τμήμα εγκρίνεται και τρίτο τμήμα εγκρίνεται. Και τέταρτο το ίδιο. 11 τροπολογία. Πρώτο τμήμα εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα τη 11 εγκρίνεται. 15 πρώτο τμήμα εγκρίνεται. 15 δεύτερο τμήμα εγκρίνεται. 17 πρώτο τμήμα εγκρίνεται. 17 δεύτερο τμήμα εγκρίνεται. Τροπολογία 20 πρώτο τμήμα εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα εγκρίνεται. 20 τρίτο τμήμα εγκρίνεται. 33 πρώτο τμήμα εγκρίνεται. 33 δύο δεύτερο τμήμα εγκρίνεται. Τροπολογία 36 εγκρίνεται. Τροπολογία 38 εγκρίνεται. Τροπολογία 28 καταπίπτει. Τροπολογία 37 εγκρίνεται και τροπολογία 7 καταπίπτει. Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού υπαριθμών 5 του Γενικού Προϋπολογισμού για το 2020. Τροπολογία 1. Απορρίπτεται. στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, για την υγειονομική κρίση μετά το COVID-19. 11 απορρίπτεται. Παράγραφος 1 πρώτο τμήμα εγκρίνεται. Παράγραφος 1 δεύτερο τμήμα εγκρίνεται. Τροπολογία 1 απορρίπτεται. Παράγραφος 2 εγκρίνεται. Τροπολογία 2 απορρίπτεται. Τροπολογία 7 απορρίπτεται. Τροπολογία 12 απορρίπτεται. Τροπολογία 13 απορρίπτεται. Τροπολογία 14 απορρίπτεται. Τροπολογία 15 Απορρίπτεται επίσης. Παράγραφος 9. Πρώτο τμήμα. Εγκρίνεται. Παράγραφος 9. Δεύτερο τμήμα. Εγκρίνεται. Παράγραφος 10. Εγκρίνεται. Τροπολογία 3. Απορρίπτεται. Τροπολογία 16. Απορρίπτεται και αυτή. Παράγραφος 11. Εγκρίνεται. Τροπολογία 17. Απορρίπτεται. Παράγραφος 12. Εγκρίνεται. Παράγραφος 13. Εγκρίνεται. Παράγραφος 14. Εγκρίνεται. Τροπολογία 25. Εγκρίνεται. Τροπολογία 22. Εγκρίνεται. Παράγραφος 25 σε δύο τμήματα. Το πρώτο τμήμα εγκρίνεται και το δεύτερο τμήμα το ίδιο. Εγκρίνεται. Τροπολογία 18. Εγκρίνεται. Τροπολογία 20, ε, παράγραφος 28 εγκρίνεται. Τροπολογία 19 εγκρίνεται. Παράγραφος 31 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα εγκρίνεται, δεύτερο τμήμα εγκρίνεται και αυτό. Παράγραφος 32 εγκρίνεται. Τροπολογία 23. Εγκρίνεται. Παράγραφος 34. Σε δύο τμήματα. Το πρώτο εγκρίνεται και το δεύτερο επίση. εγκρίνεται. Τροπολογία 24. Εγκρίνεται. Τροπολογία 26. Εγκρίνεται. Τροπολογία 20. Απορρίπτεται δυστυχώς. Παράγραφος 40. Πρώτο τμήμα εγκρίνεται. Και το δεύτερο τμήμα τη 40 επίση εγκρίνεται. Παράγραφο 42. Εγκρίνεται. Το θεωρώντα 5. Εγκρίνεται. Τροπολογία 4 απορρίπτεται. Η αιτιολογική σκέψη Β εγκρίνεται, ενώ η τροπολογία 5 απορρίπτεται. Η τροπολογία 6 επίση απορρίπτεται. Η τροπολογία 21 εγκρίνεται. Τροπολογία 9 απορρίπτεται. Τροπολογία 10 απορρίπτεται και η τροπολογία 8 απορρίπτεται επίσης. Οι ομάδε Σοσιαλιστών και Δημοκρατών και Ρηνιού μου ανακοίνωσαν κάποιε αλλαγέ στα ονόματα αντιπροσωπιών και ε, επιτρόπων που θα συμπεριληφθούν στα, στα πρακτικά ε, τη σημερινή συνόδου και θα, περιληφθούν, θα τεθούν σε ισχύ από τη στιγμή της έγκρισής του. από σήμερα δηλαδή. Και περνάμε στον τρίτο γύρο ε, ψηφοφορίων και θα δώσω πρώτο το λόγο στον κύριο Ταρντίνο που ζήτησε το λόγο δυνάμει το 159 άρθρου παράγραφος 4 σε ό,τι αφορά ε, την Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, Νέας Ζηλανδίας και τα, την ανταλλαγή δεδομένων για τα σοβαρά εγκλήματα και την τρομοκρατία επί της ουσίας αρμόδιος ο κύριος η κυρία Ταρντίνο, συγγνώμη, στην οποία δίνει και το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καταρχάς ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους και όδης συζητητέ για το έργο τους. Ποιος είναι ο στόχος να καταλήξουμε σε συστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να ε, υπογραφεί η Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Νέας Ιλανδίας για ανταλλαγές ε, δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μεταξύ Ευρωπόλ και των αρμοδίων αρχών της Νέας Ζηλανδίας για την καταπολέμηση της εγκληματικότητας και της τρομοκρατίας. Ξέρουμε ότι η τρομοκρατία εξακολουθεί να είναι σοβαρή απειλή και απόλυτη προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για όλα τα κρατημέλη καταπολέμησή της. Είναι υπερβολικός αριθμός των θυμάτων που θρηνήσαμε τα τελευταία χρόνια. Οι Ευρωπαίοι πολίτες έπεσαν ε, θύματα αυτής της άνευ προηγουμένου βίας και μίσους. Θα πρέπει να τερματιστεί αυτό. Η Νέα Ζηλανδία είναι μία από τις χώρες με τις οποίες συνεργαζόμαστε μετά από ε, τις πρόσφατες τρομοκρατικές επιθέσεις. Έχουμε κοινή αντίληψη για τα διάφορα θέματα και καλή συνεργασία με τη Νέα Ζηλανδία. Αυτή τη στιγμή η Ευρωπόλ και οι αστυνομικές αρχές ε, της Νέας Ζηλανδίας έχουν ε, συνάψει μια συμφωνία διαρθρωτικής συνεργασίας τροποτινά, ένα μνημόνιο, αλλά δεν έχουν νομική βάση για να καταπολεμήσουμε την τρομοκρατία και να προλαμβάνουμε τις τρομοκρατικές επιθέσεις το κείμενό μου επιμένω σε κάποια στοιχεία που πρέπει οπωσδήποτε να αναφέρει η συμφωνία, όπως είναι η μεταφορά ε, προσωπικών δεδομένων για την καταπολέμηση τέτοιου είδους ε, πράξεων, θα πρέπει να προστατεύονται και τα δικαιώματα των προσώπων. Έτσι, ε, προς αυτή την κατεύθυνση εργάστηκα για να έχουμε μια καλή ισορροπία ανάμεσα στα δύο. Καταπολέμηση της διεθνούς τρομοκρατίας, αλλά και σεβασμό των ανθρωπίνων και προσωπικών δικαιωμάτων. Ελπίζω αύριο ε, να αναγνωρίσει η Ολομέλεια αυτές μου τις προσπάθειες. Ευχαριστώ. Από τις 6.30 μέχρι τις 19.45 θα διαρκέσει η ψηφοφορία με την ίδια μέθοδο και τον ίδιο τρόπο που ισχύει και για τον προηγούμενο γύρο ψηφοφορίας. Λοιπόν, αρχίζει τώρα ο τρίτος γύρος ψηφοφορίας και έχετε μέχρι τις 8 για να ψηφίσετε ώρα Βρυξελών τα αποτελέσματα θα σας ανακοινωθούν αύριο στις 9 το πρωί. Στις 8 παρατέταρτο, μετά το τέλος ε, της ψηφοφορίας θα λήξει η συνεδρίαση και θα επαναληφθεί ε, ε, στις 9 το πρωί. Έχει δημοσιευθεί η διάταξη και μπορείτε να τη βρείτε στην ιστοσελίδα του Κοινοβουλίου. Σας ευχαριστώ.